Αγαπητοί συνάδελφοι, πού τους είδα. Παρακαλώ, καθίστε για να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Καταρχήν, να συγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Δεν βλέπω αντιρρήσεις, άρα εγκρίνεται. Ανακοινώσεις του Πρόεδρου. Να σας πω ότι μεταδίδεται στο διαδίκτυο η συνεδρίαση αυτή και να σας πω επίσης για την αντιπροσωπεία στο Ντακάρ, της οποίας προέδρευσα εγώ. Στο σημείο 3 έχετε τα πρακτικά ήδη των συνεδριάσεων της 24ης και 25ης Ιανουαρίου, της 1ης Φεβρουαρίου και της 14ης Φεβρουαρίου. Δεν έχω ακούσει σχόλια για αυτά, συνεπώς θεωρούνται εγκεκριμένα. Και έτσι περνάμε στο σημείο 4. Προτείνω να έχουμε, όπως προβλέπετε, ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Κώσ Ρισελ, που είναι ο νέος Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης. Είναι δηλαδή κατά κάποιο τρόπο ο συνομιλητής μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλάβατε την 1η Ιανουαρίου του 2011. Μετά από χρόνια με τα οποία ασχοληθήκατε με την ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάτι το οποίο δίχως άλλο ε, σας έχει βοηθήσει να έχετε μεγάλη εμπειρία στο θέμα των μικροπιστώσεων, που είναι ένα θέμα που και εμάς μας απασχολεί πολύ, που είμαστε και Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων. Έρχεστε από την Ολλανδία. Εκεί αναλάβατε πολλές δραστηριότητες στην Ολλανδική Δίκηση και ως Γενικός Διευθυντής για τα θέματα απασχόλησης τώρα. Θα σας δώσω το λόγο, ξέρετε, πρώτα μια παρουσίαση από εσά και μετά ερωτήσεις. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι ένα από τα πράγματα που μας ενδιαφέρουν εμάς είναι να σας δοκιμάσουμε όχι, να το πω πιο σωστά, διορθώνει ο πρόεδρο, να γνωριστούμε πρώτα απ' όλα και να υποφεληθούμε από αυτή την ανταλλαγή απόψεων για να καταλάβουμε από εσά πώ αντιλαμβάνεστε εσεί την εργασία ε, στην γενική σας διεύθυνση, πώς θα δουλέψετε, πώς βλέπετε τα κείμενα τα οποία μας έρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξέρετε ότι και εμεί ορίζουμε εισηγητή για τα κείμενα τα οποία μα έρχονται από εσά. Για να μπορέσουμε πάντως να οργανωθούμε και εμείς καλύτερα, θέλουμε να ξέρουμε πώς εσείς προγραμματίζετε ε, συνομιλίες, συνεργασία και διαπραγματεύσεις μαζί μας κάθε φορά που έχετε έτοιμο ένα νέο κείμενο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια και σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε εδώ για να μπορέσουμε να μιλήσουμε μαζί. Όντως, θέλω να ξεκινήσω ε, ξέρετε, λέμε ότι ξεκινάει κανείς μερικές φορές πέφτει στα βαθιά. Ε, λοιπόν, αυτό βλέπω και εγώ μπαίνοντα εδώ σήμερα στην Επιτροπή σας. Έχουμε τις τακτικές μας δραστηριότητες, αλλά από την άλλη μεριά έχουμε να ασχοληθούμε και με πολύ ιδιαίτερα θέματα, που είναι η συμμετοχή του πρώτου ποτέ εξαμήνου του ευρώ και επίσης να ετοιμάσουμε το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο. Όσον αφορά το ευρωπαϊκό εξάμεινο, χαιρόμαστε πολύ που συμμετέχουμε στην ομάδα των τριών που διαπραγματεύεται και συζητά με όλα τα κράτη-μέλη. Υπάρχει μια τρόικα όπου συμμετέχει η Γενική Γραμματεία για τον Συντονισμό, η Γενική Διεύθυνση για τα Μακροοικονομικά και η Γενική Διεύθυνση για την Απασχόληση. Ακριβώς για να μην μείνει απ' έξω ο κοινωνικός τομέας. Γιατί δεν θέλουμε να συζητάμε μόνο για φορολογικά μέτρα και για λιτότητα και για μακροοικονομικά ζητήματα, αλλά να υπάρχει και η κοινωνική διάσταση που να λαμβάνεται και αυτή υπόψη. Ξέρετε ότι στη στρατηγική Ευρώπη για το 2020 θέτουμε στόχους. Και το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι αν σήμερα δείτε τι αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη στα προκαταρτικά τους προγράμματα, γιατί είναι προσωρινά, θα διαπιστώσετε ότι στο κοινωνικό τομέα δεν καλύπτονται οι στόχοι. Η συμμετοχή 5% στην αγορά εργασία με 20 εκατομμύρια εκτός ένδυα μέχρι το 2020. Αυτή λοιπόν είναι και η κύρια ανησυχία μας κάθε φορά που συζητάμε με τα κράτη-μέλη. Είχαμε συζήτηση σαν πρώτο γύρο. Τώρα γυρίσαν όλοι πίσω. Τον Απρίλιο θα έρθουν με τα εθνικά προγράμματα. Και εμείς θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες συστάσεις τότε. Σε ολόκληρο λοιπόν αυτόν τον τομέα, η ΕΠΣΚΟ θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο και στις συνεδριάσεις που θα έχουμε τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου, που θα προετοιμαστεί από τα κράτη-μέλη στην Επιτροπή ΕΜΚΟ με την Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας. Συμφώνησαν μεταξύ τους να συνεργαστούν στενά Επίσημα μόνο η ΕΜΚΟ παίζει ρόλο, αλλά υπάρχει συντονισμός και με την Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας. Όσον αφορά τις ατομικές συστάσεις προς τα κράτη-μέλη, θα δούμε πόσο μακριά θα μπορέσουμε να πάμε. Είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε αυτό. Πρέπει να είμαστε σαφείς και πρέπει στα πλαίσια της στρατηγικής 2020 να βάλουμε τις συστάσεις μας. Συγχρόνως όμως πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές. Να ξέρουμε τι μπορούν να κάνουν τα κράτη-μέλη και να τα ενθαρρύνουμε όσο γίνεται περισσότερο, ώστε να θέσουν σε εφαρμογή τις δράσεις που έχουν αποφασίσει. Για το πολιετές τώρα δημοσιονομικό πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούνιο θα κοινοποιήσει την ε, θέση της. Θα είναι βέβαια ένα σημαντικό γεγονός και ενδιαφέρον και ελπίζουμε ότι και η δικιά σας Επιτροπή θα δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το αποτέλεσμα προετοιμάζουμε το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και θέτουμε στους αυτούς μας ε, στοιχειώδη και σημαντικά ερωτήματα. Για παράδειγμα, πρέπει να μπουν στόχοι για το πού θα πάνε τα κονδύλια του κοινωνικού ταμείου εξάντε ή πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι προγράμματα θα μας φέρουν οι περιφέρειες και οι χώρες της Ευρώπης. Ακόμα δεν έχουμε αποφανθεί για την πολιτική μας ε, προτίμηση. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να έχουμε κάποια ιδέα γιατί με τα χρόνια έχουμε διαπιστώσει ποιο είναι το ποσοστό του κοινωνικού ταμείου σε σχέση με το σύνολο των ε, ταμείων συνοχής που από το 40 πήγε στο 20%. Κάποιες ορισμένες περιοχές, ε, περιφέρειες τα καταφέρουν καλύτερα από άλλες. Πάντως αυτό είναι το αποτέλεσμα. Οπότε το ερώτημα είναι θα καθίσουμε σταυρωμένα τα χέρια να δούμε απλώς πώς προχωράνε τα πράγματα ή θα εκφράσουμε κάποια προτίμηση. Ορισμένοι θέλουν εξάντε στόχους. Έπειτα, δεν είναι απλώς υπόθεση δίνουμε χρήματα στον κοινωνικό ταμείο, αλλά κάνουμε και τη σύνδεση με τους στόχους της στρατηγικής 2020. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει αυτή η σύνδεση. Είναι βέβαια πολιτική συζήτηση και ορισμένες χώρες τη στάζουν. Πάντως το αποτέλεσμα θα είναι αποφασιστική σημασία και για το μέγεθος ε, του κοινωνικού ταμείου. Πέντε χώρες θέλουν περιορισμό των κονδυλίων σε κοινοτικό επίπεδο. Πρέπει να δούμε κατά πόσο θα περιοριστεί το επίπεδο κονδυλίων για τα κοινωνικά θέματα ή όχι. Και για την κοινωτική διάσταση. Το βέβαιο είναι ότι θέλουμε να διοθετήσουμε αυτό που κάνουμε. Όχι μόνο θεματικά, ανατομέα, αλλά και αναπεριφέρεια. Θέλουμε να εντοπίσουμε συγκεκριμένους στόχους. Άρα πρέπει να δούμε την περιφέρεια συνολικά, με όλα τα ταμεία ένα συμβόλαιο με κάθε περιφέρεια και εκεί μέσα να είναι όλα όσα πρόκειται να γίνουν. Αυτά λοιπόν θα συζητάμε το πρώτο εξάμεινο, προκειμένου να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα τον Ιούνιο. Επιπλέον, υπάρχει και το ε, νομοθετικό πρόγραμμα. Δύο από τα ζητήματα τα οποία πετούν μεγάλη πολιτική προσοχή είναι οι ώρες εργασίας, η οδηγία αυτή, και η οδηγία για τους αποσπασμένους εργαζόμενους. Ζητήσαμε από τους κοινωνικούς εταίρους να εκφράσουν την άποψή τους, κατά πόσο θέλουν, είναι έτοιμοι ή όχι μεταξύ τους να συζητήσουν για την οδηγία για το χρόνο εργασίας. Πρόσφατα ακούμε, δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα γραπτά, ακούμε ότι οι κοινωνικοί εταίροι πράγματι θέλουν να αναλάβουν την πρόκληση αυτή και να συμμετάσχουν στην διαπραγμάτευση για την οδηγία για το χρόνο εργασία. Υπάρχει βέβαια μια προθεσμία για την απάντησή τους. Αρχέ Απριλίου πρέπει να έχουν θέση. Πιστεύουμε πάντως ότι είναι έτοιμοι να έρθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Δεν θα πάνε γρήγορα τα πράγματα γιατί πρέπει να γεφυρωθούν διαφορετικές και αποκλίνουσες απόψεις. Φαίνεται όμω ότι αναλαμβάνουν και εκείνοι τι ευθύνε του. Για την απόσπαση εργαζόμενων τώρα. Α, και συγγνώμη να συμπληρώσω, λέει ο μιλητή, ότι η Επιτροπή πρέπει να περιμένει του κοινωνικού εταίρου, οι οποίοι έχουν στη διάθεσή του 9 μήνε. Από την έναρξη των διαπραγματεύσεων έχουν εννέα μήνε. Και αν τελικά δεν καταλήξουν σε αποτέλεσμα, τότε το μπαλάκι είναι στο γήπεδο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κληθεί να παρουσιάσει πρωτοβουλία. Έρχομαι τώρα στην άλλη οδηγία ε, για, την απόσπαση εργαζομένων, που είναι και αυτή ιδιαίτερα πολιτικού χαρακτήρα. Προ το παρόν θέλουμε το θέμα αυτό να το έχουμε με ένα κείμενο στο δεύτερο εξάμεινο της χρονιάς αυτής. Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορεί να είναι, δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα, σε δύο τμήματα. Το ένα να αναφέρεται για την εφαρμογή της οδηγίας, δηλαδή να διευκρινίζει ποιες είναι οι έννοιες και πώς πρέπει να λειτουργήσει η οδηγία και το δεύτερο τμήμα να είναι ε, δράση στα πλαίσια της νέας πράξης, που εξηγεί τη σχέση ανάμεσα στις οικονομικές ελευθερίες και τα θεμελιώδη και κοινωνικά δικαιώματα. Είναι υποσυζήτηση πάντως το θέμα και δεν θα έχουμε τίποτα έτοιμο πριν από το δεύτερο εξάμεινο της χρονιάς. Στα τέλη πάντως αυτού του εξαμήνου Μπορούμε να περιμένουμε την οδηγία για την ηλεκτρομαγνητική εκτινοβολία. Δουλεύουμε πάνω σε μία οδηγία επίσης ε, για ε, διαταρχές του ημασκελετικού συστήματος. Και αυτό για το δεύτερο εξάμεινο της χρονιάς. Δουλεύουμε επίσης και όσον αφορά το κάπνισμα. Με οδηγία που θα έρθει. Δεν ξέρουμε όμως αν θα προλάβουμε μέσα στο 2011 να έχουμε έτοιμη μια τέτοια οδηγία. Αυτό που είναι βέβαια σημαντικό είναι ότι θα έχουμε και για τις συντάξεις μια λευκή βίβλο. Έχουμε 1.700 αντιδράσεις και δουλεύουμε πάνω σε αυτές, τις εξετάζουμε. Θα έχουμε κάτι έτοιμο στις αρχές του δεύτερου εξαμήνου της χρονιάς αυτής. Θα υπάρχει κείμενο επίσης για τις δημογραφικές εξελίξεις. Για τους Ρώμα επίσης, μια ανακοίνωση. Σημαντικά θέματα πολιτικής που συζητιώνται και θα συζητιώνται ακόμα. Λίγο πολύ αυτή είναι η μερίσια διάταξη για τη φετινή χρονιά. Για τα δύο μεγάλα πολιτικά θέματα, το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο δηλαδή, και για το ευρωπαϊκό εξάμεινο υπάρχουν ήδη ημερομηνίε. Για τα άλλα προχωράμε σιγά σιγά. Προς το παρόν αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την παρουσίαση. Muchas gracias, señora presidenta. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ρισελ ίσως ε, και άλλοι σοσιαλιστές συνάδελφοι να σας ε, εκφέρουν την άποψή τους. Εγώ θα αρκεστώ ως συντονιστής ομάδας να σας ε, καλωσορίσω και να σας πω ότι από τη δική μας πλευρά θα έχετε όλη την δυνατή βοήθεια για την ανάπτυξη αυτής της Γενικής Διεύθυνσης που είναι σημαντική για εκατομμύρια Ευρωπαίους που με μεγάλη δυσκολία βλέπουν να περιπλέκονται οι εργασιακές σχέσεις και με μεγάλη απογοήτευση δεν βρίσκουν εργασία παρά το γεγονός ότι έχουν σπουδάσει και θα μπορούσαν. Αυτό το βλέπουν άντρες και γυναίκες και κυρίως νέοι. Αυτό που μας ενδιαφέρει λοιπόν είναι να βελτιώσουμε τον ορίζοντά μας και την διαθεσμική συνεργασία. Γι' αυτό με μεγάλη ικανοποίηση δέχομαι την εισήγησή σας γιατί μας είπατε ότι η Γενική Διεύθυνση της Απασχόλησης θα συνεργαστεί με την ε, Τρόικα που προετοιμάζει το Ευρωπαϊκό εξάμεινο και μέσα στα πλαίσια της ΕΠΣΚΟ θα λάβουμε υπόψη την κοινωνική διάσταση της ε, κρίσης και με τις άλλες διαστάσεις που είναι πολύ σημαντικές και όχι όμως οι μόνες. Επίσης, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο με βάση πραγματιστικά στοιχεία και με αντιμετώπιση της πραγματικότητας. Επίσης, θα ήθελα να ασχοληθούμε με αυτή την ε, εξισορρόπηση που αφορά την γενική σας διάθεση. Υπάρχει ένα ειδικό κεφάλαιο. Το θέμα της μετανάστευσης στην Ευρώπη έχει ε, δραματικές συνέπειες στην αγορά εργασίας. Γι' αυτό θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να μην ανακύψει ρατσισμός και ξενοφοβία. Δυστυχώς όμως η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης πόρο απέχει από το να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Νομίζω ότι ε, ασχολούνται άλλοι επίτροποι και άλλες γενικές διευθύνσεις, αλλά δεν αφορά τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, δεν εντάσσεται στα καθήκοντά της. Ε, νομίζω ότι θα ανακύψουν και άλλες οδηγίες, όπως αυτή που αφορά τις εταιρικές σχέσεις, το εταιρικό δίκαιο και άλλες οδηγίες. Νομίζω ότι θα πρέπει να ενταχθεί στις ε, δικές σας αρμοδιότητες για να μην ξεχάσουμε τα εκατομμύρια εργαζόμενα στους μετανάστευς που θέλουν να ενταχθούν ε, ε, συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη μια σωστή ενσωμάτωσή τους στην, ε, στις δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυρία Φιγκέιρετ και ο κύριος Κρίστινσεν Στη συνέχεια, η κυρία Φιγκέιρετ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δύο σύντομες παρατηρήσεις. Η πρώτη για τα θέματα της κοινωνικής διάστασης της κρίσης ή της κοινωνικής κρίσης ε, θα ήθελα να πω που ζούμε στις μέρες μας και που σε κάποιες χώρες είναι πολύ σοβαρή όπως στην περίπτωση τη δική μου της Πορτογαλίας αλλά μην ξεχνάμε και την Ελλάδα, την Ιρλανδία και άλλες χώρες όπου επίσης παρόμοιες περικοπές μισθών έχουμε και κοινωνικών ε, επιδομάτων και αύξηση ανεργίας και τώρα ακόμα και προαναγγελίες ε, περικοπών συντάξεων που δίνουν που είναι ήδη χαμηλές όπως είναι και στη χώρα μου εξάλλου. Όλα αυτά εξ ονόματος της αηφορίας λέει των δημοσιονομικών. Εξ ονόματος της δημοσιονομικής αηφορίας. Αυξάνεται η φτώχεια σε ασύλληπτα επίπεδα πλέον αδιανόητη υπόθεση αυτή και οι ανισότητες σε πραγματικά αδιανόητα επίπεδα. Ερωτώ και διαρωτώ με πού βρίσκεται η κοινωνική διάσταση στην κρίση, σε αυτή τη διαδικασία. Πού είναι η αρχή της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικής συνοχής. Πού βρίσκονται όλα αυτά που έχουν χαθεί. Και επίσης εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε κάποιες εκθέσεις όπως μία για ελάχιστους μισθούς ε, όσον αφορά το ευρωπαϊκό επίπεδο. Ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει κάποια πρόταση σε αυτό το επίπεδο. Επίσης υπενθυμίζω μια γραπτή δήλωση, μια διακήρυξη γραπτή για το πρόβλημα των αστέγων και που έχει προσυπογράψει η πλειοψηφία των Ευρωβουλευτών σε αυτή την Ευρωβουλή και επίσης εμένω και επιμένω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει μια πρωτοβουλία από πλευρά της. Κάτι πρέπει να κάνει. Και είναι ολόκληρη τομή, ολόκληρα πεδία αυτά που είναι πάρα πολύ ευαίσθητα για αυτά τα θέματα. Και ρωτώ, τι γίνεται, τι προετοιμάζεται σε αυτά τα επίπεδα. Ευχαριστώ. Ε, Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που θα ήθελαν το λόγο, κυρία Γιάκον Σάρη. Μάνα Μαρκίν. Μάρκιν. Ντελή. Υπάρχουν και άνδρες σε αυτή την επιτροπή. Κλείνει ο κατάλογος των ομιλήτων με αυτούς που σας προανέφερα ο κύριος Κρίστιανσεν. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ επίσης τον Γενικό Διευθυντή για τις πληροφορίες. Είναι πολύ ενδιαφέροντα θέματα αυτά που έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη και για το μέλλον πολύ ενδιαφέροντα. Ένα πεδίο θέλω να αναφέρω που δεν αναφέρατε, το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Το Ταμείο Αντιμετώπισης των Επιπτώσεων της Παγκοσμιοποίησης είναι ένα από τα πιο σημαντικά μέσα στήριξης που έχουμε στη διάθεσή μας, ώστε να μπορέσουμε τους απολυμμένους, ε, όσους έχουν χάσει θέσεις εργασίας, να τους επανεντάξουμε στην απασχόληση. Δυστυχώς επανειλημμένα καταδείχθηκε ότι, πώς να το πω, όλα αυτά είχαν ικτρό τέλος είχαν αρνητική έκβαση διότι η διοικητική περίοδος διαχείρισης μεταξύ του αιτήματο και της διάθεσης των κονδυλίων μπορεί να είναι ένα ολόκληρο έτος. Και σε κάποια κράτη-μέλη τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει δυστυχώς ότι περίπου ένα χρόνο θα έχει κανείς στη διάθεσή του για ένα τέτοιο πρόγραμμα όλο και όλο. Διότι υπάρχει εδώ ένα εδάφιο που λέει ότι τρεις μήνες λέει, μετά την υποβολή αιτήσεων ε, ξεκινά το διετές, η διετής περίοδος που υπολογίζεται. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν τον Γενικό Διευθυντή, δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή η περίοδος να ξεκινήσει αμέσως με την χρονική εκείνη στιγμή που θα γνωρίζει ότι τα κονδύλια θα είναι διαθέσιμα. Υπάρχουν καν τέτοιες δυνατότητες ή όχι. Με άλλα λόγια θα πρέπει αυτό το ταμείο να το αναθεωρήσουμε κάπως, να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Θα ήταν δυνατόν να συντμηθεί η διοικητική περίοδος, όλη αυτή η διοικητική αναμονή θα έλεγα σε αυτήν την περίοδο για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Θα μπορούσε να υπάρξει μια δυνατότητα παράδειγμα αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωκοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη συνερχόντουσαν και αξιολογούσαν όλα αυτά τα προγράμματα, τα σχέδια αυτά. Τα κράτη-μέλη τι θα έκαναν, θα είχαν εχέγγυα θα έλεγαν αν ακολουθηθεί αυτή η γραμμή τότε αυτό το πρόγραμμα θα μπορέσει να εγκριθεί και θα λειτουργήσει. Μπορείτε λοιπόν να ξεκινήσετε με όλες αυτές τις δραστηριότητες για την κατάρτιση και εκπαίδευση που είναι πολύ σημαντικές και αυτό θα ήταν μια δυνατότητα επιτάχυνσης. Αν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα θα υπάρχει ο κίνδυνος κάποιοι από τους ανέργους αυτούς να μην έχουν αρκετό χρόνο στη διάθεσή τους για να μπορέσουν να καταρτιστούν ή δεν θα υπάρχουν τα κονδύλια έγκαιρα διαθέσιμα για να γίνει αυτό. Ευχαριστώ. Thank you very Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις αυτές. Ως προς θέμα των μεταναστών, Πρόκειται για ένα θέμα που απασχολεί διάφορα τμήματα της ε, Εκτελεστικής Επιτροπής και προσδίδουμε σημασία μέσα στα πλαίσια του Κοινωνικού Ταμείου στο θέμα της ενσωμάτωσης των ε, μεταναστών που έχουν άδεια παραμονής στις ε, χώρες μας. Τότε ανήκουν στην στοχοθέτηση του Ταμείου κοινωνικού ταμείου και μπορούν να ενσωματωθούν κατά διάφορους τρόπους, λαμβάνουμε υπόψη τις δεξιότητές τους. Μιλάμε για ΜΜΕ, για μικροπιστώσεις, μπορούν να τύχουν υποστήριξης. Πρέπει όμως να κατέχουν αυτό τον τίτλο. Διαφορετικά εμπίπτουν στην αρμοδιότητα άλλων γενικών διευθύνσεων μέσα στους πόρους άλλων γενικών διευθύνσεων. Το ΕΚΤ όμως ε, τους περιλαμβάνει τη στιγμή που έχουν άδεια παραμονής, που κατέχουν άδεια παραμονής. Ως προς το κοινωνικό στοιχείο της κρίσης και το γεγονός ότι πολλά αλλάζουν, κυρία Φιγκεϊρέδο, νομίζω ότι μετά την κρίση δεν θα βρεθούμε στο σημείο εκκίνησης πριν από την κρίση, δηλαδή τα πράγματα έχουν αλλάξει έχουν αλλάξει άρδιν ως προς τη διάρθρωσή τους. Υπάρχουν αναδυόμενες οικονομίες στην Ασία και άλλες εξελίξεις όπως τον αραβικό κόσμο. Δεν μπορούμε να αποτιμήσουμε τις συνέπειες αυτής της αναπτυξιακής πορείας ακόμα. Γι' αυτό είμαστε και ευέλικτοι απέναντι σε όλα αυτά τα θέματα, διότι γνωρίζουμε ότι θέματα ως προς το συνταξιοδοτικό θα πρέπει να μας απασχολήσουν, όπως και η ηλικία συνταξιοδότησης. Είναι κάτι που προέρχεται και από τα συνδικάτα. Δεν είναι μία απόλυτη άρνηση, απλώς ζητούν τη συμμετοχή τους σε αυτή τη διαδικασία διαβουλεύσεων. από πλευράς ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, ο οποίος είναι πολύ περιορισμένος, δεν είναι δυνατόν να αντικαταστήσουμε τα κοινωνικά ευεργετήματα, τα επιδόματα δηλαδή, σε εθνικό επίπεδο. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αποφασιστεί σε εθνικό επίπεδο. Εκεί θα αποφασίσει κανείς για τα κοινωνικά επιδόματα και βεβαίως τα κράτη-μέλη διαφέρουν κατά πολύ ως προς τους διαθέσιμους πόρους, τους όρους και τη διάρκεια χορήγησης αυτών των επιδομάτων. Ξέρετε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν θέλουμε να εναρμονίσουμε αλλά να συντονίσουμε. Προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό με ανάλυση στοιχεία έτσι ώστε να βλέπει το κάθε κράτος μέλος τι κάνει ένα άλλο, τα άλλα δηλαδή τι κάνουν τι γίνεται δηλαδή σε κάθε κράτος μέλος έτσι ώστε ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του και έτσι προσπαθούμε να προωθήσουμε τη συζήτηση και σε θέματα όπως αυτό της ευελιξασφάλειας. Είναι μια λέξη του σειρμού. Θα πρέπει όμως να μας απασχολήσει, να μην είναι μια λέξη κενή περιεχομένου και όχι μόνο ε, εγγράφος αλλά και έμπρακτα σε εθνικό επίπεδο. Θέλουμε λοιπόν να ασχοληθούμε με μερικές πτυχές του θέματος κρίσης. Γι' αυτό υπάρχει και το Ταμείο Αντιμετώπισης του Φαινομένου της Παγκοσμιοποίησης, το οποίο ασχολήθηκε με τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης αρχικά και μετά διευρύνθηκε για να ασχοληθεί και με θέματα κρίσης και εκτός προϋπολογισμού και τα δύο σκέλη των αποφάσεων νομοθετικού περιεχομένου θα πρέπει να εμπλακούν για την επιβολή μιας απόφασης. Αυτό είναι ένα από τα στοιχεία της ε, μακροχρόνιας διαδικασίας για τη λήψη απόφασης. Πρόκειται για ε, μία ε, ειδικά, μία πολύ φορτωμένη διαδικασία και τη στιγμή που, μας, ε, θα μας απασχολήσει το θέμα μέσα στα πλαίσια των πολιετών δημοσιονομικών προοπτικών, θα πρέπει να βρούμε ένα modus operandi το οποίο να μην είναι ε, τόσο βαρύ ως προς τη χρήση και ανέλικτο ως προς τη χρήση του Ταμείου Αντιμετώπισης της Παγκοσμιοποίησης. Έγινε λόγος για 500 εκατομμύρια ετησίως, αλλά αν ασχοληθούμε με την περίοδο εφαρμογής, και αφού διευρύναμε το πλαίσιο, μιλάμε για 220-250 εκατομμύρια ετησίως. Και αυτό δεν αφορά την μακροσκελή διαδικασία, διότι όταν έχουμε ένα αίτημα, τότε ασχολούμαστε άμεσα με αυτό. Ερχόμαστε σε επαφή με εκείνους που το προτείνουν για να δούμε κατά πόσο έχει νόημα η πρόταση και κατά πόσο εντάσσεται στα πλαίσια του κανονισμού αυτού. Εάν κάτι τέτοιο ισχύει, τότε θα πρέπει να επιτελεστεί λεπτομεριακή εργασία. Άρα, εξ αρχής πρόκειται για ε, μία διαδικασία η οποία μας επιβαρύνει ιδιαίτερα και μέσα σε αυτά τα πλαίσια προσπαθούμε να βελτιώσουμε το πλαίσιο λειτουργίας. Ας δούμε πώς θα μας απασχολήσει και στο μέλλον, διότι στα πλαίσια των πολιετών δημοσιονομικών προοπτικών θα πρέπει να συζητηθεί το κατά πόσο το Ταμείο ε, Παγκοσμιοποίησης ή το Ταμείο Αντιμετώπισης Κρίσης θα πρέπει να τύχει προσαρμογό. Η κυρία Γιακονσάρη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Μετά την κρίση ε, σκέφτονται πολύ για το τι συνέβη, τι πήγε στραβά και τι, μπορούσε να, τι μπορεί να γίνει καλύτερα στο μέλλον. Και ένα θέμα υποσυζήτηση σε όλα τα κράτη-μέλη είναι η παραοικονομία νομίζω σε όλα τα κράτη-μέλη το συζητούν αυτό. Θα θέλω να σας ρωτήσω πόσο ψηλά ως προτεραιότητα βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη η παραοικονομία και τα συναφή και ένα άλλο ερώτημα που συνδέεται με αυτό. Πιστεύετε εσείς ότι θα έπρεπε να είχαμε κάτι σαν μια, ας το πω έτσι, ευθύνη σε σχέση με το πανευρωπαϊκό επίπεδο για να αντιμετωπιστεί αυτή η πτυχή της παραοικονομίας. Ευχαριστώ. Thank ευχαριστώ και ευχαριστώ για την παρουσίασή σας αυτό το απόγευμα. Τα σχόλιά μου ουσιαστικά ήδη ακούστηκαν, προακούστηκαν και από κάποια μέλη σε σχέση με την οικονομική κρίση. Νομίζω η δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή και η Γενική Διεύθυνση της ε, Εκτελεστικής Επιτροπής έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν για αυτή την κρίση. Εσείς κάνατε λόγο για τα ε, κοινωνικά θέματα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να μπορέσουμε να δώσουμε μια όθηση και να ε, πετύχουμε κάποια πράγματα. Οι πολίτες μας στρέφονται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση βλέποντας το τι ε, γίνεται και η μόνη δυνατότητα που βλέπουν είναι ότι μόνο οικονομικά μέτρα λαμβάνονται και τίποτα δεν γίνεται για τα κοινωνικά θέματα. Υπάρχει το ενδιαφέρον για τα δημοσιονομικά και τα οικονομικά, αλλά δεν κάνουμε πολλά πράγματα για τα κοινωνικά και πρέπει για τις μικρές, ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις να δούμε τον ρόλο που πρέπει να διαδραματίζουν και τι μπορούν να κάνουν για τα κοινωνικά θέματα και την οικονομία. Σίγουρα χρειαζόμαστε πολύ μεγαλύτερη υποστήριξη για αυτά τα θέματα. Αναφέρατε τις συντάξεις για παράδειγμα. Είχαμε το πράσινο βιβλίο, αναμένουμε τώρα το λευκό βιβλίο για την αηφορία όσον αφορά την επάρκεια των συντάξεων. Εγώ προέρχομαι από την Ιρλανδία ως Ευρωβουλευτής και γνωρίζω πολύ καλά το μνημόνιο συνεννόησης που είχε συμφωνηθεί μεταξύ του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ιρλανδίας. Σε σχέση με το 17 δίσα για το Ταμείο Συντάξεων θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τώρα γι' αυτό. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει, λέει το ένα και δεν ε, σκέφτεται το άλλο, δεν κάνει κάτι για το άλλο. Δεν ελαχιστοποιώ τα όσα έχουν γίνει. Απλά λέω ότι το μήνυμα φαίνεται να είναι ότι καλύπτουμε και αντιμετωπίζουμε τα οικονομικά θέματα σε σχέση για παράδειγμα με τις, ε, τα θέματα των μισθών, ε, την επάρκεια. Γνωρίζω ότι δεν είναι δική σας αυτή η ευθύνη αλλά γνωρίζω ότι οι πολίτες το ζητούν αυτό, να αναλυφθεί δράση από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτά τα πεδία. Και αυτά τα οποία η δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή βλέπει δεν αντανακλώνται επαρκώς με τον ίδιο τρόπο. Χρειάζεται μεγαλύτερη υποστήριξη για τα αιτήματα αυτά. Ένα ή δύο θέματα για το Ταμείο Αντιμετώπισης Παγκοσμιοποίησης που έχει ε, ήδη προαναφερθεί. Συμφωνώ απόλυτα. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να λειτουργήσει αυτό χωρίς να υπάρχει γραφειοκρατική επιβάρηση και διοικητικές ε, επιβραδύνσεις. Πρέπει να μπορέσουν τα κράτη-μέλη όταν θα έχουν υποβάλει μια αίτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, βοηθηθούν. Πολλές φορές ε, δεν είναι σε θέση να ξεκινήσουν τέτοια προγράμματα τα κράτη-μέλη και δεν γίνονται πολλές φορές, δεν υλοποιούνται αυτά τα προγράμματα και δεν υπάρχει η δυνατότητα να ξεκινήσει η δρομολόγηση τέτοιων προγραμμάτων και σχεδίων σε σχέση με τα κονδύλια που θα διατεθούν αργότερα. Θα πρέπει αντίστροφα να γίνεται, να διατίθενται τα κονδύλια πρώτα. Και θα πρέπει να διασφαλίσουμε και εμείς από πλευράς Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο μηχανισμός δεν θα είναι πλέον αργός και, βρα... Ε, και Ευχαριστώ. Merci. Ε, Ευχαριστώ. Αναφερθήκαμε στην κοινωνική κρίση, λέει η κυρία Ντέλη. Όμως πρέπει να προσέξουμε συγχρόνως και τις κοινωνικές ε, ανισότητες. Και η κυρία Φιγκερίδα αναφέρθηκε σε αυτές. Αυτές λοιπόν οι ανισότητες εκρήγνεται όταν μιλάμε για αμοιβέ. Τι θα κάνουμε με αυτό. Δεύτερον, απασχόληση. Ξέρουμε ότι σήμερα όλο και περισσότεροι φτωχοί εργαζόμενοι υπάρχουν στην Ευρώπη. Οι νέοι, 20% της ανεργίας είναι μεταξύ των νέων. Άλλα θύματα βασικά αυτής της κατάστασης είναι οι γυναίκες. Τι θα κάνουμε λοιπόν, θα κάνουμε θα πάρουμε στρατηγική σημασία αποφάσεις για το τι θα κάνουμε ώστε να έχουμε πράσινη απασχόληση, αξιοπρεπή απασχόληση, που να εγγυάται κάποια ελάχιστα, κάποιες ελάχιστες κοινωνικές προδιαγραφές. Τώρα για τη λευκή βίβλο όσον αφορά τις ε, συντάξεις. Προσοχή, όλο και περισσότεροι συνταξιούχοι επίσης είναι φτωχοί τι θα κάνετε. Έχετε στοιχεία για το τι θα παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να καταπολεμηθεί η ένδια και ο κοινωνικός αποκλεισμός στην Ευρώπη. Πρόεδρος, ευχαριστώ και εγώ έχω να σας υποβάλω κάποιες ερωτήσεις. Για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Είπατε ότι το Συμβούλιο Απασχόλησης Κοινωνικής Πολιτικής Υγείας και Καταναλωτών, η ΕΦΣΚΟ, θέλει συστάσεις αναχώρα. Δώσατε την εντύπωση ότι η πρώτη αντίδραση από πλευρά των κοινωνικών εταίρων, από τα συνδικάτα, ήταν πολύ έντονη. Και ότι αυτό σιγά σιγά άλλαξε. Τώρα δέχονται να καθίσουν και να συζητήσουν όλα αυτά τα στοιχεία. Εγώ δεν ξέρω αν έτσι πρέπει να ερμηνεύσουμε τη στάση των κοινωνικών εταίρων και τη διάθεσή τους. Όπως και να έχει το πράγμα, με απασχολεί το εξή. Παράλληλα με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο έχουμε και το Σύμφωνο για το Ευρώ, που αγνοεί πλήρως τη Στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2020. Ένα παράδειγμα θα σας δώσω μόνο για τις διορθωτικές μεταρρυθμίσεις που προτείνονται συνεχώς. Αυτό που προτείνεται είναι η μείωση των μισθών, των συντάξεων αύξηση ηλικία ταξιοδότησης και κατάργηση των συμβάσεων απεριόριστου χρόνου. Όμως για μας, αν η στρατηγική Ευρώπη 2020 αποτελεί το σημείο αναφοράς για όλα αυτά, τότε θα έπρεπε να δούμε διαφορετικά τις δαπάνες μας όσον αφορά την εκπαίδευση. Και γιατί η μόνη εξαίρεση που μας επιτρέπει να δούμε την ε, ποιότητα των δαπανών και όχι μόνο το έλλειμμα. Έχει να κάνει με ε, συνταξιοδότηση μέσω κεφαλοποίησης. Μα εγώ πιστεύω ότι τα συστήματα εκπαίδευσης πρέπει να δείχνουν ακριβώς της ίδιας ε, προσοχής όπως και το καθεστώς συνταξιοδότησης. Δεύτερη παρατήρηση. Είπατε ότι όσον αφορά τους επιθυμητούς στόχους για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, υπάρχουν πράγματα που δεν έχουν αποφασιστεί ακόμα. Και μένει να δούμε αν θέλουμε προκαθορισμένους στόχους ή όχι. Όπως και εσείς δίχως άλλο, έτσι και εγώ ήρθα σε επαφή με πολύ κόσμο επιτόπου στις περιφέρειες και εμένα πολλοί μου είπανε, μα εμείς ανάλογα με την περιφέρειά μας πρέπει να κάνουμε αυτό που έχουμε να κάνουμε αν είμαστε ένας αστικός χώρος, έχουμε διαφορετικές δυσκολίες. Δεν θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε την στρατηγική 2020. Εμείς όμως εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είμαστε συνεπείς και συνεκτικοί. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εσείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δεν είναι μοιράζουμε χρήματα, είναι ένα εργαλείο για να πετύχει μια πολιτική, μια πολιτική συνοχής, έτσι τη λέμε, διαφθορωτικών ε, αλλαγών. Αν εγκαταλείψουμε κάθε ευρωπαϊκή διάσταση, τότε το μόνο που θα κάνουμε είναι απλώς και μόνο ότι θα κρατάμε το τομείο. Και τίποτα άλλο. Και θα συνεχίσουμε εκείνη τη λογική η οποία δηλητηριάζει την πολιτική μας από την εποχή της κυρίας Μάργαρετ Θάτσερ. Με εκπλήσει λοιπόν που τίθεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό το θέμα. Μα πώς το διάλογο θα εφαρμόσετε την στρατηγική 2020 με κοινωνικούς τόσο σημαντικούς στόχους, έτσι όπως έχουν αποφασιστεί αυτοί, αν δεν κινητοποιήσετε τα λίγα μέσα που έχετε στη διάθεσή σας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σας ρωτάω. Όσον αφορά το τη σφαιρική συμφωνία αναπεριφέρεια. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα τι ακριβώς σημαίνει αυτό για σας. Είναι μια σφαιρική συνολική συμφωνία που καλύπτει το σύνολο των ποσών και ΦΕΝΤΕΡ και Κοινωνικό Ταμείο μέσα σε μία και την ίδια σύμβαση και για την περιφέρεια τι σημαίνει ότι πρέπει να μάθει και πάλι ένα καινούριο μηχανισμό γιατί πολλοί από τους εταίρους μας επιτόπου μας λένε ότι έχουν δυσκολευτεί τόσο πολύ να εξοικειωθούν με τους μηχανισμούς. Εντάξει, δεν λέω ότι δεν πρέπει να αλλάξετε τίποτα, αλλά έχετε αξιολογήσει πόσο θα κοστίσει η εκμάθηση αυτού του νέου εργαλείου, του νέου μέσου που θέλετε να εφαρμόσουν οι περιφέρειες. Τέλος, για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες ή για τις πρωτοβουλίες γενικότερα στα πλαίσια της απόσπασης των εργαζομένων. Είπατε ότι εδώ υπάρχουν δύο πτυχές που αναφέρονται. Η κλασική που ο Μπαρός από την αρχή έχει δηλώσει για το πώς εφαρμόζει την νομοθεσία, αλλά μετά αναφέρεται και κάτι άλλο για τη Single Market Act. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα για αυτό το δεύτερο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Άκουσα να μιλάτε για το διάβολο. Άκουσα τίποτα αυτή τη λέξη εντάξει δεν λέω τίποτα παραπάνω. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, λέει ο κύριος Ρισελ. Δεν μπορώ να απαντήσω για την κρίση οικονομίας στην κυρία Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι σε δύο μήνες, 14 μέρες και δύο ώρες που είμαι σε αυτή τη θέση, δεν έχω ακούσει τίποτα γι' αυτό. Θα τα κοιτάξω. Είναι οι πιο ειλικρινές απάντηση που μπορώ να σας δώσω. Δεν ξέρω, θα ενημερωθώ. Για το πώς αντιλαμβάνονται οι πολίτες το τι συμβαίνει. Είμαστε σε μια επίσημη συνεδρίαση που περνάει στο διαδίκτυο, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, αλλά σας πω το εξή. Εδώ έξω υπάρχει ένας πραγματικός κόσμος και εδώ έξω ο κύριος ή η κυρία Αγορά παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Και πολλά πράγματα που έχουν συμβεί κατά το παρελθόν έχουν γίνει υπό την πίεση αυτής της ε, ασαφούς αγοράς. Η αγορά πρέπει να ικανοποιείται. Έχουν ληφθεί πολλά μέτρα. Και μπορεί κανείς να δει ότι προς το παρόν υπάρχει κάποια ισορροπία έτσι ώστε να ανακτάται εμπιστοσύνη και να μπορούμε να προχωρήσουμε. Φυσικά πρέπει να πληρωθούν και κάποιοι λογαριασμοί. Πώς ανακτάται η εμπιστοσύνη. Πληρώνουμε τους λογαριασμούς μας και αυτό. Πολλά λοιπόν από αυτά που έχουν αποφασιστεί και θα αποφασιστούν και από άλλες χώρες στα πλαίσια της λιτότητας θα οδηγήσουν σε ανησυχίες στον κοινωνικό τομέα. Πολλά από αυτά που έχουν γίνει από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με δεκαετίες διαπραγματεύσεων βρίσκονται υπό απειλή σήμερα. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί γι' αυτά. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να επαναλάβω αυτό που είπα και πριν, ότι ο κόσμος αλλάζει. Δεν μπορούμε να ε, σκεφτούμε ότι είναι πιθανό να γυρίσουμε στο σημείο που βρισκόμασταν πριν από την κρίση. Όχι. Πρέπει να δούμε που βρισκόμαστε σήμερα, να είμαστε καινοτόμοι και ελαστικοί διατηρώντας βέβαια ένα ουσιαστικό επίπεδο ευημερίας για όλους τους πολίτες, νέους και λιγότερο νέους. Αυτό είναι σαφές. Πρέπει να δουλέψουμε σκληρά γι' αυτό. Μέχρι σήμερα μπορείτε να πείτε ότι κάποιοι εταίροι ήταν διστακτικοί, δεν έδειξαν να θέλουν να συμμετέχουν στην συζήτηση και στις διαβουλεύσεις. Αυτό αλλάζει. Διαπιστώνουμε ότι αρχίζουν όλοι οι παράγοντες σιγά σιγά να είναι έτοιμοι και να θέλουν να μπουν στη συζήτηση. Με διαφορετική οπτική γωνία ίσως ο καθένας. Αλλά δεν υπάρχει λόγος έτσι καλλιώς να σκέφτεται κανείς ότι σύντομα θα φτάσουμε σε συνένεση. Πάντως αν μη τι άλλο ξεκινάει η συζήτηση και είναι πολύτιμο αυτό. Με τις πολιτικές μας και με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προσπαθούμε να προχωρήσουμε πολιτικές και να τις εφαρμόσουμε ώστε να δώσουμε σημασία σε όσους βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας, να συμπεριληφθούν στην κοινωνία κι αυτοί. Οι νέοι, για παράδειγμα, οι ηλικιωμένοι. Είναι ωραία να καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα ότι πρέπει κανείς να δουλεύει μέχρι μια μεγαλύτερη ηλικία, αλλά πρέπει να αλλάξουν και υποδομές γι' αυτό, να τους βοηθήσουμε τους ανθρώπους για να το πετύχουν αυτό. Και σε αυτό χρειαζόμαστε και το κοινωνικό ταμείο και βέβαια τη συνεργασία των κρατών μελών. Δεν θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης από την Ευρώπη. Μπορούμε να κάνουμε προτάσεις. Μπορούμε να κάνουμε αναλύσεις. Μπορούμε να δώσουμε στατιστικά δεδομένα. Μπορούμε να προσφέρουμε παραδείγματα, να πειραματιστούμε να κάνουμε καινοτομία στο κοινωνικό τομέα. Αλλά τα κράτη-μέλη θα βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα και θα εφαρμόσουν τις δικές τους πολιτικές. Ίσως να μην ήμουν σαφής ε, στην αρχή, κυρία Πρόεδρε, αν εσείς βγάλατε το συμπέρασμα ότι οι κοινωνικοί εταίροι ήδη συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Όταν αναφέρθηκα στους κοινωνικούς εταίρους είχε να κάνει με την οδηγία για το χρόνο εργασίας. Για αυτήν έχουμε κάποια δείγματα από τα συνδικάτα ότι θέλουν να συμμετάσχουν. Δεν λέω ότι δεν ενδιαφέρονται για το ευρωπαϊκό εξάμεινο, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει τίποτα. Εμείς ε, έχουμε ζητήσει από την Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας, από την ΕΜΚΟ και το ΕΦΣΚΟ. Και μετά θα υπάρξουν και άλλες, ε, και υπάρχουν και άλλες συναντήσεις όπου συζητάμε το μέλλον με τους κοινωνικούς εταίρους, αλλά όχι συγκεκριμένα το ευρωπαϊκό εξάμεινο ακόμα. Παρέμβαση εκτός μικροφώνου από την Πρόεδρο. Ναι, απαντάει ο κύριος Ρισελ. Έχει να κάνει με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, έχει να κάνει με το μέλλον του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου χωρίς όμως να υπάρχει συγκεκριμένη συνάντηση για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο μαζί τους. Τώρα να μην σας τα ξαναπώ, καταλαβαίνω ότι υπάρχει ανησυχία στο κοινωνικό τομέα. Εσείς λέτε, μα πρέπει να δούμε και τις επενδύσεις στην εκπαίδευση. Πολλές χώρες μέλη έχουν πολιτικές που δείχνουν ότι θέλουν να επενδύσουν περισσότερα στην εκπαίδευση. Και εμείς έχουμε την δικιά μας ημερήσια διάταξη για ε, νέα επαγγέλματα και θέλουμε να προχωρήσουμε στην επαγγελματική κατάρτιση με ελαστικό τρόπο, έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση όλοι. κυρίω αυτοί που δεν έχουν καμία επαγγελματική κατάρτιση, αλλά για να υπάρξει και επανακατάρτιση και το Ταμείο για τις επιπτώσεις από την παγκοσμιοποίηση συμμετέχει. Θέλουμε επίσης να προωθήσουμε και συμπληρωματική εκπαίδευση. είναι μεταξύ των στόχων της στρατηγικής για το 2020. Αλλά όπως σας είπα και πριν, ο προπολογισμό είναι περιορισμένος και συνεπώς δεν μπορούμε παρά να βασιστούμε στα κράτη-μέλη γιατί αυτά πρέπει να θέσουν τους στόχους τους για την εκπαίδευση. Σας έκανε εντύπωση, από την άλλη, το ότι συζητάμε και το κατά πόσο πρέπει να υπάρχουν ε, στόχοι ή όχι. Μα δείτε την πραγματικότητα για την περίοδο 2007-2013 δεν υπάρχουν προκαθορισμένοι στόχοι ούτε για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Συζητάμε με τις χώρες και τις περιφέρειες και από εκεί καταλήγουμε σε αποτέλεσμα. Αν ενδιαφέρονται έχει καλώς. Μπορούμε λοιπόν τώρα να πούμε ότι για την περίοδο 2017-2013, για αυτή την περίοδο σχεδιασμού, 22% του Ταμείου Συνοχής καταλήγει στο Κοινωνικό Ταμείο. ταμείο. Αλλά σε αυτό καταλήξαμε μετά από την συζήτηση που είχαμε με τις χώρες και τις περιφέρειες. Τώρα έχουμε όμως τη στρατηγική 2020 με στόχους. Γι' αυτό τίθεται το ερώτημα. Μήπως θα έπρεπε τα χρήματα τα οποία έχουμε για την περίοδο 2014-2020 να ε, είναι ανάλογα με τους στόχους, να ταιριάζουν περισσότερο με τους στόχους. Και αυτό είναι κάτι το οποίο συζητάμε με τις χώρες και με τις περιφέρειες. Είπατε και ίδια ότι συζητήσατε με τις περιφέρειες και έχετε τη δικιά σας εμπειρία, ότι σας είπανε δώστε μας τα χρήματα, εμείς ξέρουμε καλύτερα τι θα τα κάνουμε. Ναι, αλλά αυτό είναι μια πολιτική συζήτηση. Ο Επίτροπος Άνβορ λέει ξεκάθαρα ότι προτιμάει τα χρήματα να συνδέονται με τους στόχους έτσι όπως αυτοί καθορίζονται από τη στρατηγική 2020. Αλλά στη συνέχεια θα υποβάλει τις ιδέες της Επιτροπή τον Ιούνιο και μετά θα ακολουθήσει συζήτηση, στην οποία ελπίζω ότι και εσείς θα δραστηριοποιηθείτε. Για την απόσπαση των εργαζομένων τώρα, για την οδηγία αυτή, ρωτήσατε τι ακριβώς θα συμβεί με την, ε, πράξη, με την ενία πράξη. Την πράξη για την ενία αγορά, πιο σωστά. Κοιτάξτε, πρέπει να είμαι προσεκτικός εδώ. Κάτι θα γίνει. Δεν μπορώ όμως να σας πω τίποτα περισσότερο γιατί θα προκαταλάμβανα πολιτικές αποφάσεις. Πάμε από αποσαφήνιση μέχρι κάποια μορφή ρύθμισης, αλλά αυτό θα αποφασιστεί σε πολιτικό επίπεδο. Παρόλο που ο Γενικός Διευθυντής έχει πολύ ενδιαφέροντα ρόλο, ο ρόλος αυτός είναι παρόλα αυτά περιορισμένος και δεν θα ήθελα να εκφραστώ πολιτικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και προσδοκώ σε καρποφόρα και στενή συνεργασία μαζί σας. Κύριε Γενίκε, ο εισηγητής μας ε, έφτασε κάπως αργά, αλλά ε, δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε να παραμείνετε πέντε λεπτά ακόμα για να ακούσετε και την άποψη της εισηγήτριας. Κύριε Γενικέ, ζητώ συγγνώμη για την ε, καθυστέρησή μου. Βρισκόμουν σε μία ε, διαπραγμάτευση. Ζητώ την κατανόησή σας. Συμφωνώ απόλυτα με την Πρόεδρο της Επιτροπής Απασχόλησης για την ανάγκη μιας ευρωπαϊκής πολιτικής για το ΕΚΤ και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δεν θα πρέπει να προωθεί περιφερειακές ε, πολιτικές όπου δεν θα υπήρχε ένα ευρωπαϊκό πνεύμα που να διέπει αυτές τις πολιτικές. Κατανοούμε βεβαίως ότι χρειάζονται προσαρμογές τοπικού χαρακτήρα για όλα. Είπατε όμως ότι 22% του Ταμείου Συνοχής κινείται προς τον κοινωνικό τομέα, όμως ο κοινωτικός προϋπολογισμός δεν είναι τόσο εκτεταμένος. Υπάρχουν ε, ε, μεγάλες ανάγκες και τα μία που είναι πιο, ε, πιο συνεκτικά, πιο περιορισμένα σε σχέση με αυτή την περίοδο κρίσης. Τι θα γίνει σε αυτή την περίοδο επιπτώσεων. Δεν χρειάζονται μόνο χρήματα επιτόπου ή στον κοινωνικό τομέα. Θα πρέπει τα κονδύλια να δοθούν σε άνδρες και γυναίκες που τα χρειάζονται. Και θα πρέπει να ορίσουμε μία πολιτική, ευρωπαϊκή πολιτική άναντι και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να επαληθεύσουμε επιτόπου ώστε να λειτουργήσει αυτό το, το μέτρο ως μοχλός δράσης. Δηλαδή να μην ελέγξουμε τον ε, τύπο, αλλά τις επιπτώσεις. Γιατί αυτός είναι ο απότερος πολιτικός μας στόχος. Απάντηση. Ως προς το θέμα των ε, σαφών κοινωνικών στόχων, νομίζω ότι για πρώτη φορά είμαστε σε θέση να διασυνδέσουμε τις δαπάνες του ΕΚΤ, αν ε, υπάρξει πολιτική απόφαση, σε συγκεκριμένα μέτρα, με συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία ορίζονται στην στρατηγική 2020. Έτσι θα έχουμε έναν οδηγό χρήσης, θα δώσουμε έναν οδηγό χρήσης προς τα κράτη-μέλη, από όπου θα επιλέξουν τα σημαντικά στοιχεία και ό,τι και να επιλέξουν θα πρέπει να βασίζεται σε αυτό το, το, τον οδηγό χρήσης κατά κάποιο τρόπο. Ως προς τις επιπτώσεις, των χρημάτων που χρησιμοποιούνται υπάρχει μια σειρά αξιολογήσεων. Το θέμα είναι η γενίκευση αυτών των αξιολογήσεων και είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί αναπεριφέρεια τα πράγματα μπορεί να διαφέρουν άρδιν. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να έχουμε μια καλύτερη ανάλυση του τι έχει γίνει με τα χρήματα του παρελθόντος. Μπορούμε να σας αποστείλουμε εκατοντάδες σελίδες αποτιμήσεων με πολύ μικρό αποτέλεσμα, αλλά δεν αποζητάτε κάτι τέτοιο. Θέλετε μία μελέτη αντικτύπου αναχώρα τουλάχιστον. Και αυτό προσπαθούμε να συντάξουμε. Δεν είναι εύκολο να γίνει, διότι όλες οι εκθέσεις έρχονται υπό διαφορετική μορφή και θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι αυτό που δημοσιοποιούμε ε, ευσταθεί επιστημονικά. Δεν μπορώ να σας υποσχεθώ πότε θα είναι διαθέσιμο. Θα γίνει μία μελέτη αντικτύπου για, ως προς τις ε, αποδόσεις του παρελθόντος. Αλλά αυτό θα προωθηθεί κατά τον Ιούνιο. Συντοπιώ ότι δεν απάντησα σε ένα ερώτημα της ε, Προεδρού ε, σε σχέση με τις ε, συμβάσεις. Αυτό που θα θέλαμε στο μέλλον είναι να γίνει μία διαπραγμάτευση με ένα κράτος μέλος ή περιφέρεια σε σχέση με, όλα, με όλους τους ε, πόρους έτσι ώστε να μην έχουμε θεματική προσέγγιση για αυτή την περιφέρεια ή χώρα αλλά να ορίσουμε ποιες δραστηριότητες θα χρηματοδοτηθούν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί, για παράδειγμα τώρα, αν αποφασίσουμε να χρηματοδοτήσουμε την επαγγελματική κατάρτιση, πολλές φορές χρειάζονται σχολεία. Αλλά εμείς ε, δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε οι υποδομές. Γι' αυτό θα πάμε σε ένα άλλο ταμείο για να ζητήσουμε τα χρήματα υποδομών. Αυτό είναι ένα δυσχύριστο πλαίσιο. Άρα έχουμε τη Στρατηγική Ευρώπη 2020, μετά έχουμε τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων, τα οποία θα συζητήσουμε με τις χώρες κατά το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και στη συνέχεια θα γίνει μια συζήτηση με τις χώρες για την εφαρμογή αυτή που θα ορίσουμε τις διάφορες δραστηριότητες. Και αναδραστηριότητα θα πρέπει να υπάρχει μία ενιαία εφαρμογή. Με αυτή την τάξη και σειρά θα δούμε τα πράγματα. Ευχαριστούμε τον Γενικό Διευθυντή, όπως είπατε. Θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες να συζητήσουμε αυτά τα θέματα, να τα διαπραγματευτούμε, αλλά είναι πολύ σημαντικό το ότι είχαμε μία πρώτη ανταλλαγή απόψεων και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις μελλοντικές σας δραστηριότητες που είναι ύψης της σημασίας και για εμάς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πρόεδρος, στρεφόμαστε στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης και δίνω το λόγο στον κύριο Μάρτιν Κάστλερ για να μας παρουσιάσει την πρόταση νομοθετικού περιεχομένου για το Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργούς Γύρανσης που θα είναι το 2012 θα συζητήσουμε τις 25 τροπολογίες συμβιβασμού ε, με βάση τις αρχικές 150 γνωρίζοντας ότι υπάρχει και ένα δημοσιονομικό θέμα διότι μας προτείνεται ένα έτος χωρίς χρήματα. Έχει λόγο κύριε Σιγητά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το θίξατε το ένα θέμα ήδη, ένα θέμα κέρια σημασίας αυτό τον προϋπολογισμό, τα κονδύλια και το θέμα του όταν έχουμε ένα ευρωπαϊκό έτος 2012 αλλά δεν έχουμε κονδύλιο γι' αυτό δυσχεραίνονται τα πράγματα, δυσκολεύουν. Και από ό,τι γνωρίζουν η δεύτερη φορά στην ιστορία των ευρωπαϊκών ετών που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και νομίζω καλό θα ήταν εμείς ως Ευρωκοινοβούλιο να δείχναμε ποια είναι η θέση, η τοποθέτηση που υιοθετούμε. Και αυτό συνδέεται και από κοινού με τους σκιώδους εισηγητές όλων των κοινοβουλευτικών ομάδων που σε αυτή τη θέση θα ήθελα τώρα σε αυτή, από αυτή τη, στιγμή να ευχαριστήσω όλους για την καλή συνεργασία που είχαμε και έτσι το μεγάλο αριθμό τροπολογιών καταφέραμε τον συρρυκνώσουμε στις συμβαστικές τροπολογίες που προαναφέρατε. Ευχαριστώ λοιπόν όλους τους σκιώδους εισηγητές. Νομίζω έχει νόημα να υπάρχουν αυτοί οι συμβιβασμοί με τον τρόπο και τη μορφή που έχουν τώρα μπροστά σας κάποια σημαντικά σημεία επιτρέψτε μου να αναφέρω που εγώ συγητής θεωρώ ότι είναι σημαντικά για μένα. Θα ήθελα να τα αναφέρω ξεχωριστά. Ο πρώτος τομέας είναι φυσικά σαφής. Η πρόταση δηλαδή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει την απαρχή της και τον κύριο στόχο της ε, την ενεργό γύρανση λαμβάνοντας, εντάσσοντας την στην πολιτική για την αγορά εργασίας. Εμείς ως Ευρωβουλευτές διευρύναμε αυτή την προσέγγιση και ήδη στη συζήτηση τα συζητήσαμε και με συνένεση ομόθυμα τα έχουμε οδηγήσει σε αυτές τις συμβιβαστικές τροπολογίες. Δεν πρόκειται λοιπόν μόνο για πτυχές της αγοράς εργασίας. Πρόκειται για μια μεταξύ των γενεών εργαζομένων και με την αλληλεγγύη των ε, γενεών μια προσέγγιση για μια ενεργό γύρανση του πληθυσμού. Για κάτι πολύ περισσότερο δηλαδή από ότι μόνο η πολιτική για την απασχόληση της αγοράς εργασίας. Έχουμε εδώ ένα πολύ ευρύτερο πεδίο για την διαβίου ε, μάθηση ε, για την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και άλλα συναφή τέτοια θέματα. Και αυτός ο ορισμός για μια αηφορία στην, ε, στον πολιτισμό, στην προσέγγιση της γύρανσης θέλουμε με τον τίτλο να το εκφράσουμε αυτό. Και είναι το πρώτο σημείο που θέλω να εκφράσω. Ότι θα έχουμε μια δεσμευτική κοινή γραμμή πορεία στην οποία δεσμευόμαστε Κοινοβουλευτική Επιτροπή και ευχαριστώ όλου για, για αυτό, ιδιαίτερα του κοιόδης εισηγητέ. Ένα πολιτισμό λοιπόν τη ενεργού γύρανση ε, μεταξύ αλληλεγγύη των γενεών και μια ε, δραστήρια γύριση. Αυτό πρέπει να είναι ο τίτλο ε, όταν εξετάζουμε αυτό το θέμα και τι συμβαστικέ τροπολογίε. Ευρωπαϊκό Έτο ενεργού γύρανση και αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Με ένα υπότιτλο διατηρώντας ε, την ε, ε, θα έλεγα ζωντάνια όλων. Αυτά εκφράζουν την αξιοπρέπεια όλων που πρέπει να διασφαλιστεί, η αναζωογόνηση όλων, ζωντάνια όλων που πρέπει να διασφαλίζεται, άσχετα ποιοι είναι αυτοί, εντάσσονται όλες οι γενναίες μέσα σε αυτό το πλαίσιο που θα πρέπει να εκφράζονται υπέρ της ενεργογύρανσης, όχι μόνο για τις πιο ηλικιωμένες γενναίες, αλλά και τις νεότερες γενναίες που και αυτές σιγά σιγά γερνούν. Δεύτερο σημαντικό θέμα, προϋπολογισμός, κονδύλια. Λοιπόν, νομίζω είναι χωρίς καμιά αμφιβολία ότι είναι αναγκαίο να διασφαλίζονται κονδύλια δηλαδή πόροι δημοσιονομικά, ώστε να καταφέρουμε ένα ευρωπαϊκό έτος για την γύρανση να το προωθήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί διαφορετικά δεν έχει καμιά δυνατότητα να σταθεί στα πόδια του κάτι τέτοιο. Η κοινή θέση που καθορίσαμε στις, ε, σε, στις συμβαστικές τροπολογίες και ευχαριστώ όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες θερμά, διότι ήταν το πιο επίμαχο σημείο αυτό. τι κονδύλιο θα ήταν δηλαδή αυτό, ποια χρήματα θα δινόντουσαν έτσι έχουμε λοιπόν ένα σταθερό κονδύλιο ελέγξιμο 6 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτή την πρωτοβουλία. Τι σημαίνει αυτό και ευχαριστώ για την ε, προσπάθεια αυτή και την διάθεση ε, της επιστολής του συναδέλφου Λαμασούρ που ε, διανεμήθηκε ή διανέμεται για αυτό το 2 εκατομμύρια για εφέτος και η αρχική αυτή εκκίνηση και μετά για το 2012 άλλη μία φορά μία δόση 4 εκατομμυρίων, σύνολο 6, ώστε να είναι ε, ε, θα έλεγα ευδιάκριτος ο χαρακτήρας των δράσεων και των εκδηλώσεων αυτού του έτους ώστε κάπως να μας ικανοποιεί ποτέ δεν υπάρχουν τα κονδύλια. Θα θέλαμε να είχαμε περισσότερα, όπω έχει προταθεί, είχε προταθεί και από συναδέλφου. Αλλά 6 εκατομμύρια σε ένα σταθερό δημοσιονομικό πλαίσιο ω κονδύλιο, γιατί όπω είπαμε στο, το κυριότερο σημείο στι συζητήσει με την Επιτροπή και το Συμβούλιο ήταν, δεν ήταν ότι πρόκειτο για συγχρηματοδότηση, αλλά για καθαρά 6 εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια για φέτο και 4 εκατομμύρια για του χρόνου 2012. 6 σύνολο. Αυτά η περίληψή μου συνολικά εισαγωγικά. Αυτά για τον συμβιβασμό από πλευρά μα. Ελπίζω ότι θα είναι δυνατόν να υπάρξει συνένεση από πλευρά σα σε ευρύτερο πλαίσιο και αύριο σχετικά γοργά να μπορέσουμε να εγκρίνουμε και να προχωρήσουμε. Όπω και από πλευρά μα είναι σημαντικό να γίνει. Θέλουμε αυτό το Ευρωπαϊκό Έτο Ενεργού Γύρανση και Αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών να προχωρήσει 2012, να προετοιμαστεί σωστά και να ξεκινήσει σωστά. Δηλαδή το δυνατόν πιο γοργά να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτό το χαρτοφυλάκιο. Αν τώρα θα γίνει σε μια πρώτη ε, ανάγνωση και συμφωνία και τα καταφέρουμε ή όχι θα το δούμε μετά την ψηφοφορία, θα το ξέρουμε και θα σφιγμομετρήσουμε με το Συμβούλιο και την Επιτροπή τι θα γίνει. Αλλά κατά τούτο πρέπει να θέσουμε εντάξει τα, των θεμάτων αυτών, διότι μπορεί η μία ή άλλη συζήτηση του ενός ή άλλου θέματος να είναι αναγκαία. Αλλά υπερκομματικά ως Ευρωκοινοβούλιο θέλουμε να δώσουμε ένα μήνυμα. Προς τα πού θα πορευθούμε σε αυτό το ταξίδι με το Ευρωκοινοβούλιο, ποια θα είναι η πορεία μας. Ευχαριστώ και θα το κάνουμε αυτό αύριο. Και χαίρομαι και για τη συζήτηση αυτών των θεμάτων. Ευχαριστώ. Euh, Madame Rovana puis Η κυρία Ρωμάνα Πλόμπ και μετά ο κύριος Μαν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να εκφραστώ εκ μέρους της συναδέλφου Κορίνα Κρέτσου που είναι σκιώδης συζυγήτρια, αλλά δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα. Η κυρία Κρέτσου λοιπόν συγχαίρει τον κύριο Κάσλερ για την έκθεσή του και για την επιμονή του όσον αφορά τις διάφορες γραμμές του προπολογισμού για το Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργούς Γύρανσης και Ζωτικότητας. Θα ήθελα λοιπόν να σας μεταφέρω από την κυρία Κρέτσου ταξί. Είναι πολύ ικανοποιημένη για το ότι πετύχαμε συμβιβασμούς σε σημαντικά σημεία της έκθεσης αυτής και θεωρεί ότι επιβάλλεται πιο ευθύς τρόπος χρήσης των ε, πιο μεγάλων εργαζόμενων, γιατί έχουν εμπειρία από την οποία δεν αποφελούμαστε αρκετά. Αντίθετα, υπάρχει διάκριση σε βάρος τους, που πρέπει να καταπολεμηθεί πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένα μέτρα που να διασφαλίζουν ισορροπία ανάμεσα στην ε, αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και μια μεταρρύθμιση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Επίσης, εκτιμάει η κυρία Κρετσού το γεγονός ότι ο κύριο Κάσλερος εισηγητής επιμένει για το ότι ανάμεσα στους τρεις πυλώνες όπου βασίζεται η Ευρωπαϊκή Αποστολή συμπεριλαμβάνεται η γύρανση μαζί με την αξιοπρέπεια και την αλληλεγγύη. Η κυρία Κρέτσου στηρίζει το ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε τι έχουν προσφέρει οι ηλικιωμένοι στις κοινωνίες μας. Και αυτό να φαίνεται στα ταμεία τα συνταξιδιωτικά και ε, κοινωνικής ασφάλισης οι ηλικιωμένοι δεν θα πρέπει να βλέπουν να μειώνονται οι συναντάξει του ή να μην μπορούν να αγοράσουν τα φάρμακά τους όπω συμβαίνει στη Ρουμανία για παράδειγμα. Από την άλλη πιστεύει ότι πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στην οικονομική κρίση και στα μέτρα λιτότητας που πλήττουν ευαίσθητες κατηγορίες του πληθυσμού όπως είναι οι γυναίκες Γυναίκε οι οποίες είναι θύματα πολλαπλών διακρίσεων. Τέλος, πιστεύει ότι πρέπει να υπογραμμίσουμε πως η κοινωνική προστασία δεν είναι αναγκαία μόνο για τους ηλικιωμένους, αλλά είναι μια υποχρέωση και αποτελεί και το βαρόμετρο λίγο πολύ ε, με το οποίο μετράμε μια κοινωνία, από το πόσο δηλαδή σέβεται αυτούς που έχουν προσφέρει τη ζωή τους για διάφορους στόχους. Ο κύριος Μαν τώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Μαρτιν Κάστλα για την έκθεση που έχουμε. Και αν δει κανείς αυτές τις 159 τροπολογίες, είναι κατευθύνονται προς κοινή κατεύθυνση όλες. Δηλαδή είναι όλες υπέρ του να ενταχθεί αυτό το θέμα στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Χαίρομαι και για το ότι θα έχουμε την δικαιοσύνη και αλληλεγγύη των γενεών. Ένα αίτημα ήταν ότι το 2012 πρέπει να είναι το έτος ενεργούς γύρανσης. Όμως είναι πολύ σημαντικό και αυτό το οποίο αναφέρθηκε και ευχαριστώ όλους ε, ότι πρέπει να διευρυνθεί όπως είπαμε το ε, θέμα με την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Είναι θεμελιώδους σημασία θέμα. Το βλέπουμε και το ζούμε τώρα αυτό μέσα στο πλαίσιο τη παρουσία τη έκθεση. Όχι μόνο στην εκλογική μου περιφέρεια, όχι μόνο στη Γερμανία. Να επισημαίνουμε πόσο σημαντικό είναι ότι πρέπει να διευρύνουμε όταν έχουμε νέους να μην έχουμε μόνο τα θέματα των νέων και όταν έχουμε ενώσεις ε, ε, υπερηλίκων να έχουμε μόνο δικά τους θέματα. Να γίνει από κοινού μεταξύ των γενεών η προσπάθεια αυτή. Να γνωρίζουμε ότι πρώτον η αλληλεγγύη πρέπει να εκφράζεται και δεύτερον να μεριμνούμε ότι θα διασφαλίζεται και η χρηματοδότηση. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει μόνο θετικά. Από κοινού να δράσουμε. Και έτσι έχουμε μια σωστή προσέγγιση συνολικά. Και όταν το έτος 2012 θα το χρησιμοποιήσουμε γι' αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλο αυτό. Δηλαδή να μην παραμείνουμε σε ένα στενότερο πλαίσιο μόνο για μας με εσωστρέφεια αλλά να περάσουμε προς τα έξω. Προαναφέρθηκε αυτό ότι δεν πρέπει μεταξύ μας να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Με το web streaming περνάμε προς τα, τα έξω ούτως ή άλλως στη συνεδρίασή μας. Να έχουμε λοιπόν απήχηση προς τα έξω. Εμείς να μεταφράσουμε έτσι αυτό το έργο που θα γίνει και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο ώστε να είναι ελέγξιμα αυτά και να ξέρουμε τι γίνεται, να είναι υποέλεγχο και να ξέρουμε πώς θα υλοποιηθούν με σωστό τρόπο. Νομίζω με αυτό θα έχουμε μια πολύ καλή βάση λοιπόν. Ένα θέμα κάπως με προβληματίζει ακόμα. Αλλά υπάρχει ένας κοινός συμβιβασμός. Είναι το θέμα των κονδυλίων, των πόρων. Στην τροπολογία μου 77 επεσήμανα και είπα ποια κονδύλια το 2010 είχαμε στη διάθεσή μας. Και ξέρουμε ότι ήταν το έτος καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Είχαμε 17 εκατομμύρια ευρώ τότε στη διάθεσή μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από αυτά 9 εκατομμύρια δόθηκαν για μέτρα στα κράτη-μέλη και 8 εκατομμύρια από αυτά για ευρωπαϊκά μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και είπαν τα κράτη-μέλη από τα δικά τους κονδύλια θα ήθελαν να μεριμνήσουν άλλα 9 εκατομμύρια να διασφαλιστούν. Είναι νομίζω ποσά και το ότι ζήτησα 20 εκατομμύρια ίσως ε, δεδομένης ε, της κατάστασης αυτής, σε αυτή την κατάσταση οφείλεται. Ζητάμε κάτι που εντωμεταξύ ήταν κάτι παραπάνω, θα ήταν κάτι παραπάνω από τα 6 εκατομμύρια. Πήρα την επιστολή της 9ης Δευτέρου από τον κύριο Λαμασού προς την πρόεδρό μας, κυρία Μπερές, και αναφέρεται σε αυτή την επιστολή, δηλαδή 4 ε, ε, εκατομμύρια θα είναι 2 εκατομμύρια τώρα και μετά 4, σύνολο 6. Είχα, θα είχα την παράκληση, μια και καταλήγουμε σε ένα συμβιβασμό μεταξύ των ομάδων, να πούμε τουλάχιστον 6 εκατομμύρια κονδύλια θα διασφαλιστούν, θα διατεθούν. Διότι θα, μπορούσε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι στις διαπραγματεύσεις με τους φίλους μας στην Επιτροπή Προϋπολογισμών υπάρχει, υπάρχει κάποια, κάτι, κάποια επιφύλαξη, κάποιο αποθεματικό. Δεν είναι μόνο τα κονδύλια το σύνολο. Όταν συζητάμε τέτοια θέματα, όταν έχουμε μία, ας το πω έτσι, ποιότητα στην επικοινωνία και διαθέσουμε με αυτό, διασφαλίσουμε με αυτή την προσπάθεια τα κονδύλια. Δηλαδή να πούμε πρέπει να έχουμε επαρκή κονδύλια να δράσουμε. Παράκληση να πούμε τουλάχιστον 6 εκατομμύρια να διατεθούν για, αυτή την προσπάθεια. Ε, και έτσι θα μειωθούν βέβαια από τα 20 τόσα εκατομμύρια που είχαμε, εμείς είχα εγώ αρχικά προτείνει, αλλά εκφράζεται έτσι η πρόθεση που θέλουμε να υλοποιήσουμε. Ευχαριστώ. Θα σας δώσω στο τέλος της συζήτησης το λόγο κύριε Σιγητά. Έχω ακόμα όμως την κυρία Ίσιο και μετά εσείς. Ευχαριστώ. Μιλάω εκ μέρους του κύριου Κατσίν, σκιώδους εισηγητή. Ευχαριστούμε τον εισηγητή για τη συνεργασία του, για τη συνενετική του διάθεση, το οποίο καταλήξαμε στις 27 συμβασμούς που θα στηρίξουμε. Όπως είπαμε και στην αρχή, πρέπει να συμπεριλάβουμε επιπλέον εκπαίδευση και κοινωνικές δραστηριότητες όπως και πολιτιστικές δραστηριότητες και αθλητισμό για να ενισχύσουμε την ε, ζωή των ηλικιωμένων, τα οποία θέλουμε να παραμείνουν ενεργά όσο γίνεται περισσότερο. Όλες αυτές οι δραστηριότητες βοηθάν τους ε, ανθρώπους, ακόμα και όταν έχουν λιγότερο δραστήρια, λιγότερες δραστηριότητες στον οικονομικό ταμέα, να κρατάνε το ενδιαφέρον τους και να συμμετέχουν στην ε, ζωή. Πιστεύουμε ότι διαφορετικές τάσεις που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτούν ε, τοπική προσέγγιση. Στο χαμηλό επίπεδο ε, πρέπει να λαμβάνονται οι αποφάσεις για τους ηλικιωμένους. Έχουμε τις προτάσεις Κώστας που πιστεύουμε ότι προσφέρουν μια καλή ισορροπία. Πρέπει να ελέγξουμε βέβαια και τα οικονομικά του έτους αυτού. Τα 6 εκατομμύρια ευρώ είναι ένα ικανοποιητικό ποσό και η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη έχουν προχωρήσει αυτό. Στηρίζουμε επίσης το συμβιβασμό που περιλαμβάνει και έναν υπότιτλο και ελπίζουμε να επιτευχθεί συμφωνία με το Συμβούλιο, ώστε οι προετοιμασίες για το Ευρωπαϊκό Έτος Γύρανσης του 2012 να προχωρήσουν όσο γίνεται καλύτερα. Ευχαριστούμε, η κυρία Λάμπερτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την καλή συνεργασία που είχαμε μεταξύ μας σε αυτή την υπόθεση. Θέλω επίσης να επαναλάβω και αυτό που είπε η κυρία Χέρς, δηλαδή να λυθεί γρήγορα το ζήτημα, ώστε να έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας να προετοιμαστούμε για αυτό το ευρωπαϊκό έτος. Είναι το συνήθως παράπονο εδώ. Τα ευρωπαϊκά έτη που αποφασίζουμε υποφέρουν από ελλειπή σχεδιασμό και άρα υποφέρει η ποιότητά τους. Κρίμα. Και αυτό έχει να κάνει και με το οικονομικό ζήτημα βέβαια. Πόσα χρήματα έχουμε στη διάθεσή μας πρέπει να πρωτοστατεί η δικιά μας η Επιτροπή. Εδώ σας πενθυμίσω τροπολογία 75 στο 14α προκειμένου να έχουμε μια καλή προσέγγιση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να σας πω ότι η ομάδα μας καταλαβαίνει και συμφωνεί με όσα είπε ο Τόμας Μαν πριν από λίγο γιατί πολλά από αυτά τα ευρωπαϊκά έτη ε, προχωράνε και προσπερνάνε χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Θα υπάρξουν και άλλες τροπολογίες με τις οποίες ζητάω να βρούμε τρόπο χρηματοδότησης και για άλλες δραστηριότητες. Ε, σε ρευστό ίσως για διάφορα δίκτυα τα οποία πιέζονται οικονομικά. Κάτι άλλο που θα θέλαμε να δοκιμάσουμε είναι η ποικιλομορφία ποιοι συμμετέχουν. Να φροντίσουμε να συμμετέχουν όσο γίνεται περισσότερες ομάδες πολιτών, όχι μόνο διαφορετικές γενιές, αλλά που να προέρχονται και από διαφορετικούς τομείς της κοινωνίας. Χαίρομαι λοιπόν για ε, την άποψη του εισηγητή όσον αφορά τις τροπολογίες μας, που τη συμπεριλαμβάνει, όπως είπε, στους ε, συμβιβασμούς που και εμείς είμαστε διατεθειμένοι να στηρίξουμε. Για το σημείο 2 γίνονται ενδιαφέρουσε προτάσεις από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Πώς θα συμπεριληφθούν όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, ώστε να προωθηθούν ιδέες που περιλαμβάνονται στην πρότασή μας. Κάτι άλλο που υπάρχει στις συμβαστικές τροπολογίες είναι μία συνέργεια μεταξύ των διαφόρων ετών που οργανώνουμε και αυτό θα το στηρίξουμε. Δεν λέω πολλές φορές θετικά πράγματα για τη χώρα μου, αλλά αυτή τη φορά έγιναν προσπάθειες για μια μετάβαση από το Ευρωπαϊκό Έτος ένδιας στο Ευρωπαϊκό Έτος για τον Αθλητισμό. Οπότε και εδώ πρέπει να συμπεριληφθούν όλα τα επίπεδα διακυβέρνηση και στο έτος αυτό για την γύρανση. Ας δούμε εμείς ως Κοινοβούλιο τι μαθήματα έχουμε ήδη πάρει και πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε και εδώ. Ευχαριστούμε. Εισηγητή για γνωμοδότηση από την Επιτροπή Πολιτισμικών Υποθέσεων, ο κύριο Στάκουλα είναι εδώ. Θέλετε να πάρετε το λόγο εκ μέρου τη Επιτροπή σα. Ευχαριστώ εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού. Θα ήθελα και εγώ να πω λίγα λόγια σε σχέση με την έκθεση Μάρτιν Κάσλερ σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργούς Γύρανσης. Καλύτερα να το κάνω φιλανδικά, γι' αυτό βάλτε τα ακουστικά σας και θα συνεχίσω στα φιλανδικά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Κάστλερ για την εξαιρετική έκθεση και για το γεγονός ότι δέχτηκε τα όσα του ανέφερε η Επιτροπή Πολιτισμού. Το αναγνωρίζουμε αυτό και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Ελήφθη υπόψη το πολιτισμικό αυτό πλαίσιο. Μιλάμε για αθλητισμό, για φυσική αγωγή, την σημασία του πολιτισμού για την ευημερία των ανθρώπων και εδώ μιλάμε για το πνευματικό τομέα τόσο και όχι για τη φυσική ευεξία. Επίσης, η... ο εθελοντισμός έχει μεγάλη σημασία και η διαβίου μάθηση. Όλα αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στις διάφορες ηλικίε, στο ηλικιακό φάσμα και ο εισηγητής γνωρίζει ότι και η γύρανση μπορεί να είναι ένας παράγοντας συνεισφοράς. Και αυτός είναι ένας πολύ καλός θεματικός στόχος. Πρόεδρε, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε στους πολιτικούς που λαμβάνουν αποφάσεις ότι θα πρέπει να υπάρξει μία μεταστροφή ως προς την, ε, τις ιδιοσυγκρασίες. Δηλαδή, μιλάμε για το ηλικιακό φάσμα μεταξύ 25 και 55, που είναι η ενεργός γύρανση. Αυτή είναι η περίοδος ενεργούς γύρανσης, τουλάχιστον μέχρι τούδε. Αλλά ο βασικός στόχος ε, δεν είναι να αυξήσουμε το ΑΕΠ στην Επιτροπή Απασχόλησης. Υπάρχουν και άλλα σημαντικά θέματα στη ζωή των ανθρώπων και η ίδια η ζωή είναι ένα πολύ σημαντικό δώρο. Άρα, ε, για όσους αφήνουν την ενεργό φάση πίσω τους, θα πρέπει να αποτιμήσουν τις εμπειρίες τους και να τους σεβόμαστε και σαν ανθρώπους για τη μελλοντική τους πορεία. Δηλαδή θα πρέπει από πνευματικής ε, πλευράς και από πλευράς φυσικής ευεξίας να μπορούν να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα, να νιώθουν ότι τους έχουν ανάγκη οι άλλοι άνθρωποι Αυτό που έχει σημασία είναι να αγαπάμε τους ανθρώπους ως ενεργά μέλη της κοινωνίας και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό και για τον γυράσκοντα πληθυσμό. Θα μπορούσα να σας πω πολύ περισσότερα ή να γράψω πολύ περισσότερα. Ο κύριος Κάσλερ προσπαθεί να βελτιώσει την ποιότητα αυτού του εγγράφου και χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτό το συμβιβασμό και γιατί λάβατε υπόψη τις δικές μας απόψεις. Χαίρομαι που υπάρχει αυτό το θεματικό έτος. Ελπίζω να μην παραμείνει νεκρό γράμμα, αλλά να έχει επίπτωση στη στάση των ανθρώπων απέναντι στη ζωή. Δηλαδή να σεβόμαστε περισσότερο τον γυράσκοντα πληθυσμό. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω κατά πόσο ο εισηγητής θέλει να μας μιλήσει, να μας πει ορισμένα συμπεράσματα από τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Ουσιαστικά δύο παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω μόνο. Πρώτον, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια μπορώ να επιστρέψω τους επένους και μένα μου έκανε μεγάλη χαρά αντίστροφα να εργαστώ ώστε να καταλήξουμε σε συμβιβασμούς για αυτήν την έκθεση και γι' αυτό ευχαριστώ θερμά. Νομίζω κατανόησα σωστά και την, τον κύριο Τόμασμαν Μαν και την συνάδελφο κυρία Λάμπερτ όσον αφορά τις ε, τροπολογίες τους που πάνε πιο πέρα τις αποσύρουν και είναι υπέρ των συμβιβασμών με προφορική τροποποίηση ώστε at least, ε, τουλάχιστον να πούμε τουλάχιστον 6 εκατομμύρια ευρώ απαιτούμε. Σωστό αυτό από πλευρά ερμηνεία μου. Αν είναι σωστό, ευχαρίστω να το εντάξω και σε σχέση με τη γραμματεία θα το εντάξουμε. Να ρωτήσω Ποιος θα θέσει αυτή την προφορική τροποποίηση, ποιος θα την διατυπώσει, πώς θα γίνει διαδικαστικά κάτι τέτοιο. Ωραία, υστερότερα μπορούμε να το αποσαφηνίσουμε. Και κατά τα άλλα ευχαριστώ και την Επιτροπή Πολιτισμού, δεύτερη παρατήρηση αυτή, για σημαντικές προτάσεις που δώσατε κύριε Τάκουλα, ώστε έτσι να είναι ολοκληρωμένη η εικόνα τώρα και θα έρθουμε σε επαφή ώστε να είναι πλήρηση. Ε, προσέγγιση αυτή. Αύριο στην ψηφοφορία θα μπορέσουμε νομίζω με απλό τρόπο χωρίς να υπάρχει επιβάρυνση να ολοκληρώσουμε όσον αφορά τις διαδικασίες με την ψήφιση της Επιτροπής μας και μετά με το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ολοκληρώσουμε σύντομα όταν υπάρχει ομοθυμία για το κονδύλιο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Τα σχόλια της κυρίας Λαμπέρ θα ληφθούν υπόψη θα έχουμε και τον κατάλογο ψηφοφοριών που θα διανεμηθεί απόψε. Θα ψηφίσουμε αύριο γιατί υπάρχει και μια προφορική τροπολογία για να λάβουμε υπόψη την συμφωνία που επήλθε. Θα ψηφίσουμε λοιπόν αύριο την έκθεσή σας κύριε Κάσλερ και θα δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε μέχρι την Ολομέλεια του Μαΐου. Και να φτάσουμε σε μια συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Περνάμε στο σημείο 6, Ευρωπαϊκή Συνεργασία στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για την υποστήριξη της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Θα εξετάσουμε τις ε, τροπολογίες συμβιβασμού στην έκθεση της κυρίας Νάντια Χίρς. Έχετε το λόγο για να μας ε, παρουσιάσετε τις 13 τροπολογίες συμβιβασμού. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ θερμά επίσης τους σκιώδη εισηγητές των άλλων κοινοβουλευτικών ομάδων. Θα έλεγα 116 τροπολογίες συνολικά που μπορέσαμε να τις εντάξουμε με καλό τρόπο σε κάποιες συμβαστικές τροπολογίες που τώρα τις έχετε στα χέρια σας. Επίσης εξίσου και για τη γνωμοδότηση, γνωμοδοτήσει άλλων κοινοβουλευτικών επιτροπών που πολύ ενδιαφέρουσες πτυχές έχουν προσθέσει για αυτό το θέμα μας και κάποιες τροπολογίες επίσης που φαινόντουσαν αρχικά ότι δεν θα μπορούσαν να ενταχθούν με κάποιες ε, συζητήσεις που έγιναν και αποσαφηνήσεις καταφέραμε με ομοθυμία τις περισσότερες να τις εντάξουμε μέσα σε ένα ενιαίο πλαίσιο τροπολογιών, συμβαστικών τροπολογιών. Νομίζω ένα κέριο σημείο θεμελιώδους σημασίας για όλους τους κοιόδης εισηγητές ήταν η ελκυστικότητα τα θέλγητρα της επαγγελματικής κατάρτισης και η ποιότητα αυτής της κατάρτισης που πρέπει να διασφαλίζεται. Εδώ κάποια σημεία απαριθμήθηκαν μεταξύ αυτών και μια αλλαγή σε μια ιστερότερη χρονική στιγμή από μια επαγγελματική κατάρτιση σε μια εκπαίδευση πανεπιστημιακού επίπεδου που πρέπει και, αυτή να είναι, αυτό να είναι εφικτό ως βήμα. Αυτό ήταν ένα κέριο σημείο. Ένα άλλο κέριο σημείο το οποίο είχε απήχηση σε αρκετές ε, τέτοιες ε, σε τροπολογίες ήταν το, ο τομέας της, ε, δια, της περαιτέρω επιμόρφωσης, κάτι που αφορά πολλούς εργαζόμενους λόγω της δημογραφικής αλλαγής που παραμένουν περισσότερο στο χώρο εργασίας τους οι εργαζόμενοι. Πρέπει να καταφέρουμε περισσότεροι εργαζόμενοι να έχουν την προσφορά της επιμόρφωσης και της διαβίου εκπαίδευσης ε, και κατάρτισης. Να υπάρξει συνειδητοποίηση, μεγαλύτερη συνειδητοποίηση για αυτά τα θέματα, μεγαλύτερη ευαισθησία και να έχουμε και προσφορά επαγγελματική που θα προσφέρεται. Και έτσι στοχοθετημένα εντάξαμε ομάδες εργαζόμενους, μεταναστές, εθνοτικές μειονότητες, άτομα με αναπηρίες, αλλά επίσης και οικογένειες με μικρά παιδιά, με παιδιά που πάνε σχολείο ακόμα, διότι για αυτή την ομάδα δεν είναι τα πράγματα πάντα τόσο ευέλικτα ιδιαίτερα όταν έχουμε έναν ε, και μόνο εργαζόμενο. Πρέπει να ληφθεί υπόψη η επιμόρφωση, η κατάρτιση και στη στρατηγική για την Ευρώπη του 2020 και η συμμετοχή αυτής της ομάδας στοχοθετημένα να αυξηθεί. Και ήταν ένα σημείο πώς επιπρόσθετα νέες γυναίκες, κορίτσια, θα μπορέσουμε να τις προσελκύσουμε σε επαγγέλματα που κλασικά βρίσκονται υποπριτανεύων, υποδεσπόζοντα ρόλο των ανδρών. Και αυτό είναι ένα σημείο που στις τροπολογίες βρήκε απήχηση και στις συμβαστικές τροπολογίες. Ένα άλλο σημείο ήταν, πράγμα που ήταν σημαντικό και αυτό για μας, το σύνολο μέσω της διαδικασίας της Κοπενχάγης των μηχανισμών και αρχών και tools, εργαλείων ή μέσων που εκπονούνται όπως το πλαίσιο προσόντων και δεξιοτήτων όσον αφορά διπλώματα, πτυχία, ώστε αυτά το δυνατόν να μπορέσουν να υλοποιηθούν από τα κράτη-μέλη και να συνοδευτούν με τον καλύτερο τρόπο και να βελτιωθούν κιόλας όταν είναι αναγκαίο να υπάρξουν βελτιώσεις. Και για παράδειγμα ότι τα μη τυπικά, οι άτυπες, ε, ας το πω έτσι, δεξιότητες ή τα άτυπα προσόντα που έχουν αποκτηθεί από ένα εργαζόμενο να αναγνωρίζονται. Και αυτό είναι, ήταν ένα θέμα που μας απασχόλησε. Μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή ήταν η πτυχή της κινητικότητας για τους εργαζόμενους. Να υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης στο δυνατόν μεγαλύτερον αριθμό τέτοιων εργαζόμενων στην ευρωπαϊκή αγορά να βρουν απασχόληση με κινητικότητα. Αυτό ταιριάζει καλά και με την Youth on the Move. Οι νέοι κινητοποιούνται και βρίσκονται ε, ας το πω έτσι ε, καθοδόν και αυτό με θελούσια εθελοντική βάση να μπορέσει να προαχθεί και η πτυχή της ε, διασφάλισης κονδυλίων και εδώ με συμβιβασμούς ε, καταφέραμε να καταλήξουμε δεν θα υπάρχει αποκλειστική πρόσβαση κάποιων λίγων σε μια δεύτερη επιμόρφωση ή κατάρτιση, αλλά θα πρέπει το δυνατόν με ευρύτερη βάση για μεγαλύτερο αριθμό εργαζόμενων να υπάρξει χρηματοδότηση σε τέτοιου είδους προσφορές και δράσεις και μέσω και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου να υπάρχει δυνατότητα τα κράτη-μέλη να έχουν κίνητρα, να δράσουν και εκείνα για την υλοποίηση τέτοιων προτύπων, ώστε το δυνατόν περισσότεροι εργαζόμενοι, να έχουν πρόσβαση στην επιμόρφωση και κατάτηση. Ευχαριστώ. Merci. Ευχαριστώ. Και μετά ο κύριος Κοσλόφσκι, ο κύριος Σέλμερ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα παραδοσιακά να ευχαριστήσω την κυρία Χίρς για την εξαιρετική της εργασία. Θα ήθελα όμως να εκφράσω την απογοήτευσή μου, διότι ως κοιόδης από πλευράς συντηρητικών και ε, μεταρρυθμιστών δεν ε, έλαβα μέρος στις ε, τροπολογίες συμβιβασμού, στη διαδικασία τροπολογιών συμβιβασμού, διότι δεν μου έφτασε ποτέ η πρόσκληση. Και, εν πάση περιπτώσει, δεν θα ανταποκρίνονταν στη σκέψη της ομάδας. Θεωρούμε ότι η επαγγελματική κατάρτιση είναι ζωτική σημασίας και για να επικρίνω και τη δική μου χώρα, θα πρέπει να πω ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο τονίζουμε ιδιαίτερα την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία και όχι τόσο την επαγγελματική κατάρτιση όσο θα έπρεπε. Νομίζω ότι η κυβέρνηση θα διορθώσει την κατάσταση. Το ζήτημα είναι ποια είναι η προστιθέμενη αξία που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα κράτη-μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις οι οποίες είναι κατάλληλες ως προς ανάγκες τους, την πείρα, τον πολιτισμό τους, το εκπαιδευτικό σύστημα και ούτω καθεξής. Επίσης, αυτή, αυτή την έκθεση την είδαμε σαν ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο όπου βάζουμε πολλά στολίδια, μιλάμε για το γεγονό ότι δεν θα πρέπει να γίνονται φιλετικέ διακρίσεις, εθνοτικέ διακρίσεις και ούτω Όλα αυτά συσσωρεύονται και δεν οδηγούν σε τίποτα. Θα υπερψηφίσουμε βεβαίως, αλλά είμαστε απογοητευμένοι για την όλη έκβαση της υπόθεσης και το πώς την χειρίστηκε η συγγήτρια Κοσλόφσκη και μετά η κυρία Λάμπερτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστώ τον κυρία Χίρς για τις προσπάθειες που κατέβαλε στην κατάρτιση αυτής της έκθεσης και θα ήθελα για μια ακόμα φορά να πω ότι η έκθεση αυτή είναι ιδιαίτερα συνεκτική. Πολλά στοιχεία υπάρχουν για την επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση και θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την αγαστή συνεργασία. Εργαστήκαμε από κοινού για τη σύνταξη αυτού του εγγράφου και μαζί με άλλους σκιώδεις φτάσαμε σε τροπολογία συμβιβασμού που πρότεινε η συγγήτρια. Φτάσαμε σε συνένεση και έχουμε 13 τροπολογίες συμβιβασμού που δέχομαι και θα ήθελα να ενθαρρύνω όλους να υπερψηφίσουν αυτές τις τροπολογίες συμβιβασμού. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένες τροπολογίες που δεν έχουν ενταχθεί στο συμβιβασμό αυτό, στο συμβιβασμού αυτούς. Και έχω προτείνει προφορικές τροπολογίες. Στην 78 προτείνεται να υπάρχει η λέξη encourage και όχι call, δηλαδή ενθαρρύνει και όχι καλή. Στην 76 Πιστεύω ότι οι βιώσιμες εργασίες, η βιώσιμη εργασία αντικατοπτρίζει καλύτερα το όλο πλαίσιο. Και μαζί με έναν συνάδελφο έχουμε υποβάλει προφορικές δικέ του τροπολογίες για να μην μιλάμε για calls αλλά για encourages στην 41 και να μιλήσουμε στην 106 για καλύτερη εποπτεία. Επίσης, θα ήθελα να λάβετε υπόψη και αυτές τις ε, προφορικές μαζί με την έκθεση. Η κυρία Λάμπερτ και δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχουν και άλλοι ομιλητές. Λάμπερτ και μετά θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος δεν μπόρεσε να παρευρεθεί εδώ σκιώδης και θα ήθελα να πω ότι η συγγήτρια ε, θα τύχει της υποστήριξής μας μαζί με τις τροπολογίες συμβιβασμού. Εξαιρετική είναι πράγματι η εργασία της. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, το προγράμματος Λεωνάρντο Νταβίντσι και ούτω καθεξής. Ως προς την τροπολογία 21 παράγραφος 1, θέλαμε, θελήσαμε να αναφερθούμε σε ορισμένες χρηστές πρακτικές ε, της Δανίας, Γερμανίας και της Αυστρίας σε σχέση με την επαγγελματική κατάρτιση ε, σε σχέση με άλλα κράτη-μέλη που δεν ε, το επιτελούν αυτό. Θα έπρεπε λοιπόν να εκθιάσουμε αυτές τις χώρες, αλλά δυστυχώς αυτός ο εκθιασμός δεν εντάχθηκε στις τροπολογίες συμβασμού. Δεν υπάρχουν άλλοι εγγεγραμμένοι. Ξαναδίνω το λόγο στην κυρία Χίρς. Ähm, Ευχαριστώ πολύ. Για να στραφώ αμέσως στα θέματα αυτά που τέθηκαν. Τροπολογία 21. Αυτό με διάφορες, στις διάφορες χώρες, όπου δηλαδή επαγγελματική κατάρτιση σε ένα διοικό, σε δύο σκέλη ως σύστημα υιοθετείται. Είχαμε κάποιες συζητήσεις που έγιναν μεταξύ των σκιωδών εισηγητών και το πρόβλημα ήταν ότι υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη που, ας το πω έτσι, έχουν ένα παρόμοιο ή συγκρίσιμο σύστημα, είχαν ένα τέτοιο συγκρίσιμο σύστημα. Αν μπορούμε δηλαδή να απαριθμίσουμε όλα αυτά τα κράτη, ποια μπορούν να απαριθμηθούν, ποια όχι, και γι' αυτό στο τέλος συμφωνήσαμε και είπαμε, εντάξει, τα άτομα εκείνα που αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα γνωρίζουν ποια είναι τα κράτη-μέλη που έχουν διοικό τέτοιο σύστημα κατάρτισης σε δύο σκέλη. Γι' αυτό είναι δύσκολο τώρα να απαριθμηθούν εδώ ένα προς ένα σε ποια ισχύει κάτι και σε ποια όχι. Οι αρμόδιοι γνωρίζουν. Ένα άλλο θέμα ήταν οι προφορικές τροπολογίες, οι τροποποιήσεις. Καθότι είδα θα μπορούσα όλες να τις υποστηρίξω. Είναι πολύ καλές συμπληρώσεις οι τροποποιήσεις προτάσεων τροπολογιών που δίνουν κάτι επιπρόσθετο ακόμα ως αξία και δημιουργούν και κάποια διευκρίνηση, διευκρινίζουν περισσότερο τα πράγματα. Λυπούμε, ας το πω έτσι, αν δεν κατάφερε η πρόσκληση να φτάσει στα χέρια σας να συμμετάσχετε. Από την άλλη πλευρά επανειλημμένα έχουμε ανταλλάξει απόψεις στην Κοινοβουλευτική μα Επιτροπή και είδαμε τέτοιε τροπολογίε. Λυπούμε για το ότι δεν καταφέρατε να συμμετάσχετε, αλλά νομίζω συμφωνούμε όλοι ότι η επαγγελματική κατάρτιση έχει υψηλή προτεραιότητα και ελπίζω λοιπόν ότι παρόλα αυτά θα υπερψηφίσετε την έκθεση στο τέλος. Κατά τα άλλα και πάλι ευχαριστώ θερμά, διότι για αυτή τη χρονική στιγμή οι πτυχές ε, της ε, ανεργίας των νέων είναι ιδιαίτερα σημαντικές, ιδιαίτερα για την επαγγελματική κατάρτιση. Να προαχθεί η πτυχή αυτών των νέων ανέργων. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Θα ψηφίσουμε την έκθεσή σας Αύριο. Και έτσι φτάνουμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη, στο σημείο 7 δηλαδή. Εδώ γνωμοδοτούμε για την Επιτροπή Πολιτισμού. Πρόκειται για την πρωτοβουλία νεολαία σε κίνηση. Το λόγο έχει η συγγήτριά μα για να μας παρουσιάσει και τι 18 τροπολογίες. Παρακαλώ κυρία Στάινβρου και έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Λοιπόν, ο αριθμό των τροπολογιών 186 δείχνει ο αριθμός ότι υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτή την έκθεση και πραγματικά πρέπει να πω χάρηκα ότι σχεδόν όλοι στην ίδια κατεύθυνση στόχευαν και η συνεργασία με τους συναδέλφους διευκολύνθηκε και με τους ε, εισηγητές κατά τα άλλα. Ήταν εξαιρετικά καλή αυτή η συνεργασία και σε αμοιβαία εμπιστοσύνη ως βάση. Όλοι θέλουμε την κατάσταση των νέων να την βελτιώσουμε και θέλουμε όλοι πώς να το πω, το μέλλον των νέων να είναι καλύτερο, να βελτιωθεί και αυτό. Πέρα από ιδεολογικούς φραγμούς και όρια, διακομματικά καταλήξαμε σε καλούς συμβιβασμούς που τα πιο σημαντικά σημεία νομίζω τα καλύπτουν που είναι η μετάβαση από το σχολείο στην επαγγελματική ζωή για τους νέους, υποστήριξη στην επιλογή επαγγέλματος αλλά και χωρίς μεγάλες μεταβατικές ή ενδιάμεσες περιόδους ή καθυστερήσεις να γίνεται αυτή η μετάβαση. Δεν πρέπει να γίνεται υπό, πιο επιδεινωμένες συνθήκες και όρους η έναρξη επαγγελματικής ζωής για τους νέους από σε σχέση με άλλους. Το χρωστάμε στους νέους αυτό και ασχοληθήκαμε και με την πρακτική εξάσκηση των νέων στη μαθητεία που είναι πολύ χρήσιμη περίοδος για την εκμάθηση επαγγελμάτων Χρειάζονται όμως ένα ποιοτικό πλαίσιο και κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές. Το θέμα της κινητικότητα σήμερα και αυτό προαναφέρθηκε. Χρειάζεται κινητικότητα, αλλά έχει τα όρια της και η κινητικότητα. Πρέπει εθελοντικά να μπορεί να λειτουργεί με εθελούσιο πλαίσιο, εθελοντικό πλαίσιο. Όσον αφορά τα όσα είχαμε συζητήσει, είχαν εμπλακεί όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Θα ήθελα σίγουρα στο ένα ή άλλο σημείο να είχαμε πιο ισχυρές, πιο αυστηρέ διατυπώσεις όταν πρόκειται για τη μαθητεία των νέων και την περίοδο άσκησης, ώστε να αποφύγουμε διακριτική αρνητική μεταχείριση νέων. Αλλά συνολικά στο τέλος τέλος νομίζω καταλήξαμε σε μια καλή γνωμοδότηση. Σας ευχαριστώ. Κύριος Σέλμερ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευθύς εξ αρχής θέλω να σας πω ότι όλοι θα θέλαμε να βοηθήσουμε τους νέους να περάσουν από το σχολείο στην επαγγελματική ζωή, όλοι θα θέλαμε να τους βοηθήσουμε να έχουν καλή δουλειά, αλλά και έτσι καλώ με εμπιστοσύνη μπορώ να σας πω ότι κανένας δεν θα σηκωθεί εδώ πέρα να πει ότι όχι δεν το θέλουμε. Εννοείται, όλοι το θέλουμε. Οπότε και πάλι ε, το ζήτημα δεν είναι το κατά πόσο συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε, αλλά το κατά πόσο η συγκεκριμένη γνωμοδότηση μα βοηθάει να πετύχουμε και το στόχο. Και εγώ δεν πιστεύω ότι το κάνει. Το είπα και στην προηγούμενη έκθεση. Δεν βλέπω ποια είναι η προστιθέμενη αξία εδώ με αυτή τη γνωμοδότηση. Θέτουμε αυθαίρετους στόχους που τι είναι, μια ασπιρίνη για μια σοβαρή αρρώστια. Δεν νομίζω λοιπόν ότι στην πράξη προσφέρουμε καμία σοβαρή μέθοδο για να πετύχουμε τους στόχους. Την ίδια παρατήρηση έχω και εδώ λοιπόν όπως και με την προηγούμενη έκθεση. Τα συστήματα που θέλουμε να εφαρμόσουμε ή που εφαρμόζουμε μάλλον θα πρέπει να προσαρμόζονται στην κατάσταση που επικρατεί στην κάθε περίπτωση, είτε πρόκειται σε μια χώρα, σε μια περιφέρεια ή για τον καθένα χωριστά και όχι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έπειτα, η γνωμοδότηση δεν πρόκειται να προσφέρει τίποτα παραπάνω είναι απλώς μια πολιτική χειρονομία. Δηλαδή ότι η Επιτροπή μας να προσπαθεί να δείξει ότι κάτι έχει να πει, ότι τους νοιάζεται τους νέους. Αλλά δεν προσφέρει κανένα αποτέλεσμα. Γι' αυτό και η ομάδα μου θα καταψηφίσει αυτή την γνωμοδότηση. Πρόεδρο, η κυρία... Όχι, ο κύριο Μπατ πρώτα και μετά η κυρία Ντελή. Σα ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω στην εισηγήτριά μου την αναγνώριση και εκτίμηση για αυτή την έκθεση. Ήταν καλή συνεργασία μας και ευθύ εξ αρχής από πλευράς της εισηγήτριας στόχευε σε συμβιβασμούς στη δουλειά αυτή όπως προαναφέρθηκε ένα εγχείρημα το οποίο δεν ήταν εύκολο, δεδομένων διαφορετικών απόψεων που επικρατούν στις διαφορετικές ομάδες. Όσον αφορά τα προβλήματα, τα ίδια, τα θέματα, συμφωνούμε όσον αφορά την κατάσταση των νέων στην Ευρώπη, που είναι δραματική η κατάσταση των νέων στην Ευρώπη σήμερα και από όλε τι πλευρέ πρέπει να γίνουν προσπάθειε ώστε να βελτιωθεί η κατάστασή του. Επιμέρου σημεία παριθμήθηκαν από την εισηγήτρια. Θα έλεγα πιο, τα πιο σημαντικά σημεία είναι ο καλύτερο συντονισμό μεταξύ των διαφορετικών συστημάτων εκπαίδευση και τη αγορά εργασία. Αναφέραμε και την βελτίωση τη κινητικότητα των νέων. Δηλαδή διασυνοριακά να μπορούν να κινητοποιούνται οι φοιτητέ και οι εργαζόμενοι όμω έχουν και αυτοί εξίσου μεγάλη σημασία να διακινούνται διασυνοριακά. Έχουμε όμως και κάποια προβλήματα σε σχέση με τα κράτη-μέλη. Είναι κατά τούτο σημαντικό λοιπόν από πλευράς μας να επισημαίνουμε τα προβλήματα αυτά και για να επιληθούν. Τα υφιστάμενα προγράμματα για τους νέους που πρέπει να υποστηριχθούν και αυτά είναι σημαντικά. Αναγνώριση ελάχιστων προδιαγραφών, κοινωνικών δικαιωμάτων. Αυτά είναι πολύ σημαντικά και θέλω να τονιστούν. Θέλω να τονίσω ότι αυτή η έκθεση μόνη της δεν θα επιλύσει τα προβλήματα, αλλά δίνει ενδιαφέρουσε προσεγγίσεις για την επίλυσή τους. Καλούνται τα κράτη-μέλη να συντάξουν και να καταρτήσουν εθνικές στρατηγικές για την κατάρτιση και εκπαίδευση των νέων σε υψηλής ποιότητα θέσεις απασχόλησης. Ελπίζω ότι αυτή η έκθεση θα υπερψηφιστεί με μεγάλη πλειοψηφία. Ευχαριστώ. Ε, η κυρία Ντελή και μετά η κυρία Λίν. Συγχαρητήρια προς την εισηγήτρια και από μένα. Με τη συνάδελφο Ζουμέν θέσαμε και υποβάλαμε διάφορες τροπολογίες με τις οποίες συμφώνησε και η ε, διακοινοβουλευτική ομάδα για την νεότητα. Τώρα οι τροπολογίες μας συμπεριλαμβάνονται σχεδόν όλες ε, στο συμβασμό. Άρα είμαστε ικανοποιημένοι. Εκτός, εκτός από το ότι υπάρχει ένα συμβασμός που μας προβληματίζει. Πρόκειται για τον συμβασμό ΒΑ. Στη δική μας τροπολογία λέγαμε αυτό το οποίο έλεγε και η έκθεση Φιγκερέιδο, ότι δηλαδή απλά οι χώρες μέλη πρέπει να καταργήσουν κάθε διάκριση βάσει της ηλικία, ιδιαίτερα όσον αφορά την πρόσβαση στον ελάχιστο μισθό και την κοινωνική προστασία. Δυστυχώς σήμερα στον συμβασμό αυτό ΒΑ δεν υπάρχει αυτό το σημείο. Αν δεν υπάρχει αυτή η φράση, ο συμβασμός δεν έχει νόημα και γι' αυτό ζητάω αύριο οι συνάδελφοι να υπερψηφίσουν την τροπολογία μας αριθμό 43. Η κυρία Λίν και μετά η κυρία Χαρκίν. Θα ήθελα μία αναθεωρημένη έκδοση των συμβασμών και γι' αυτό θα ζητήσω συγγνώμη αν, έχω, αν αναφέρω λάθος αριθμούς. Ορισμένες ε, τροπολογίες έχουν συμπεριληφθεί στις τροπολογίες συμβιβασμού. Δεν μιλήσαμε για αυτές η ΑΒ μιλά για μέτρα λιτότητας και για περικοπές στην εκπαίδευση. Δεν ξέρω κατά πόσο η αρρύθμιση παραμένει η ίδια, αλλά αυτό παραμένει αρμοδιότητα των κρατών μελών. Άρα από αυτή της πλευράς μας ενδιαφέρει το επιχείρημα επικουρικότητας. Ο Συνδεσμός Β τονίζει τις συμβάσεις κατάρτισης και μιλάμε για πολύ περισμένο πλαίσιο, μάλλον είναι πολύ γενικό και δεν ξέρουμε κατά πόσο ε, μιλάμε για συμβάσεις απασχόλησης που παραμένουν αρμοδιότητα των κρατών μελών. Το F δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει υποστήριξη του οικογενειακού ρόλου, του ρόλου της οικογένειας, αλλά είναι κάτι το οποίο συζητήσαμε πολλές φορές. Γνωρίζω ότι πολλοί λένε ότι θα πρέπει να εντάξουμε τα νοικοκυριά και όχι την οικογένεια, γιατί υπάρχουν μερικοί που αντιτίθενται στη χρήση της λέξης οικογένεια. Ίσως θα ήταν καλύτερα να μιλάμε για νοικοκυριά αντί για οι οικογένειες. Για το J, για ε, τα, τις ελάχιστες προδιαγραφές για την εσωτερική εργασία, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα πρέπει να επαφίεται στα κράτη-μέλη. Ζητώ συγγνώμη αν η αρρύθμιση δεν είναι η σωστή. Και υπάρχουν και ορισμένες άλλες τροπολογίες συμβασμού που δεν με βρίσκουν σύμφωνοι, αλλά θα τις δούμε πριν από αύριο το πρωί. και μετά ο κύριος Τόμας Μαν. Άρκιν, Χάρκιν. Όπως ξέρετε, ε, η Σκιώδης ε, μου ζήτησε να πω ότι είναι ε, ικανοποιημένη με τις τροπολογίες συμβασμού και δεν έχει ουσιώδη σχόλια επί της έκθεσης. Το μόνο που θα ήθελα να αναφερθώ σε σχέση με αυτά που είπε η Λίζ Μερικοί δεν θέλουν να γίνει χρήση της λέξης οικογένεια. Εγώ δεν το βλέπω υπό αυτή την οπτική γωνία, γιατί όλοι ανήκουμε σε οικογένειες διαφορετικού τύπου ε, από τη στιγμή που κανείς δεν είναι περιοριστικός για το πώς ορίζει την οικογένεια. Δεν βλέπω γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε αυτό τον όρο που είναι ένας όρος κοινή χρήση και που γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά τι σημαίνει και τι διαστάσεις μπορεί να λάβει. Ο κύριος Τόμας Μαν και μετά κυρία Χίρς. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ήθελα να πω στην Γιούτα Στάινμπορκ επειδή η έκθεση ήταν τόσο καλή δεν είχα καμιά ευκαιρία να θέσω τροπολογίες. Διότι πιστεύω ότι τα θέματα καλύπτονται και διατυπώνονται σωστά ιδιαίτερα για τον τρόπο πώς θα καταφέρουμε σε στοχοθετημένες ομάδες να καταλήξουμε καλύτερα. Πολύ σωστά έχουν διατυπωθεί. Αν δει κανείς αυτές τις τροπολογίες που οδήγησαν σε συμβαστικές τροπολογίες έχουμε μια καλή βάση. Το τι γίνεται με το ΕΛΚΑ μπορούμε πραγματικά να πούμε, μπορούμε να υποστηρίξουμε την έκθεση που έχουμε μπροστά μας. Και αν, μια και έχουμε και τους δύο από τη, εδώ κοντά την Μία και τον Ρότζερ. Ο Ρότζερ είπε με επικριτικό πνεύμα ποια είναι η πρόσθετη αξία που απορρέει. Φυσικά τα κράτη-μέλη είναι αρμόδια για την επαγγελματική κατάρτιση, την επιμόρφωση. Δεν χρειάζεται εδώ να αυτό, δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Αυτό που προσφέρουμε όμω, Ρότζερ είναι η δυνατότητα να βοηθήσουμε ω αρρωγή ή να κάνουμε κάποια πράγματα ω Ευρωπαϊκή Ένωση για την κινητικότητα. Ένα σημαντικό θέμα αυτό. Είναι αναγκαίο να πούμε τι μπορούμε από τα άλλα κράτη-μέλη να αντιγράψουμε, να υιοθετήσουμε και τι πρέπει να δούμε με ιδιαίτερη προσοχή για τα συστήματα που έχουμε στα κράτη-μέλη για την κατάρτιση και ε, με επιμόρφωση. Και υπάρχει ένας συμβιβασμός με το με θέματα τα οποία εντάσσονται για το πλαίσιο της επαγγελματικής αναγνώρισης. Και εδώ πάλι ένα πλαίσιο δημιουργούμε. Θέλουμε μελλοντικά στην Ευρώπη τα πτυχία ή τα προσόντα να καθορίζονται με αυτόν τον τρόπο για να μπορούμε να ξεκινήσουμε κάτι από κοινού. Αν έχουμε κοινού ορισμούς τότε δεν επιβάλλονται από την Ευρώπη, δεν επιβάλλονται εκ των άνω προς τα κάτω, θέλουμε να καταλήξουμε σε μια κατάσταση win-win, να κερδίζουμε όλοι, να έχουμε έναν ορισμό, να ξέρουμε ποιες προϋποθέσεις ισχύουν, ώστε να μπορέσει μια επαγγελματική, ας το πω έτσι, σταδιοδρομία να έχει αναγνωρισμένο ε, πτυχίο ή ε, δίπλωμα. Έτσι μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα ενιαίο πλαίσιο. Αν το καταφέρουμε έχουμε added value, πρόσθετη αξία, χωρίς να αναμειγνιόμαστε στα θέματα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών. Τι κάνουμε. Έχουμε συνέδρια, έχουμε έγγραφα στις διάφορες ε, γλώσσες μας, να κατανοούμε περί τίνος πρόκειται και να στοχεύουμε προς την ορθή κατεύθυνση. Αυτή είναι η σωστή βάση. Συγχαρητήρια Γιούτα, από πλευρά μου. Έχουμε μια καλή βάση για να εγκρίνουμε. Εμείς ως ΕΛΚΑ θα, νομίζω μπορούμε να το πούμε, έχουμε σαφή θέση για την υπερψήφιση. Ευχαριστώ. Ε, ε, um, Σας ευχαριστώ και από δικής μου πλευράς. Ευχαριστώ και συγχαρητήρια θερμά στην εισηγήτρια και ευχαριστούμε θερμά για την πολύ καλή συνεργασία, για τις πολλές ε, τροπολογίες ε, που είναι πάντα μια πρόκληση θα έλεγα πολύ καλά τα καταφέρατε και βλέπουμε και με τους συμβιβασμούς ότι τις πολλές αυτές τροπολογίες τις καλύψατε και ιδιαίτερα για την προς την ορθή κατεύθυνση. Κατά τούτο πολλά σημαντικά σημεία αναφέρονται, ιδιαίτερα σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση για την επαγγελματική κατάρτιση. Χαίρομαι που εδώ καταφέρνουμε προς την ίδια κατεύθυνση να πορευθούμε. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε αυτά τα θεματικά πλέγματα να το κάνουμε. Παρόλα αυτά όμως και από σκιωδών εισηγητών στη συνάντηση είπαμε ότι σε ένα συμβιβασμό δυστυχώς δεν μπορούμε να τον υποστηρίξουμε. Το, το G, το G πρόκειται για ελάχιστες προδιαγραφές ε, για, ε, που θα μπορούσαμε να, τους, να τις υποστηρίξουμε αλλά αναφέρεται εδώ επιπλέον και αυτό είναι η πρόκληση ότι πάντα λέει πρέπει να καταβάλλεται μισθός σε αυτούς τους ασκούμενους. Πράγμα το οποίο έχει νόημα να γίνεται, αλλά υποχρέωση όμως αν εισαχθεί από την άλλη πλευρά θα οδηγήσει ενδιαφέρουσες θέσεις μαθητείας να μην μπορούν να καλύπτονται με τέτοιους μισθούς και έτσι να μην μπορούν να λειτουργήσουν και να χάνονται αυτές οι θέσεις μαθητείας και άσκησης. Όταν λέμε πάντα πρέπει να καταβάλλεται μισθό στον ασκούμενο κτλ. Γι' αυτό, γι αυτό το συμβιβασμό π, π διορθώνω, θα απόσχουμε για το π, το π. Και κατά τα άλλα έχουμε και την πρόκληση για τα κράτη-μέλη. Πολλά από αυτά τα σημεία να μπορέσουν να, να υλοποιηθούν σωστά. Πρόκειται και για πεδία που δεν έχουμε αρμοδιότητα στο ευρωπαϊκό επίπεδο εμείς. Είναι μόνο προτάσεις που υποβάλλουμε για να κινητοποιηθούν τα πράγματα στα κράτη-μέλη. Είναι όμως σημαντικό να το κάνουμε αυτό για να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα προς τα κράτη-μέλη και στο τέλος τέλος να έχουμε μια ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και το θέμα των, της ανεργίας των νέων είναι ευρωπαϊκό θέμα. Πρέπει όλους σε ευρωπαϊκό επίπεδο να απασχολήσει, να αναζητηθούν λύσεις στα προβλήματα σε μια κοινή βάση. Έτσι να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε. Η συγκεντριά μας τώρα, κύριε Στάνμπρου, και έχει το λόγο. Είναι πολύ σημαντική η θέση μας, ακόμα και αν γνωμοδοτούμε απλώς. Και αυτό γιατί συμμετέχουμε με την Επιτροπή Πολιτισμού. Έχετε το λόγο κύριε Συγήτρια. Ναι. Και πάλι ευχαριστώ όλες τις συναδέλφους και τους συναδέλφους. Έχω κάποιες παρατηρήσεις να κάνω. Η πρώτη προς τον κύριο Χέρμερ. Παρότι... Και ο Τόμας Μαν και η Νάντια Χίρς το ανέφεραν επίσης. Θα ήθελα, αν έχει κάποιος κάποιες εξειδικεύσεις, να δω κάποιες εξειδικευμένες τροπολογίες, ώστε η συνεργασία στις διαπραγματεύσεις να διευκολύνεται. Χρειάζομαι αυτές τις ιδέες να υποβάλλονται. Το να ασκεί κανείς επικρίσεις είναι μία υπόθεση, αλλά για να πηγαίνουν καλύτερα τα πράγματα πρέπει ενεργά να συμμετέχει κανείς. Ευχαριστώ όσους ενεργά συμμετείχαν. Είναι μια γνωμοδότηση στην οποία Έγινε πολλή δουλειά από πλευράς μας. Προσπαθώ τα θέματα που εκκρεμούν να απαντήσω. Για την κυρία Ντέλη αναφέρθηκε για το θέμα του συμβιβασμού ε, για την διακριτική μεταχείριση σε σχέση με την ηλικία η ανάγκη συμβιβασμού υπάρχει εδώ, αλλά η στοχοθέτηση νομίζω, η κατεύθυνση παρέμεινε, ακόμα και αν στη διατύπωση είμαστε πιο αποδυναμωμένοι, ας το πω έτσι, σε αυτή την πρόθεση. Είχα άλλη αρρύθμιση εγώ από πλευράς μου, γι' αυτό δεν κατάφερα να παρακολουθήσω την παρέμβασή σας πιο εξειδικευμένα. Μπορούμε διμερώς να το συζητήσουμε στη συνέχεια. Νομίζω σε πολλά σημεία οι σκιώδεις εισηγητές ε, εξοικειωθήκαμε και τα εξειδικεύσαμε. Όσον αφορά το συμβιβασμό Π, το Π, ήταν πρόθεση από πλευράς εισηγήτριας και από πλευράς και οδών εισηγητών θέλαμε να αποφύγουμε νέοι για πολλά χρόνια να δυσχεραίνονται να βρουν απασχόληση στο επάγγελμά τους και μάλιστα έχοντας πολυετή και χωρίς μισθό ε, έτη μαθητείας και άσκησης. Θέλαμε να πούμε δεν μπορεί αυτό να είναι ο κανόνας άμυστα να απασχολούνται και να ε, εξασκούνται. Γι' αυτό καταθέσαμε αυτήν την τροπολογία. Κατά τα άλλα πιστεύω ότι η Επιτροπή Πολιτισμού με μεγάλη πλειοψηφία υποστηρίζει αυτή τη γνωμοδότηση, διότι αυτά τα θέματα είναι θεμελιώδους σημασίας για το, το νέο, τους νέους και το μέλλον τους. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε. Θα ψηφίσουμε λοιπόν τη γνωμοδότηση αυτή αύριο. Και έτσι φτάνουμε στο σημείο 8 στην ημερήσια διάταξη. Πρόκειται για γνωμοδότησή μας για την Ένωση Καινοτομίας. Γνωμοδοτούμε λοιπόν για την Επιτροπή Ήτρε εμείς εδώ. Η συγκίτριά μας είναι η κυρία Σάρι Εσάγια, στην οποία και δίνω το λόγο ευθύς αμέσως για να εξετάσουμε τις τροπολογίες μαζί της. Παρακαλώ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τους συναδέλφους για τις επικοδομητικές ε, τροπολογίες. Το πνεύμα αυτό αυτής της έκθεσης και των τροπολογιών σχετίζεται στο γεγονός ότι οι καινοτομίες θα πρέπει να θεωρούνται κοινωνικού χαρακτήρα καθώς και ως προς τις, στον τομέα των υπηρεσιών για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και τις δημογραφικές αλλαγές. Υπάρχουν πέντε τροπολογίες συμβιβασμού που έχουν γίνει αποδεκτές από αυτούς που τις έχουν, και από αυτούς που τις έχουν υποβάλει και από τους υπόλοιπους. Οι περισσότερες έχουν γίνει αποδεκτές από το ΕΛΚ. Υπάρχει μία τοπολογία, η 20, που είναι πολύ σημαντική, δηλαδή να προωθήσουμε την ισότητα των δύο φύλων στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης και της τεχνολογίας, αλλά στην 20 ζητούμε ε, γενικές κατευθυντήριες γραμμές, ειδικές κατευθυντήριες γραμμές, αλλά εντάσσονται στην επικουρικότητα οι κατευθυντήριες γραμμές και θα πρέπει να αποφασιστούν από τα κράτη-μέλη. Δηλαδή να αποφασίσουν τα κράτη-μέλη και να δουν κατά πόσο θα χρησιμοποιήσουν τις κατευθυντήριες γραμμές της. Στην 21 μιλάμε για πράσινη εργασία και θα θυμόσαστε ότι στην Επιτροπή είπαμε ότι σύμφωνα με τον ορισμό του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας ε, θα ήταν βιώσιμες, ε, πιο βιώσιμες οι εργασίες αν έχουν ε, ένα πιο βιώσιμο βάθρο. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να μιλήσουμε για πράσινη εργασία, πράσινες θέσεις εργασίας. Δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχουν πράσινες, κόκκινες, γκρίζες. Σε πάση περιπτώσει δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να μιλάμε για πράσινες θέσει εργασία, αλλά βιώσιμες θέσει εργασία. Αυτή είναι η ουσία. Στι 37, στις 37 και 38 δεν ε, βρήκαμε μια κοινή ε, σύνταξη με μια σκιώδη. Γι' αυτό θα ψηφιστούν ξεχωριστά με την κυρία Σρέντερ. Ε, διαφορετικά οι υπόλοιπε μπορούν να γίνουν αποδεκτές και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξή σας αυτή της ε, γνωμοδότησης. Κυρία Στρέλα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ την εισηγήτρια για την εξαιρετική αυτή εργασία και για το γεγονός ότι προσπάθησε να διευρύνει το πλαίσιο εργασίας και γι' αυτό ακριβώς έγιναν αποδεκτές και οι προτάσεις των άλλων ομάδων. Γι' αυτό θα υποστηρίξουμε, η ομάδα μου θα υποστηρίξει τις έξι τροπολογίες συμβασμού στις οποίες προαναφερθήκατε. Σε σχέση με τις δικές μας προτάσεις ε, τροπολογιών, έχουμε υποβάλει οκτώ προτάσεις, η 7 με τις 7 συμφώνησε η εισηγήτρια εκτός από την 20 στην οποία αναφερθήκατε. Και είπατε ότι θα πρέπει να, είναι, να φορά ευθύνε των κρατών μελών. Ε, δηλαδή κατά πόσο θα υπάρχουν αυτές οι ειδικέ κατευθυντηρίες γραμμές. Αλλά αυτή η πρόταση έχει λόγο ύπαρξης όπως ξέρετε το θέμα της ισότητας των δύο φύλων είναι ένα θέμα ευαισθητοποίησης και χρειάζεται καλύτερη κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού. Γι' αυτό υποβάλαμε αυτή την πρόταση τροπολογίας. Θεωρούμε ότι η γνωμοδότηση αυτή είναι σημαντική, είναι εξισορροπημένη και λαμβάνει υπόψη την Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020 και υπ' αυτή την ε, έννοια και στα πλαίσια της παρούσης ε, κρίσης έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Και γι' αυτό ακριβώς θα υποστηρίξουμε αυτή την τροπολογία και την έκθεση γενικότερα. Κυρία Στρέτερ. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, αρκετά έχουμε, εκτενώς αρκετά συζητήσαμε με την εισηγήτρια και διαπραγματευθήκαμε για τις διαφορετικές τροπολογίες. Υπήρξαν διαφορετικές προοπτικές όσον αφορά το περιεχόμενο αυτής της ίδιας της έκθεσης για τις συζητήσεις. Και είναι σαφές ότι εγώ πιστεύω ότι η καινοτομία είναι ένα σημαντικό πεδίο, ιδιαίτερα όσον αφορά την αηφορία στην ανάπτυξη. Και έχουμε και πολλές εκθέσεις όπου προσπαθήσαμε η κοινωνική διάσταση πραγματικά να αναγνωριστεί και να ε, προωθηθεί. Και έχουμε και τροπολογίες που κατέθεσα, τροπολογίες που έχουν εγκριθεί ήδη και στο παρελθόν εδώ από πλευράς μας. Και υπήρξε ένα επίμαχο θέμα, το γνωρίζουμε αυτό. Και παραμένει και εκκρεμεί αυτό το θέμα. Όχι με όλους του ΕΛΚ, αλλά φυσικά σε σχέση με την εισηγήτρια, το γνωρίζουμε αυτό. Ταυτόχρονα όμως η εισηγήτρια την καινοτομία την εισήγαγε και σε που θα έλεγα δύσκολο είναι να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Είναι τομεί που δεν, τα, δεν τους έχουμε, όπως ο τομέας των κοινωνικών λέει υπηρεσιών. Ποιος είναι ο στόχος της καινοτομία εδώ, δεν μπορώ να το κατανοήσω. Πολλά μπορώ να κατανοήσω, επειδή γνωρίζω τα παραδείγματα από την Φινλανδία και τις φινλανδικές ε, ιδιομορφίες. Αλλά τώρα Κάτι το οποίο δεν έγινε δεκτό ως ε, το υπόδειγμα, το πρότυπο της ε, Φινλανδίας από την εισηγήτρια. Αλλά συνολικά μας λέει, τι για άλλα κράτη-μέλη λέει πρέπει να ισχύει. Και το βρίσκω προβληματικό αυτό και το λέω αυτό ξεκάθαρα σε αυτό το σημείο, είναι ένα επίμαχο σημείο που παραμένει. Δεν θέλω κάποια σημεία να καλύπτονται από καινοτομία χωρίς να υπάρχει εξειδίκευση για αυτή την καινοτομία και τις δράσεις. Ιδιαίτερα όσον αφορά εξαρτημένους από ναρκωτικά και άλλα τέτοια άτομα. Δεν μου είναι αδιάφορο τι θα γίνει με, αυτά τα, με αυτές τις πρωτοβουλίες θέλω ο κοινωνικός τομέας να διαδραματίζει κέριο ρόλο. Και μια και η διατύπωση είναι κάτι που ταιριάζει για όλα τα κράτη, πρέπει να ταιριάζει σε όλα τα κράτη-μέλη και όχι μόνο σε ένα. Αλλά θα ρυθμιστεί αυτό το θέμα το επίμαχο αύριο ψηφίζοντας και θα δούμε ποια θα είναι η έκβαση. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, θα ήθελα να πω υποστηρίζω το αίτημα των σοσιαλδημοκρατών ότι φυσικά πρέπει να πούμε ότι η αναγνώριση της συνιστώσας του φίλου είναι κάτι που πρέπει να αναγνωριστεί και να ενταχθεί σε αυτές τις πολιτικές. Ε, Μάνα Μαρκίν. Η κυρία Χάρκιν. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ την εισηγήτρια για τη δουλειά της. Συμφωνούμε να έχουμε βιώσιμη εργασία για πράσινες θέσεις απασχόλησης. Και συμφωνούμε επίση ότι η καινοτομία πρέπει να έχει να κάνει και με την απασχολησιμότητα. Καλό είναι που υπάρχουν πρακτικές προτάσεις. Στηρίζουμε επίσης να αρθούν τα εμπόδια που μπαίνουν για την ε, κινητικότητα των ερευνητών. Πρόεδρος, θέλει κανείς άλλο το λόγο? Όχι από ό,τι βλέπω. Ε, Θέλετε να πάρετε εσείς τώρα το λόγο, κύριε Σιγήτρια. Απλώς να πω ότι έχουμε να κάνουμε με έναν τάχιστα γυράσκοντα πληθυσμό και υπάρχουν ε, τέτοια παραδείγματα. Δεν ήθελα να αναφερθώ στη δική μου χώρα, γιατί αν αναφερθεί μία τότε οι άλλοι παραπονιούνται, γιατί δεν αναφέρθηκε η δική τους. Γι' αυτό την απέκλεισα. Αλλά νομίζω ότι αύριο θα έχουμε μία εύκολη ψηφοφορία και σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας. Ευχαριστώ. Θα μπορέσουμε λοιπόν να ψηφίσουμε αύριο και για την έκθεση αυτή. Φτάνουμε τώρα στο πακέτο 6 κειμένων. όπου μαζί με τον David Κάζα. David Κάζα, ε, μάλλον εγώ και ο David Κάζα έχουμε αναλάβει αυτό το πακέτο από κοινού. Δεν θα εξετάσουμε αναπερίπτωση αυτό, αυτά τα θέματα της συζήτησης. Πιστεύω ότι θα δούμε τα σημεία που μας απασχολούν και τις διχογνωμίες αν υπάρχουν τώρα. Εφόσον ε, ζητείται η γνωμοδότησή μας από την Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή, θα πρέπει να δούμε καταρχήν την ενίσχυση της εποπτείας της ε, δημοσιονομικής κατάστασης και το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών. Αυτή είναι η πρώτη τροποποίηση του κανονισμού. Έχετε ορισμένες τροπολογίες συμβιβασμού που προτείνονται και θα ήθελα να σας πω ότι το νήμα, ε, ποιο είναι το νήμα που διατρέχει όλες τις ε, προτάσεις συμβιβασμού. Η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιλάει για prudent fiscal policy. Ξέρετε, όσοι ασχολείστε με τη, τις σπουδές οικονομίας, ξέρετε ότι πρόκειται για μια νέα έννοια. Ε, δεν μπορεί να ενταχθεί πουθενά και αποτέλεσε αντικείμενο αρκετών τροπολογιών και τροποποιήσεων. Προτείναμε ως τροπολογία συμβιβασμού να λάβουμε υπόψη το efficient και sustainable και όχι prudent. Η δεύτερη τροπολογία εγκάρσιου χαρακτήρα που διέπει αρκετού συμβιβασμού προτάσει συμβιβασμού που σας προτείνονται αφορά την ΕΠΣΚΟ, το Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ, Απασχόληση Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας και Καταναλωτών, σε σχέση με τις αποφάσεις που λαμβάνει το ΕΚΟΦΗΝ. Ο Γενικός Διευθυντής Απασχόλησης ακριβώς αυτό μας είπε. Όταν η Επιτροπή ε, εξετάσεις προτάσεις αναχώρα μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η ΕΚΦΙΝ και η ΑΜΠΛΟΑ θα ασχοληθούν με αυτό το θέμα. Θα δούμε δηλαδή πώς έχει αυτή η διάρθρωση σε επίπεδο Συμβουλίου για να ορίσουμε τις προτάσεις με βάση το άρθρο 148 που επιτρέπει τον συντονισμό των πολιτικών απασχόλησης. Η τρίτη εγκάρσια τροπολογία που βρίσκουμε στους συμβιβασμούς αφορά τον συνεκτικό χαρακτήρα μεταξύ ενίσχυσης δημοσιονομικού χαρακτήρα και συντονισμός οικονομικών πολιτικών μέσα στα πλαίσια της ε, στρατηγικής 2020, μετά από τις συζητήσεις που είχαμε. Επειδή πρόκειται για μια πρόταση νομοθετικού περιεχομένου, αναφερόμαστε σε μια συγκεκριμένη, δεν αναφερόμαστε σε μια συγκεκριμένη στρατηγική, γιατί πρόκειται για ένα πλαίσιο αναφοράς για τα, για τα επόμενα 50 χρόνια. Άρα αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το περιεχόμενο αυτής της στρατηγικής και γι' αυτό μιλάμε για ανάπτυξη και απασχόληση στη τροπολογίες συμβασμού. Ως προς το πρώτο αυτό θέμα θα ήθελα να σταθώ στους συνδυασμούς K, K και S σε σχέση με το συνταξιοδοτικό όπου σε συμφωνία με τον κύριο Κάζα και με άλλους ε, συναδέλφους προτείναμε μια γενική σύνταξη που δεν προδικάζει τα συνταξιοδοτικά συστήματα τα οποία θα τεθούν σε εφαρμογή στα διάφορα κράτη-μέλη. Δηλαδή κάθε κράτος μέλος μέσα στα πλαίσια των ε, δημοσιονομικών θα πρέπει να δει κατά πόσο μπορεί να υποστηρίξει το συνταξιοδοτικό του σύστημα και δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να ασχοληθεί με αυτό το θέμα, όπως είπαμε και στην έκθεση ο Μενορόιτεν, να αποφανθούμε κατά πόσο μια χώρα θα πρέπει να δεχτεί ένα συνταξιοδοτικό σύστημα με κεφαλαιοποίηση ή με κατανομή ή με επιμερισμό. Ανοίγουμε λοιπόν τη συζήτηση και δίνω το λόγο στον κύριο Κάζα σε πρώτη φάση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα προτιμούσα, πρέπει να πω, να είχαμε μια συζήτηση για όλες αυτές τις εκθέσεις Φέρικα, διότι έχουμε τροπολογίες που θα μπορούσε να βρει κανείς και να εντάξει σε όλες αυτές τις εκθέσεις θεματολογικά. Θα μπορούσαμε αυτά τα θέματα να τα εξετάζαμε δηλαδή, ας το πω έτσι, εκ του είναι πιο, πιο, από πιο κοντά. Όμως πρώτα απ' όλα, πρωτού ξεκινήσω συζητώντας αυτό το, με τη συζήτηση αυτού, αυτού, αυτού του χαρτοφυλακίου, πρέπει να πω ότι υπήρξαν πολλές ιδέες οι οποίες προτάθηκαν όσον αφορά την σύνεση όσον αφορά φορολογικά και δημοσιονομικά θέματα. κάνει τη συνάντηση των σκιωδών εισηγητών, νομίζω μια εγκάρσια τροπολογία καταφέραμε να πετύχουμε που βελτιώνει την διατύπωση για την αποτελεσματικότητα και για την αηφορία. Είναι ένα συμβιβασμό, θα έλεγα, που όλοι μπορούμε να υποστηρίξουμε από κοινού. Αυτό που χρειάζεται είναι να θυμόμαστε πάντα ότι υπάρχει κάτι που πρέπει να αναγνωρίσουμε. Πολλή δουλειά έγινε σε αυτές τις εκθέσεις. Είχαμε πολλές συναντήσεις με πολλούς ε, ε, ε, κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους. Δεν ήταν εύκολο και σε σχέση με τους ευρωβουλευτές και τις ομάδες τους να καταλήξουμε στους συμβιβασμούς που πετύχαμε. Ήδη πρωτού ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση θα ήθελα να σας ενθαρρύνω να δείτε αυτές τις τροπολογίες, τις συμβιβαστικές υπό αυτό το πρίσμα ακριβώς. Γιατί αν καταψηφιστούν κάποιες από τις τροπολογίες, κάποιες από τις συμβιβαστικές τροπολογίες, θα έχουμε χάσει τα πάντα νομίζω. Θα έχει το σύνολο απολεστεί. Και είχαμε και αρκετές ιδέες για το τι θα έπρεπε να γίνει όσον αφορά τα κονδύλια, αποκυρώσεις, πρόστιμα κτλ. Και εδώ είχαμε συμβιβασμό σε ένα κείμενο που διατυπώνει την επιθυμία μας να μεριμνήσουμε ώστε αυτά τα κονδύλια να καταλήξουν στο Ευρωπαϊκό Μέσο για την Σταθερότητα και την ε, Ευρωπαϊκό Μέσο Διευκόλυνσης ε, Δημοσιονομικής Σταθερότητας και όσον αφορά το σημείο 9 στο, στην ημερήσια διάταξή μας ε, προβλέπεται ότι ο κανονισμός 1156 saving effect θα βελτιωθεί. Ως ομάδα δεν θέλουμε να διαγραφεί ο όρος ε, προς εξοικονόμηση, αποτελεσματική εξοικονόμηση κονδυλίων. Ενώ συμφωνώ λοιπόν με τις παρατηρήσεις που έκανε η Πρόεδρος, ε, το αναφέρω αυτό. Έχουμε ένα πρόβλημα όσον αφορά αυτή, αυτές τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Και έτσι δεν μπορούμε δυστυχώς να υποστηρίξουμε τις τροπολογίες 18, 29, 41, 52, και 69. ή τον συμβιβασμό J, το Ι. Κατά τα άλλα, συμφωνώ με αυτά που αναφέρθηκαν από την Πρόεδρο προηγούμενα. Ευχαριστώ. Euh, Ευχαριστούμε. Εντάξει, εκείνη είναι η συζήτηση. Έτσι ξεκινήσατε κι εσείς. Μια αναφερθήκατε στις κυρώσεις, θα επανέλθω κι εγώ. Αλλά να στραφώ και στους άλλους συναδέρφους. Μήπως θέλει κάποιος το λόγο. Παρακαλώ, κύριος Κρότσμαν. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Χαιρετίζω αυτά που αναφέρθηκαν από τον συνάδελφο τώρα τελευταία. Είχαμε διαφορετικές απόψεις. Δεν θέλαμε τα κονδύλια αυτά μεταξύ των κρατών μελών ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επενδύονται έτσι, αλλά θέλαμε για τον μηχανισμό, ευρωπαϊκό μηχανισμό κρίσης ε, να συνεισφέρουν και γι' αυτό το χαιρετίζουμε αυτό. Χαιρετίζουμε επίσης την πρόταση του εισηγητού όσον αφορά την απαγόρευση των υψηλών ελλημάτων ή του υψηλού χρέους και να ξεκινήσουν οι διαδικασίες κύρωσης. Εμείς οι φιλελεύθεροι είμαστε κατά της χαλάρωσης των διαδικασιών και των προτάσεων όπως έχουν προταθεί. Δυστυχώς εδώ υπάρχουν πολλά στοιχεία που ε, στοχεύουν στη χαλάρωση και δεν μπορούμε να τα δεχτούμε. Και επειδή θέλω να συνεχιστεί η συζήτηση, θα ήθελα τη μία ή άλλη παρατήρηση να την κάνω υστερότερα. Όσον αφορά το sustainable, την αποτελεσματικότητα, συμφωνούμε με αυτό και το έχουμε ήδη προαναφέρει. Ευχαριστώ. Merci, Μάλιστα, πρώτα σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε εσάς. Επίσης ευχαριστώ για τις τροπολογίες και τις συμβαστικές τροπολογίες που έχουμε. Έτσι μπορούμε να έχουμε μια βάση που θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε. Θέλω να επισημάνω ότι στον συμβιβασμό ΔΕΛΤΑ, D, η ε, έννοια του social downturn, δεν ξέρω ακριβώς τι εννοεί social downturn, τι μπορεί να είναι αυτό, κοινωνική επιδείνωση ή απομείωση και δεν ξέρω τι θα σημαίνει αυτό σαν συνέπεια αυτής της διατύπωσης, διότι τη στιγμή εκείνη όπου υπάρχει επιδείνωση κοινωνική, δηλαδή σε δείκτες κλειδιά ή άλλους δείκτες που έχουν σημασία για την ανεργία η έννοια επιδείνωση τι σημαίνει. Να πούμε ότι από τη στιγμή που διαπιστώνεται κάτι τέτοιο μπορεί κανείς στην πολιτική του να παρεκκλίνει από κανόνες. Τι εννοούμε. Εδώ έχω προβλήματα και έχω αμφιβολίες αν κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει και αν κάτι τέτοιο είναι όριμο όσο αφορά τη σύλληψή του. Δεν νομίζω ότι αυτό έχει ε, εντάσει στις δικές μας αρμοδιότητες, αλλά είναι στις Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ. Ε, δεν υπάρχουν άλλοι ομιλητές. Ως προς τις τροπολογίες 18, 29, 41, 69 και μία άλλη που δεν κατέγραψα, που αναφέρατε. «96». 18, 29, 41, 69, 96 λέει πρόεδρο. Να Νομίζω κι άλλη μία υπάρχει. Α, όχι, εντάξει, καλώς. Θα τις κοιτάξουμε ως προς το συμβιβασμό. J. Αυτή η συζήτηση έγινε. Νομίζω ότι είναι σημαντική αυτή η τροπολογία, διότι η διάρθρωση όπως προτείνεται μεταξύ των στόχων που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η δημοσιονομική πολιτική όπως θα τεθεί από τα κράτη-μέλη είναι δύο αλληλένδετα ζητήματα. Αν θέλετε μπορούμε να δεχτούμε μία εναλλακτική διατύπωση αλλά θα πρέπει να παραμείνουμε στο πνεύμα της ε, χρησιμότητας της στρατηγικής Ευρωπαϊκή Ένωση 2020 έναντι των στρατηγικών των κρατών μελών. Διαφορετικά δεν βλέπω πώς θα μπορούσε να προωθηθεί διαφορετική διάρθρωση. Διαφορετικά θα βρεθούμε στο ίδιο σημείο με τη στρατηγική της ε, Λισαβόνας. Δηλαδή ωραία και παχιά λόγια και στη συνέχεια το ΕΚΤ, τα κράτη-μέλη μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν χωρίς να τηρήσουν τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020 ή μπορεί τα κράτη-μέλη να προβάλλουν δημοσιονομικές στρατηγικές που δεν τηρούν το πλαίσιο του 2020. Δεν είναι ο σωστός τρόπος διεκπαιρέωσης. Ως προς την τροπολογία συμβιβασμού ΔΕΛΤΑ, νομίζω ότι υπάρχει πραγματικός κίνδυνος, δηλαδή εάν η κοινωνική ε, κατάσταση επιδεινωθεί, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να λάβουν ε, έκτακτα μέτρα. Αλλά για να ικανοποιήσουμε τον κύριο Γκίγκολτ, μπορούμε σε αυτή την τροπολογία συμβασμού να έχουμε ξεχωριστή ψηφοφορία ως προς τον όρο social Ε, μου κάνει εντύπωση όμως το ότι στάτε κάτι τέτοιο, δηλαδή να απαλληφθεί ο όρος κοινωνικός, κοινωνικά. Ο κύριος Κάζα θέλει να παρέμβει εκ νέου. Ναι. Σε σχέση με το J, με την πρώτα σύμβαση μου, αρχικά είχαμε προτείνει μια διαφορετική διατύπωση η οποία ίσως να είχε γίνει αποδεκτή από όλους. Όμως δεν έγινε δεκτή αρχικά. Ίσως όμως πριν από την αυριανή ημέρα να βρούμε μια διαφορετική διατύπωση η οποία να περιλαμβάνει τις λέξεις cost saving effects θα δούμε πώς μπορούμε να παλύψουμε αυτές τις ε, δυσκολίες έτσι ώστε να φτάσουμε σε ένα συμβιβασμό που να γίνει αποδεκτός από όλους. Um, on the Ως προς το J, αυτό το συμβιβασμό, θα ήθελα εντάχει να πω ότι η διατύπωση της Επιτροπής είναι κάπως ε, περίεργη, διότι όταν μιλάμε για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις δεν έχουν μακροχρόνιες επιπτώσεις εξοικονόμησης. Μπορεί να γίνει η εξοικονόμηση, αλλά όχι άμεσα. Και αυτό δεν ισχύει εάν υπάρχει ενδυνάμει ανάπτυξη. Θα ήμουν πολύ προσεκτικός σε αυτή τη διατύπωση. Θα δεχτώ ένα συμβιβασμό, όχι κρατώντας την παλαιά διατύπωση, όμως διότι είναι καθόλου λογική. Δεν έχει λογική συνέπεια. Ως προς τα σχόλια, τα δικά σου περβάνς, πάλι είναι θέμα ορισμού. Το ζήτημα είναι πώς ε, διαμορφώνεται η κατάσταση και πού μπορούμε να ε, επιτρέψουμε επιπρόσθεο έλλειμμα. Ε, όταν μιλάμε για κοινωνική επιδείνωση σημαίνει ότι υπάρχει μεγαλύτερη ανισότητα, ανισορροπία μεταξύ ανδρών και γυναικών. Δηλαδή, όταν μιλάμε για οικονομική επιδείνωση, γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνει υπό οικονομικούς όρους, αλλά υπό δεν το ξέρουμε. Εάν υπάρχει οικονομική επιδείνωση και αυξανόμενη ανεργία, αυτός είναι ένας λόγος απόκλησης των ε, κρατών. Και υπ' αυτή την έννοια η τροπολογία συμβιβασμού κινείται πέραν από τις ε, προτάσεις της Επιτροπής. Αλλά υπάρχει κάποια ασάφεια με αυτό τον όρο, η οποία δεν γίνεται κατανοητή από μένα τουλάχιστον. Άρα για να είμαστε σαφέστεροι, θα πρέπει να μιλάμε για έκτακτη ή μη προβλεπόμενη ανεργία. Κύριε Κάζα, τι λέτε. είναι θέμα ερμηνείας. Όλα αυτά είναι θέματα ερμηνείας. Κατανοώ αυτά τα οποία λέει ο συνάδελφος. Είναι όμως θέματα ερμηνείας αυτά. Εμείς τα ερμηνεύουμε διαφορετικά, τα ερμηνεύσαμε. Προτείναμε λοιπόν το cost saving effects να αντικατασταθεί από το wealth creation, creation effects Αντί να εξοικονομήσουμε κόστος, να έχουμε μέτρα τα οποία θα προαγάγουν τη δημιουργία πλούτου. Ας αναμείνουμε να δούμε σε σχέση με την ερμηνεία αυτή και από την έκβαση αύριο. Είναι τελείως διαφορετική όμως η ερμηνεία αυτή από την άλλη ερμηνεία που δόθηκε από τον συνάδελφο. Ευχαριστώ. Μικρόφωνο, δεν ακούστηκε. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με το Συμβασμό 2 και τον Τζέι, αλλά νομίζω ότι υπάρχει σύγχυση ως προς το στόχο του κυρίου Γκίγκολτ σε σχέση με το Τζέι. Ο κύριος Κάζα εκ νέου. Έχετε το λόγο. Μιλάτε για το D ή για το J γιατί αν σχετίζεται με το τι μπορώ να το δεχτώ. Α, εντάξει, εντάξει, με συγχωρείτε πρόεδρε. Ε. Έχω Εγώ έκανα λάθος. Άρα η δέλτα τροποποιείται και στη λέξη του social μιλάμε για ανεργία, εκ, ιδιαίτερη, ιδιαίτερα υψηλή ανεργία. reviens Ή να βρούμε μία προφορική για αύριο και κύριε Κάζα θα επανέλθετε στο EJ. Σας προτείνω, γιατί δέχομαι την υπόδειξή σας να έχουμε μία συνολική συζήτηση, έχω την εντύπωση, είχα την εντύπωση ότι θα ήταν ε, καλύτερα να το δούμε αναθέμα, αλλά αν θέλετε μπορούμε να τα δούμε τα υπόλοιπα πέντε συλλήβδιν και σας δίνω το λόγο για να μας κάνετε μια εισαγωγή. Στο δεύτερο μέρος της συζήτησης θα ήθελα όμως να πω λίγα λόγια ως προς τη χρήση των κυρώσεων, σε σχέση δηλαδή με τις προτάσεις Κρόιτσμαν, διότι στο συμβιβασμό είχαμε προτείνει το πλαίσιο κυρώσεων να σχετίζεται με διαφορετικές χρήσεις για την χρηματοδότηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και για την υποστήριξη της σταθερότητας των κρατών μελών. Ο κύριος Κρόιτσμαν μας είπε ότι αυτή η διατύπωση δεν τον βρίσκει σύμφωνο. Άρα εφόσον δεν δέχεται το συμβιβασμό, τότε δεν ισχύει. Εγώ όμως θα ήθελα να τον κρατήσουμε. Απλώς ο κύριος Κρόιτσμαν θα πρέπει να μας πει αν μπορεί να τον δεχτεί υπό όρους. Δηλαδή ο κύριος Κρόιτσμαν μιλάει για τα χρήματα από τις κυρώσεις που θα ε, πρικοδοτούν το Ταμείο Σταθερότητας, ενώ η τροπολογία συμβιβασμού μιλά για τη σταθερότητα και άλλες χρήσεις, δηλαδή την χρηματοδότηση των γενικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να το αποσαφηνίσουμε, τη θέση των μεν και των δε. Κύριε Κάζα, έχετε το λόγο για τη συνέχεια της παρουσίασης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το σημείο 10 συζητάμε τώρα στην ημερήσια διάταξη, που είναι το 522 για τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Το πιο σημαντικό θέμα στη συζήτηση εδώ ήταν το τι μπορούμε να καθορίσουμε και πώς θα προχωράμε με την διαδικασία αυτή. Τα κύρια ζητήματα έχουν να κάνουν με το πώς θα ερμηνεύουμε το κείμενο. Υπάρχει το παράδεκτο που έχει να κάνει με την ε, μεταρρύθμιση, αλλά το σύστημα πολλαπλών πυλώνων το βγάλαμε. Γιατί θέλουμε να παραμένει ότι η μεταρρύθμιση των συντάξεων θα έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις και συνεπώς η μεταβατική περίοδος των 5 ετών έφυγε. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να πετύχουμε συμβασμούς και για άλλες τροπολογίες. Αλλά βέβαια ήμασταν κατά όλων των τροπολογιών που πρότειναν να βγαίνουν ολόκληρα κομμάτια από το κείμενο. Όπως για παράδειγμα να διαγραφούν ολόκληροι συμβιβασμοί αυτό ισχύει βέβαια και για τα άλλα θέματα που θα συζητήσουμε σε λίγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δεν έχει νόημα, πρέπει να πω, και θέλω να απαντήσω. Τα πρόστιμα να μην είναι τόσο λέει ψηλά, ώστε να μην δίνουν ένα αξιόλογο ποσό ώστε για περαιτέρω κρίση τα χρήματα αυτά να μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Γι' αυτό έχει πολύ μικρό νόημα τα μικρά αυτά ποσά που κατά τη διάρκεια των ετών ίσως θα μπορούσαν να συναθρήσουν μεγάλα ποσά να χρησιμοποιηθούν για διαφορετικό σκοπό. Παραμένω στην παρατήρησή μου. Αρχικός στόχος είναι τα έσοδα των κυρώσεων να χρησιμοποιούνται για τον αρχικό σκοπό για τον οποίο είχαν συλληφθεί. Δηλαδή να υπάρξει πρόληψη, να έχουμε χρηματοοικονομικά μέσα ώστε αν υπάρξει τέτοια κρίση να μπορέσουμε να βοηθήσουμε από αυτά τα κονδύλια πάλι. Ευχαριστώ. Simplement, Πρόεδρος, αντιλαμβάνομαι την ανησυχία σας. Όμως η διευκόλυνση για την δημοσιονομική σταθερότητα των χωρών μελών δεν αποφασίστηκε για τον ε, μηχανισμό αντιμετώπισης. Η διευκόλυνση αυτή Αλλιώς, διακόπτη η Πρόεδρος, ο κύριος Κρότσον. Όχι πρόεδρε, αλλά συνεισφέρουν. Θα είναι μια μικρότερη συνεισφορά σε σχέση με τις κυρώσεις. Αλλά με αυτή την μετριόφρονα συνεισφορά για μελλοντικές ε, κρίσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Γιατί διαφορετικά σε σχέση βέβαια με τα, ε, ε, τα πρόστιμα αυτά δεν επαρκούν να επιληθεί η κρίση αλλά μπορούν να συνεισφέρουν. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, είναι σημαντική αυτή η συζήτηση γιατί το ζήτημα είναι πρώτον σε τι χρησιμεύουν τα χρήματα που παίρνουμε από τις κυρώσεις αυτές και δεύτερον πώς χρηματοδοτείται ο μηχανισμός, αυτό που λέμε σήμερα διευκόλυνση και μεθαύριο θα είναι ο μηχανισμός. Δεν υπάρχει αυτόματη σύνδεση των δύο. Η συζήτηση που έγινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την έκθεση Προκ Γκουαλτιέρη των συναδέρφων έδειξε ότι υπάρχει προοπτική να έχουμε έναν πιο κοινοτικό μηχανισμό και άρα όχι αναγκαία μια χρηματοδότηση που να βασίζεται στην διακυβερνητική διάσταση. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι η ιδέα ότι τα χρήματα αυτά δεν πρέπει να χρησιμεύσουν παρά για να βοηθούν τις χώρες που βρίσκονται σε κρίση, στο το κάνουμε μεθαύριο μπορεί να μην υπάρχει κρίση, αλλά να υπάρχουν χώρες οι οποίες αποκλίνουν. Τι θα κάνουμε με τα χρήματα αυτά. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψη του κύριου Κάσα. Αλλά τότε ας ψηφίσουμε τις τροπολογίες χωρίς συμβασμό. Κύριε Κάζα, τι λέτε. Όπως είπα και στην αρχή της παρέμβασής μου, συμφωνούμε με τον ε, συμβιβασμό που προτείνεται, γιατί δείχνει την βούλησή μας οι πόροι αυτοί, τα χρήματα αυτά, να πάνε την ε, διευκόλυνση για την οικονομική σταθερότητα. Είναι ο συμβασμός που συζητήσαμε πριν από μερικές μέρες στη συνεδρίασή μας, όπου είπαμε και πάλι γιατί η ομάδα μου δεχόταν κάτι τέτοιο. Τόμας Μαν. Ευχαριστώ. Σήμερα σε ένα μικρότερο κύκλο είχαμε ευκαιρία με δύο ή τρεις σημαντικές προσωπικότητες να συζητήσουμε. Ο κύριος Ρόμπαϊ, ο πρώτος, ο οποίος στην Επιτροπή ΕΚΟΝ είπε τι έγινε με την Task Force και είπε πόσο σημαντικό είναι το σύμφωνο σταθερότητας και ότι θέλουμε να υπάρξουν μέσα τα οποία θα τροφοδοτούν αυτό το μέσο. Είναι σημαντικό αυτό σε σχέση με την Task Force. Και το δεύτερο ήταν η ανοιχτή συνάντηση των συντονιστών σε σχέση με την ΕΚΟΝ. Είχαμε δύο υπουργού εκεί που προσήλθαν οι οποίοι κάθονται ένας δίπλα στον άλλον επειδή έχουν και καλή κατανόηση. Είχαμε από τη Γερμανία και την ε, άλλη υπουργό που κατανοούν ο ένας τον άλλον θέλουν να είναι πρότυπα και θέλουν να έχουν ηγετικό ρόλο που θα διαδραματίσουν. Το καλύτερο θα ήταν αν μπορέσουν να διαδραματίσουν αυτό το ρόλο αλλά να μην το ε, μάθουν όλοι ώστε να μην ε, ε, υπάρξει εντύπωση ότι υπάρχει διπλή κινητήρια δύναμη. Αλλά αν γίνεται αυτό και τότε μπορούμε να καταλήξουμε σε μια ε, προσέγγιση της σταθερότητας και συνεισφέρουν, τότε έχει δίκιο ο κύριος Κρότσμαν να πει ότι αυτά τα πρόστιμα στην αρχή είναι πολύ μικρά ποσά. Δεν μπορούν να σώσουν αυτόν τον πολιτισμό σταθερότητας ή την προσέγγιση σταθερότητας. Είναι όμως μια σημαντική συνεισφορά για την χρηματοδότηση και έτσι σταδιακά θα μπορέσει να διαδοθεί στα κράτη-μέλη μια ευαισθησία για τη σταθεροποίηση και τη σταθερότητα. Αυτό δεν συνέβη ακόμα. Η Γαλλία και άλλες χώρες ε, ε, που έχουν μια ε, τοποθέτηση όμως το να βασιστεί κανείς ότι θα έχουν triple A για την χρηματοδότηση όλοι αυτοί δεν μπορεί να διασφαλίσει μακροπρόθεσμα. Να μην ξεχνάμε ότι αναμένουν οι πολίτες να γίνει κάτι για να συμμετάσχουν άλλες χώρες Κάποιοι επώδυνα αναγκάστηκαν οδυνηρά να μάθουν αυτά τα μαθήματα, αλλά και οι Ιρλανδοί θα πρέπει από ε, παλιές τους συνήθειες να απόσχουν, να παρεκκλίνουν. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα να δράσουμε παρά μόνο αυτή. Λοιπόν, η έννοια με το ειδικό μέσο ειδικό μέσο είναι σημαντική προσέγγιση. Συμφωνώ με αυτό σε σχέση με αυτό το πεδίο, με αυτό το θέμα για, με τον κύριο Κρόισμαν. Ίσως σε σχέση με τη σταθερότητα και σταθεροποίηση θα πρέπει να αποτελέσει θεμέλια για μας. Ίσως εκεί του συναδέλφου Γκίγκορ θα τον είχαμε και στο πλευρό μας αν καταφέρναμε κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Βλέπω το συμβασμό ως έχει. Εάν πρέπει να άρουμε το if, το including, τότε γιατί αντιτάσσεστε εσείς. Τι σας ενοχλεί το including. So this the compromise would Δηλαδή και θα χρησιμοποιηθεί υποστηρίζον... Κύριε Κρόιτσμαν, μπορείτε να συμφωνήσετε και θα χρησιμοποιηθεί για να φτάσουμε στους στόχους επένδυσης και απασχολησιμότητας με βάση τους μηχανισμούς ε, σταθερότητας χρησιμοποιώντας χρηματοδότηση για οικονομικά βιώσιμη και ε, αποδεκτή, επέμβαση, ε, επένδυση. Με συγχωρείτε. Um, Συμφωνούσατε κύριε Κρότσμαν. Euh, Ωραία, συμφωνούμε. Και ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κάζα για τη βοηθειά του. Για τις διάφορες εκθέσεις, κύριε Κάζα, έχετε να πείτε κάτι ακόμα. Για τελειώς θα ήθελα να πάμε στην έκθεση 527. Εκτός αν έχετε κάτι άλλο εσείς να πείτε. Αφού είπατε να πάμε μία έκθεση μετά την άλλη, περνάω στην επόμενη έκθεση. Και πρόκειται για την έκθεση 524. σημεία 11 στην ημερήσια διάταξη. Εδώ πρόκειται για την έννοια των κινήτρων και των κυρώσεων. Μπορώ να συμφωνήσω με τις περισσότερες από τις τροπολογίες που υποβλήθηκαν. Κάποιε έχουν υποβληθεί από τον συνάδελφο Κρότσμαν. Αυτές που έχουν να κάνουν ε, με το υπερβολικό χρέο και το τι πρέπει να ληφθεί υπόψη για την εποπτεία του προπολογισμού, συμφωνώ με τι τροπολογίε αυτές. Είμαι κατά όμως όλων των τροπολογιών που θέλουν να αλλάξουν το σύστημα απόφασης στο Συμβούλιο. Ο μηχανισμός πρέπει να υποβάλλεται σε ημι-αυτοματισμό και είμαι κατά των τροπολογιών που αναφέρονται σε δομές που δεν υπάρχουν. Είμαι υπέρ της διασφάλισης ισχυρού ρόλου για το Κοινοβούλιο στη λήψη αποφάσεων κάθε φορά που αυτό ενδείκνυται. Συγχρόνως πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές. Αυτά είχα να πω. Για τις υπόλοιπες τροπολογίες συμφωνώ μαζί τους. Οπότε έχουμε συμφωνήσει στο συμβιβασμό. Ο κύριος Κρότσμαν, μήπως ο κύριος Γκίγκολτ. Όχι. Λέει η Πρόεδρος. Για το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχετε υπόψη σας κάποια συγκεκριμένη τροπολογία και το είπατε. Κύριε Κάζα. Ποιες είναι οι τροπολογίες που σας δημιουργούν πρόβλημα. Well, I don't have... Δεν έχω μεγάλα προβλήματα, απλώς υπήρχαν κάποιες τροπολογίες. ούτες. Ο συμβασμό D που συζητήσαμε πριν. Όχι, όχι. Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη τροπολογία. Αντικατοπρίζονται στο συμβασμό. Πρόεδρος, άρα δεν υπάρχει ιδιαίτερη δυσκολία εδώ, ωραία. 524. εφαρμογή της δημοσιονομικής εποπτείας για αποτελεσματική δημοσιονομική εποπτεία στα κράτη-μέλη στη ζώνη ευρώ. Κύριε Κάσα. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι λέει η πρόεδρο. Έχετε δίκιο. Λάθο έκανα εγώ. Είμαστε στο δημοσιονομικό πλαίσιο 523, σημείο 12 στην ημερήσια διάταξη. Έχουμε 18 τροπολογίες εδώ. Τώρα κύριε Κάζα, γι' αυτό. Θα συζητήσουμε την ε, έκθεση 523 για, στο σημείο 12 της ημερήσιας διάταξης για τα δημοσιονομικά πλαίσια. Χαίρομαι για τις ε, τροπολογίες που έχουν υποβληθεί από την ε, Πρόεδρο, από την κυρία Μπερές και νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε μια καλή πλαισίωση για τον προϋπολογισμό με βάση τις βέλτιστες πρακτικές των κρατών μελών. Με βρίσκει σύμφωνο αυτή η ιδέα. Επίσης συμφωνούμε με το κείμενο της τροπολογίας 16, δηλαδή να αναφερθούμε σε αυτή την πλαισίωση που να μην είναι τόσο αυστηρή και έτσι να αντικατοπτρίζει τις ανάγκες των κρατών μελών. Ως προς το θέμα αυτό δεν έχω τίποτα άλλο να προτείνω. Άλλοι συνάδελφοι που θέλουν να παρέμβουν, λέει πρόεδρος, όχι, άρα θα ψηφίσουμε και αυτή την έκθεση αύριο. 527 τώρα. Έκθεση 527 για την πρόληψη και διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών όπου υπάρχει μία σειρά τροπολογιών συμβιβασμού που συμπεριλαμβάνουν αυτό που είπαμε σε σχέση με το πρώτο θέμα, τα όσα είπαμε για το πρώτο θέμα Και εδώ έχει σημασία να δούμε πώς θα έχει η εποπτεία των ε, μακροοικονομικών ανισορροπιών και να δούμε πώς θα προληφθούν. Ο κύριος ε, Κάζα, κύριε Κάζα, συμφωνούμε, έτσι δεν είναι, και αυτό αφορά και τον κύριο Κρόιτσμαν και Γκίγκολντ. Θα θέλαμε να υπάρχει ένας πίνακας για να εποπτεύουμε τις ε, μακροοικονομικές ανισορροπίες και με κατεξουσιοδότηση πράξης ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορέσει να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία πρόληψης και διόρθωσης. Αυτό είναι το πρώτο. Και δεύτερον, θα πρέπει να επαληθεύσουμε και να δούμε πώς θα προτείνουμε κατευθυντήριες γραμμές για το περιεχόμενο αυτού του πίνακα, αυτού του βαθμολογίου και να το κάνουμε με έναν ενδεικτικό κατάλογο στο ε, παράτημα των νομοθετικών πράξεων. Αυτά είναι τα στοιχεία συμβιβασμού επί του κειμένου αυτού. Ο κύριος Κάζα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πιστεύω ότι το πιο σημαντικό σημείο για μας είναι ο πίνακας επιδόσεων, scoreboard και οι συντελεστές, οι παράγοντες εκείνοι που θα έπρεπε να ενταχθούν μέσα σε αυτό το πίνακα επιδόσεων. Είμαστε λοιπόν υπέρ ενός μικρού, μικρών διαστάσεων πίνακα επιδόσεων και καλά προσδιορισμένου με όρους και προϋποθέσεις. Συμφωνώ με του συναδέλφους άλλα με τον κύριο Γκίγκορντ ότι εμεί ω Ευρωκοινοβούλιο θα δρατώμεθα τη ευκαιρία και θα προτείναμε τι θα έπρεπε να ενταχθεί στον πίνακα αυτών των επιδόσεων. Ωστόσο θα ήταν πρόημο πιστεύω να καθορίσουμε έναν εξαντλητικό κατάλογο σε αυτή τη φάση. Παρ' όλα αυτά όμω, ένα αριθμό εξαιρετικών ιδεών προδιατυπώθηκαν και προήχθησαν και αυτό θα έπρεπε να αποτελεί και μέρος αυτού του χατοφυλακίου. Ο συμβιβασμό στον οποίο καταλήξαμε τοποθετεί τέτοιες προτάσεις ε, που δεν θα είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα, αλλά που θα μπορούν ενδεικτικά να χρησιμοποιηθούν για αυτά που θεωρούμε ότι θα έπρεπε να συναποτελούν μέρος του πίνακα επιδόσεων. Θα μπορούσαν και μελέτες να υποβληθούν πιο εξειδικευμένες σε υστερότερη φάση. Δεν συμφωνούμε από την άλλη πλευρά ότι οι ανισότητες θα έπρεπε να αναφέρονται και στη συνέχεια δεν θα έπρεπε να τύχουν εξέτασης ως ανισότητες στη συνέχεια. Γι' αυτό δεν μπορούμε να είμαστε υπέρ όπως ε, προεπιχειρηματολογήσαμε ε, και δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε τους ε, συμβιβασμούς I, K και H. Ωστόσο όμως, αν μπορούμε να βρούμε κάποιες συμφωνίες μέχρι αύριο, συμβιβαστικά, θα εξετάσουμε τη συζήτηση και αλλαγή της θέσης μας. Ευχαριστώ. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention Άλλος κανείς Κύριε Κάζα, για την Η δυσκολία σας που έγινε στο, στο πλεόνασμα, στο επιπλέον, να έχουμε χωριστεί κατά τμήματα ψηφοφορική. Ναι, δεν μας αρέσει το excessive surpluses. Γιατί δεν πιστεύουμε ότι αυτό αποτελεί στοιχείο ανισορροπίας. Να είναι μια ανισορροπία, λέει πρόεδρος, άμα κοιτάξουμε την κατάσταση στην Κίνα. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Κιγόλ και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε με τον κατάλογο ψηφοφορίας για αύριο. Κύριε Κιγόλ. Πρέπει να σχολιάσω για δύο πράγματα. Πρώτον, εκπλήσωμε. Στο Συμβούλιο, ακόμα και ο κύριος Ρόμπλερ που στηρίζει τη χώρα με το μεγαλύτερο μακροοικονομικό απόθεμα, κανείς δεν λέει ότι δεν πρέπει να αναφέρεται το πλεόνασμα και ούτε υπάρχει κανένα ταμπού να μιλάμε για δυνητικά υπερβολικά πλεονάσματα. Το πρόβλημα είναι κατά πόσο η διόρθωση πρέπει να είναι συμμετρική ή ασυμμετρική. Τη συζήτηση αυτή την είχαμε για πολύ καιρό και στην ε, πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Εγώ προσωπικά και η ομάδα μου πιστεύει ότι πρέπει να έχουμε μια συμμετρική προσέγγιση για να διορθώνονται οι ανισορροπίες αυτές, αλλά άκουσα ότι αυτό δεν πρέπει να αναφέρεται καν. Εδώ έχω πρόβλημα. Και θέλω να σας ζητήσω να σκεφτείτε αν έχετε ένα έλλειμμα, πάντα θα έχετε κάπου αλλού ένα πλεόνασμα. Οπότε, το να μην αναφέρετε το πλεόνασμα, για μένα είναι δυσνόητο, οικονομικά μιλώντας. Έχω και μια δεύτερη παρατήρηση για τη συμβαστική τροπολογία Α. Ε. Ακόμα και αν ε, στηρίζουμε τους κοινωνικούς στόχους, ιδιαίτερα έντονα, είναι λίγο περίεργο να λέμε ότι πρόκειται για τον εντοπισμό κοινωνικών ανισορροπιών. Πρόκειται για μακροοικονομικές ανισορροπίες, οι οποίες μπορεί να έχουν κοινωνικές αιτίες. Γι' αυτό και συμφωνώ απόλυτα με την προσέγγισή σας, κυρία εισηγήτρια και πρόεδρε που θέλετε να συμπεριλάβουμε κοινωνικά κριτήρια στο βαθμολόγιο, γιατί εκεί είναι η θέση τους, εκεί πρέπει να βρίσκονται. Συχνά οι μακροοικονομικές ανισορροπίες έχουν κοινωνικές αιτίες. Όλος στόχος της ρύθμισης αυτής είναι ο εντοπισμός μακροοικονομικών ανισορροπιών. Γι' αυτό δύσκολα θα τις έβαζα στο κοινωνικό. Πάντως για να είμαστε λογικοί. Είναι ένα πολιτικό θέμα είναι νόμος συγχρόνως. Θέλω να είμαι προσεκτικός με τη διατύπωση γιατί δεν ε, τα ξέρουμε πάντα. Και ούτε θέλω να υπεσκελίσω κατά κάποιο τρόπο τους συναδόρφους που βρίσκονται από πίσω εδώ και μπορεί να ξέρουν περισσότερα. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Κάζα για να δούμε πώς θέλει να απαντήσει στον κύριο Κιγόλ για τη συμπερίληψη των πλεονασμάτων, παρόλο που συμφωνώ με τον κύριο Κιγόλ το θέμα των πλεονασμάτων και των ελλημάτων. Εντάξει, αυτό είναι ένα γεγονός. Το θέμα είναι ποιος πρέπει να κάνει τι και πώς. Για τις κοινωνικές ανισορροπίες από την άλλη, δεν ξέρω αν είναι πολιτική αυτή η προσέγγιση ή όχι, διαπιστώνω όμως ότι αν δούμε την προέλευση της κρίσης, οι κοινωνικές ανισορροπίες και άρα οι ανισορροπίες στον κοινωνικό τομέα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο ε, στο ξεκίνημα της κρίσης. Άρα πρέπει να εντοπίσουμε μέσα από το βαθμολόγιο το πώς ε, ξεκίνησαν οι ανισορροπίες αυτές και να παρακολουθούμε το πώς εξελίσσονται αυτές οι κοινωνικές ανισορροπίες. Για μένα δεν υπάρχει έλλειψη συνεκτικότητας εδώ όταν μιλάμε και για μακροοικονομικές ανισορροπίες και για κοινωνικές, αν δεν προχωρήσει ο συμβιβασμός, μπορούμε να κάνουμε και χωριστή ψηφοφορία. Αν είναι στο βαθμολόγιο, είναι γιατί πιστεύουμε ότι τα κοινωνικά δεδομένα μπορούν να οδηγήσουν σε ανισορροπίες. Παρακαλώ κύριε Κρότσμαν. Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να πω έχει δίκιο ο κύριος Γκίγκοτ. Αν πάρουμε το παράδειγμα της Γερμανίας, τότε σίγουρα για το ότι η Γερμανία έχει λέει χαμηλό κοινωνικό επίπεδο δεν μπορεί να το δεχτεί κανείς κάτι τέτοιο έχουμε ένα από τα υψηλότερα όμως εντάξει ας μην ε, συγκρουόμαστε τώρα γι' αυτό ας μην έχουμε πει με αυτό θέμα ναι αλλά κύριε Γκίνκολ το αποφασιστικό γιατί έχουμε μακροοικονομικό πλεόνασμα είναι το ότι τα τελευταία χρόνια εμείς γίναμε πιο ανταγωνιστικοί, πιο ανταγωνιστικοί από άλλες χώρες. Αυτό συνδέεται με το ότι οι συμβάσεις, οι συλλογικές συμβάσεις για παράδειγμα ή το κόστος το μισθολογικό βελτιώθηκαν σημαντικά όσον αφορά τις ε, επιβαρύνσεις. Είμαστε πιο ανταγωνιστικοί για τις εξαγωγές. Στις παγκόσμιες αγορές είμαστε πιο ανταγωνιστικοί. Μπορούμε τα εμπορεύματά μας να τα διοχετεύσουμε, να τα διαθέσουμε στις παγκόσμιες αγορές. Αυτό είναι αποφασιστικό αν έχω πλεόνασμα ή έλλειμμα κύριε Γκίγκολ. Όλοι θα χαιρόμαστε αν είχαμε πλεονάσματα όλες τις χώρες. Δυστυχώς δεν υπάρχουν αυτά τα πλεονάσματα. Υπάρχουν ελλείμματα, διότι η ανταγωνιστικότητα πολλών χωρών δεν διασφαλίστηκε όπως θα έπρεπε. Και αυτό είναι κύριο πρόβλημα. Και γι' αυτό θίγεται το σωστό πρόβλημα, με σωστό τρόπο ότι ο πίνακας επιδόσεων πρέπει έτσι να εξεταστεί όσον αφορά τα αίτια, που ε, συνεπάγονται αυτή την κατάσταση. Πρόκειται για μακροοικονομικές όμως, ε, μακροοικονομικά ελλείμματα, όχι κοινωνικά ελλείμματα. Θέλω να το ξανααναφέρω αυτό. Και κύριε Κίγκολτ, όταν έχουμε τη συνδιαχείριση στα εργοστάσια στην Ευρώπη, σε σχέση με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουμε πολύ υψηλό επίπεδο συνδιαχείρισης ε, των συμβαλωμένων μερών στις συλλογικές συμβάσεις στην Γερμανία, στις βιομηχανίες μας και λειτουργεί εξαιρετικά αυτή η συνδιαχείριση αλλά επικεντρώνεται σε θέματα επιχειρήσεων και όχι σε θέματα πολιτικά όταν έχουμε τις διαπραγματεύσεις για τις συλλογικές συμβάσεις και γι' αυτό μπορώ να πω δεν έχει νόημα όλα αυτά να τα συγχαίουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κρόιτσμαν. Εδώ δεν μιλάμε για κοινωνικά ελλείμματα. Μιλάμε για ανισορροπίες, κοινωνικές ανισότητες, οι οποίες ε, οφείλουν να τύχουν αναγνώρισης. Θα πρέπει να υπάρχει συνοχή στο Σύμβασμο Α. Ο κύριος Γκίγκολντ όμως θέλει να παρέμβει και του δίνω το λόγο. Τώρα δεν ξέρω ποια γλώσσα να μιλήσω, αλλά και με εσά κύριε Κρόσμα. Ναι, μιλάμε γερμανικά. Ναι, δεν το αμφισβητούσα καθόλου, λέει σε παρατήρηση χωρί μικρόφωνο. Όταν μιλάμε για τη Γερμανία, α μιλήσουμε και γερμανικά, έστω κατ' εξαίρεση. Το πρώτο σημείο είναι ότι χάρηκα για το ότι είπατε ότι στον τομέα της ανάλυσης, στον πίνακα επιδόσεων scoreboard, ότι υποστηρίζεται λέει τις τροπολογίες μας σε σχέση με αυτό. Καλό αυτό, γιατί υπάρχουν κάποιες άλλες φωνές που λένε να είναι στενό το πλαίσιο του πίνακα επιδόσεων του scoreboard, ώστε σε σχέση με τα αίτια της κρίσης να μην μπορούν να αναλυθούν. Γι' αυτό είναι καλό αν εσείς εκεί εγκρίνετε τον συμβιβασμό, τη συμβαστική τροπολογία για το scoreboard. Πολύ καλό αυτό. Το επιχείρημά μου για τον κύριο Κάζα δεν ήταν εδώ η συζήτηση για πλεονάσματα και ελλείμματα να ανοίξει σε πλήρες μέγεθος γιατί τότε θα ξεπερνούσαμε τα όρια σε αυτή την Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Ήθελα να απευθύνω έκκληση. Αν θα μπορούσε το ΕΛΚ, το PPE, να ακολουθήσει την κατεύθυνση ότι τα πλεονάσματα τουλάχιστον ίσως να δεχτούμε ότι υπερβολικά αναφέρονται εδώ. Όχι ότι ε, δεν θέλουμε να εξεταστούν σε βάθος. Το θέμα όμως του αν θα εξεταστούν σε βάθος είναι άλλο ζήτημα άλλο ζήτημα. Αλλά να δούμε αν θα μπορέσουν να αναλυθούν σωστά και να αναγνωριστούν ως συντελεστές και να δούμε αν με τα πλεονάσματα μπορούμε να καταλήξουμε στο ότι οι μισθολογικές, ας το πω έτσι, οι μισθολογικοί περιορισμοί από πλευράς εργαζομένων είχαν, ε, προώθησαν τις εξαγωγές. Να δούμε όμως ότι μισθολογικά χαμηλών μισθών εργαζόμενοι δεν μπορούν να θεωρηθούν υποχρεωτικά ένα διαρθρωτικό στοιχείο. Δεν οδηγούν σε πλεονάσματα διαρθρωτικά υποχρεωτικά. Αλλά είναι μια συζήτηση που μπορούμε να τη διεξαγάγουμε σε ευρύτερο πλαίσιο και να δούμε τα οικονομικά στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, ποια είναι και να το αποσαφηνίσουμε άλλοτε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τόμας Μάν έχει το λόγο πριν από εσάς. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε μια συνεδρία του Bundestag εδώ. Ναι, αλλά είχαμε και δύο υπουργού ε, σήμερα που συνάντησαμε. Εντάξει, ήθελα αν θα είμαστε μόνο εμείς ανάμεσά μας και ήταν κλειστός ο κύκλος, εντάξει, θα το συζητούσα. Αλλά είμαστε στην ιστοσελίδα, στο, στον, στο δίκτυο και δεν είναι σωστό. Είναι κρίμα να επιβαρύνουμε μόνο μερό στη συζήτηση. Για τον συνάδελφο Κρόισμαν, τα πλεονάσματα συσχετίζονται, λυπούμε για αυτό που θα πω, ότι σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα μάθαμε πολλά πράγματα. Υπάρχουν και τα θέματα των μισθών και για το θέμα των ελάχιστων μισθών ή ελάχιστων εισοδημάτων, εισοδημάτων υπάρχουν διαφορές στις απόψεις. Ότι όμως προχωρήσαμε στην ανταγωνιστικότητα συνδέεται με την ευφυΐα των υπεύθυνων εργαζομένων. Σωστά είπατε, αναφέρθηκε ότι γνωρίζουμε τι θα πει συνυπευθυνότητα. Έχουμε όμως και την αυτονομία στα θέματα, την ε, ε, αυτοδυναμία σε σχέση με τις συλλογικές συμβάσεις και δεν υπάρχει κρατική ανάμειξη. Χρειαζόμαστε κάποια εισοδήματα που πρέπει να είναι συγκεκριμένου επίπεδου. Εντάξει, όταν περάσει η κρίση θα το δούμε αυτό. Αλλά θέλουμε να συνεισφέρουμε να υπάρξει ανταγωνιστικότητα, είπαν οι εργαζόμενοι. Η κυρία Λαγκάντα προσπάθησε να πει ότι εσεί ε, οι Γερμανοί περιορίζετε όλα αυτά. Εμεί τι, τι έγινε στη συνέχεια και κυρία Μπερές εσείς θα το πείτε ήταν μια καλή απόφαση προσκλήθηκε ως μια Γαλλίδα υπουργό να συμμετάσχει σε μια συνάντηση της γερμανικής κυβέρνησης των υπουργών, υπουργική ε, συνεδρία και όταν συζητήσαμε αυτά ο ένας με τον άλλο με συνετό, με λογικό τρόπο μπορούν πολλές προκαταλήψεις να αντιμετωπιστούν και να υπάρχει συμβιβαστική διάθεση, διάθεση σε συμβιβασμούς. Αυτό ήθελα να πω. Και για τη θέση του κυρίου Γκίγκολτ ότι στο scoreboard, στον πίνακα επιδόσεων πρέπει πολύ διαφορετικοί συντελεστές να συμμετάσχουν και να μην οδηγηθούμε στη συζήτηση με ακραίο άλλο ε, σημείο να μην ενταχθούν στη συζήτηση αυτά τα σημεία. Έχουμε λοιπόν εδώ πολυμορφία των επιχειρημάτων μπορώ να ευχηθώ να πετύχουμε στο εγχείρημα αυτό. Ευχαριστώ. Κύριος Καζά παρακαλώ. Ε, Δεν χρειάζεται να μακρηγορήσουμε για αυτό το σημείο. Συμφωνώ λοιπόν με τον κύριο Κρότσμαν και προφανώς και με τον κύριο Τόμας Μαν. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι παρόλα αυτά. Και αυτό είναι ότι αυτό το θέμα το συζητήσαμε με τους συναδέφους και όδης εισηγητές στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Αλλά ακόμα και εκεί είδα ότι υπήρχαν πολλές αντιστάσεις ε, στις προτάσεις του κυρίου Γκίγκορντ. Έπρεπε, θα, μπορούσαμε να, θα έπρεπε να μπορούμε να τα δεχθούμε, αλλά δεν υπάρχει συμφωνία. Υπάρχει αντίσταση, ακόμα και στα μέλη, ε, υπάρχει αντίσταση στα μέλη της Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής. Γιατί διαφορετικά θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε ότι είναι ένα θέμα που πρέπει στην οίκον να συζητηθεί και όχι στην Επιτροπή Απασχόλησης. Δεν είναι δική μας αρμοδιότητα να συζητάμε τέτοια θέματα, γιατί αυτό είναι ένα θέμα που καλύπτεται από τις αρμοδιότητες της Επιτροπής ΕΚΟΝ και όχι της Επιτροπής Απασχόλησης. Ο κύριος Λούτβιξεν και μετά θα συνοψίσουμε. Ευχαριστώ. Απλώς Ήθελα να σας πω ότι είναι πολύ σημαντικό για τους κοινωνικούς εταίρους στην αγορά εργασίας, δηλαδή ε, για εκείνους που είναι υπεύθυνοι για τις συλλογικές συμβάσεις, να φτάσουν σε λογικούς όρους συνένεσης. Εάν αποφασίσουμε στις Βρυξέλλες ότι θα παρέμβουμε στις διαδικασίες συλλογικών συμβάσεων εργασίας, θα έπρεπε να πω ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ κοινωνικών εταίρων οδηγούν σε μισθούς που επιτρέπουν ευελιξία έτσι ώστε να κρατήσουμε και την ανταγωνιστικότητά μας διότι οι μισθοί θα πρέπει να αυξηθούν, να μειωθούν ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς. Ε, εγώ ανησυχώ κάπως σε σχέση με το μισθολογικό αυτό πλαίσιο, διότι οποιοδήποτε θελήσει να άρει τις αρμοδιότητες των κοινωνικών εταίρων και εκείνοι οι οποίοι θέλουν να αποσύρουν αυτή την αρμοδιότητα από τους κοινωνικούς εταίρους ε, οδηγούνται σε, ένα επικίνδυνο, σε μια επικίνδυνη εξέλιξη. Οι κοινωνικοί εταίροι έχουν το δικαίωμα διαπραγμάτευσης. Έτσι η Ευρώπη μπορεί να αυξήσει και την ανταγωνιστικότητά της. Έχω υποβάλει ορισμένες τροπολογίες επί του θέματος. Είναι θέμα ύψης της σημασίας. Κύριε Λούτβικσον, νομίζω ότι ότι δεν υπάρχουν ε, δυσκολίες ως προς την υποστήριξη των ε, τροπολογιών καθεαυτών. Πριν φτάσουμε στα συμπεράσματά μας, στα τελικά μας συμπεράσματα, θα ήθελα να επισύρω την προσοχή του κυρίου Κάζα και του κυρίου Τόμας Μαν στο J, διότι στην τροπολογία συμβασμού J ορίζουμε το πνεύμα το οποίο διέπει το βαθμολόγιο και το πώς θα πρέπει να καταρτιστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν λέμε ότι οι χώρες που έχουν πλεόνασμα θα πρέπει να διορθώσουν τη θέση τους και να μην προβαίνουν σε εξαγωγές. Δεν λέμε κάτι τέτοιο. Λέμε ότι Εφόσον πρόκειται για εξωτερικές ανισότητες, θα πρέπει να προσέξουμε το υπερβολικό έλλειμμα καθώς και το πλεόνασμα. Όταν δούμε την κατάσταση Ευρωπαϊκής Ένωσης αντικειμενικά και ειλικρινά, θα πρέπει να δούμε τι συμβαίνει με τα πλεονάσματα ορισμένων ανταγωνιστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα θέμα κοινή λογική. Δεν είναι καθόλου ιδεολογικό το ζήτημα. Ελπίζω λοιπόν να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε. Ή πείτε μου, ποιο είναι το πρόβλημά σας με την πρόταση σύμβασμου J. Πού έγκυται η δυσκολία. Donc, Κύριε Κάζα, δεν έχω κανένα πρόβλημα με το σύμβασμο J υπό τον όρον ότι η λέξη shall αλλάξει σε may και νομίζω ότι ήδη έχει αλλάξει. Άρα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με το σύμβασμο J. Προτείνω τα υπόλοιπα προβλήματα να τα δούμε μέχρι αύριο με τους Κρόιτσμαν Γκίγκολτ. Αλλά και τώρα να συνοψίσουμε, να τελειώσουμε εδώ, διότι επειδή ε, έχουμε και μία τελευταία έκθεση για τα διορθωτικά μέτρα των μακροοικονομικών ανισορροπιών, αυτό το έχουμε ήδη θίξει, το θίξαμε ήδη όταν συμφωνήσαμε στον αποκλεισμό της λέξης including και ο κύριος Κρόιτσμαν συμφώνησε, άρα κάνουμε την ίδια διόρθωση. Ζητώ συγγνώμη από τους συναδέλφους για αυτή την σκληρή διαπραγμάτευση μεταξύ ημών και ημών, αλλά χρειαζόταν για να δώσουμε τελική μορφή στις ε, τροπολογίες. Τελειώνουμε λοιπόν με αυτή την ομάδα που θα ψηφίσουμε αύριο και φτάνουμε στο τελευταίο θέμα της ημερήσιας διάταξης και δίνω το λόγο στον Αλεχάνδρο Θέρκας για να εξετάσουμε τις τροπολογίες. Α, ο κύριος Κάζα. Πρόεδρε, αναλύσαμε ε, προβλήματα σε σχέση με πτυχές αυτού του χαρτοφυλακίου. Θέλω να σας ευχαριστήσω Πρόεδρε να ευχαριστήσω τον κύριο Κρόισμαν και τον κύριο Γκίγκολτ για τη συνεργασία, το πνεύμα συνεργασίας, για το χρόνο που αναλώσατε και μου δώσατε εμένα και πιστεύω ότι χωρίς αυτή τη συνεργασία δεν θα είχαμε καταλήξει σε αυτό το θετικό συμπέρασμα. Ευχαριστώ. Euh. Συμμερίζομαι τα λόγια σας κύριε Συν εισηγητά. Ο κύριος Θέρκας για να εξετάσουμε τις τροπολογίες ως προς την ενιαία άδεια παραμονής και εργασίας. Κύριε Θέρκας, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ακόμα και για λίγο χρόνο Χρειαζόμαστε όμως κάποια συζήτηση γιατί υπάρχουν κάποια θέματα που συνοδεύονται από κάποια επίμαχα θέματα και ίσως και για κάποια ε, θέματα που δημιουργούν κάποιες παρερμηνίες, γλωσσικά ίσως θέματα. Ε, ξεκινώ ευχαριστώντας σχιώδεις εισηγητές ε, όλους και την κυρία Τζιν Λάμπετ και άλλους που με βοήθησαν σε πολύ μεγάλο βαθμό για τους συμβιβασμούς ε, που καταλήξαμε. Επίσης και την κυρία Μέισεν και για τις γραπτές προτάσεις που υποβλήθηκαν και ευχαριστώ πολύ για αυτό αυτό το ε, ε, σχέδιο το οποίο έχω συντάξει το παρουσιάζω υπό τρία κριτήρια. Το πρώτο κριτήριο πρέπει να είναι μια, ένα συμβιβασμό χωρί καμιά αμφιβολία. Γιατί στο Ευρωκοινοβούλιο δεν προχωρήσαμε ποτέ παρά μόνο με συμβιβασμού. Ποτέ δεν μπόρεσε κανεί να επιβάλλει τίποτα σε, σε άλλου. Και αυτό είναι καλό. Έχουμε ένα συμβιβασμό λοιπόν μπροστά μα και θα προσπαθήσω να εκθέσω τα σχετικά. Γιατί καθώ είμαστε σε, κάποιο, ε, σε κάποια τριβή ή σύγκρουση όσον αφορά θέματα ερμηνεία με άλλε κοινοβουλευτικέ επιτροπέ, πρέπει να είμαστε ενωμένοι εμεί ω Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τα δικαιώματα στην εργασία και την κοινωνική προστασία. Μέσα σε αυτή τη συγκυρία θα πρέπει να πούμε καμιά κοινοβουλευτική επιτροπή δεν μπορεί να λύσει προβλήματα αν δεν έχει μια τέτοια ε, προσέγγιση. Αν μπορούμε όμως να τα επιλύσουμε, στη δική μας επιτροπή μπορούμε να τα επιλύσουμε. Και θα βοηθούσε αυτό, γιατί δεν έχει ακόμα ρυθμιστεί το θέμα αυτό, παρόλη την έκθεση της ε, ΑΦΚΟ θα βοηθούσε πολύ μια ομόφωνη θέση της δικής μας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής σε σχέση και με την ε, Επιτροπή ΛΥΜΠΕ που θα προσπαθούσε να προχωρήσει δικά τη θέματα θέματα χωρίς να είναι δική της αρμοδιότητας όμως. Το θέμα είναι ότι αυτή η ε, προσέγγιση είναι απόλυτα αναγκαία, συμβιβαστικά δηλαδή. Και αυτό γνωρίζει, γνωρίζοντας ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε το 100% αυτών που ζητούμε. Ξέρουμε όμως ότι κανένας δεν μπορεί να πετύχει ποτέ 100% τα αιτήματά του. Και αυτό είναι η ιδέα που εμπνέει ένα συμβιβασμό. Τώρα, ανέλησα τις 52 τροπολογίες, έγινε μεγάλη προσπάθεια. Μπορώ να πω ότι από τις 18 τροπολογίες που υποβλήθηκαν από το ΕΛΚ υπάρχουν 16 που είτε τις δεχόμαστε είτε αντανακλώνται σε συμβιβασμούς. Από την ε, Ενωμένη Αριστερά, Νοτική Αριστερά, από τις 6, τρεις εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία. Από τις 5 των Πρασίνων, δύο εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία. Και μία από, ε, από την, ε, η μία της Άλντε. Έγινε μεγάλη προσπάθεια λοιπόν. Θα θα προσπαθήσω να είμαι περιεκτικός για, αυτές, για αυτούς τους έξι συμβιβασμούς παρουσιάζοντας τα κυριότερα στοιχεία. Ο πρώτος συμβιβασμός είναι ο συμβιβασμός Α. Αναφέρεται σε όλα τα προβλήματα που αφορούν τους... Ε, ε, κατά εργαζόμενους. Εδώ υπήρχαν ακραίες θέσεις. έπρεπε να ερμηνεύσουμε, να δούμε ποιο είναι το εύρος ε, της οδηγίας που μπορεί να λύσει το θέμα των αποσπόμενων εργαζομένων. Ακολουθώντας τώρα μία γραμμή σε σχέση με την πρόταση των σοσιαλιστών που ήθελαν να την περιορίσουν σε μία αρχή και μεταξύ άλλων που ήθελαν να τα να διευρύνουν. Έτσι λοιπόν θα αφήσουμε τα πράγματα όπως ε, πρότεινε η Επιτροπή ε, αρχικά ξεχνώντας τις θέσεις μας ε, και επιτρέποντας αυτό το θέμα να ρυθμιστεί όταν θα προχωρήσει η συζήτηση σε σχέση με την αναθεώρηση της οδηγίας για αποσπόμενους εργαζόμενους αυτή η ε, προσέγγιση σε σχέση με την ε, ε, υιοθέτηση της ίσης αντιμετώπισης εδώ θα δούμε αυτό το θέμα ή σε άλλο πλαίσιο. Θα το θέσουμε στην τομεακή οδηγία. Εγώ θα προτιμούσα να είχαμε ένα, μια οδηγία πλαίσιο εδώ, αλλά αυτό είναι ανέφικτο. Ας αφήσουμε λοιπόν τη συζήτηση για την ισότητα της μεταχείρισης των posting εργαζόμενων όταν θα έρθει εκείνη η ώρα. Κατά τα άλλα, την οδηγία θα την ε, αφήσουμε λοιπόν ε, σε αυτό το πλαίσιο και έτσι δεν υπάρχουν νικητές και εκτιμένοι. Στο συμβιβασμό Β αναφέρεται σε μια άλλη πτυχή που εμείς οι σοσιαλιστές θα θέλαμε οι εργαζόμενοι που φτάνουν στην Ευρώπη να έχουν και αυτή πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες ε, και στην δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στην ε, κοινωνία σε ένα πλαίσιο απασχόλησης. Ε, όμως οι εθνικοί νόμοι όσον αφορά την προσφορά και την ελευθερία, την συμβατική θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Ο συμβιβασμός Β λαμβάνει υπόψη και τις δύο πρόπτικες. Δίνει την δυνατότητα να έχουν τα δικαιώματα αυτά αυτοί οι εργαζόμενοι. Γίνεται σεβαστό το αίτημα του ΕΛΚ όμως η πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίε όσον αφορά τα κράτη-μέλη να βρίσκεται υπό την αρχή της συμβατικής ελευθερίας. Δεν νομίζω να υπάρχει κανένα πρόβλημα, ούτε θα δημιουργηθούν προβλήματα. Ο συμβασμός Γ είναι ένα απλό σχετικά θέμα, αλλά που δυστυχώς ενέχονται εδώ δυσκολίες και παρερμηνίες. Αναφέρεται στο άρθρο 12, παράγραφο 2, άρθρο α, που είναι θέματα ίσης μεταχείρισης στην εκπαίδευση. Η Ενωτική Αριστερά θα ήθελε αυτό το άρθρο να επιτρέπει στα κράτη-μέλη να θεσπίζουν περιορισμούς όσον αφορά την ίση ε, μεταχείριση εκτός από την εκπαίδευση. Υπήρχε από άλλους η πρόθεση να αρθεί ο περιορισμός. Το ΕΛΚΑ ήθελε να αποσαφινιστούν κάποιες πτυχές. Εγώ νομίζω ότι το σημαντικό είναι να ε, ληφθεί υπόψη το εξή, ότι αυτή είναι μια οδηγία που δεν δίνει δικαιώματα, αλλά το δικαίωμα μόνο ίσης μεταχείρισης. Δεν λέμε ότι ένας ε, μετανάστης θα έχει δικαίωμα ε, εκπαίδευσης ή πανεπιστημίου ή όταν θα φτάσει μία ε, μέρα στην Ευρώπη. Λέμε όμως ότι πρέπει να έχει ίσα δικαιώματα όπως οι, ε, εθνικά, οι υπήκοοι του κράτους σε σχέση με συγκεκριμένα δικαιώματα. Εδώ να υπάρχει η δυνατότητα αυτή ίσης δικαιωματα οπως η εθνικα η ίσο πλαίσιο δικαιωμάτων. Εγώ σε 80% δέχτηκα την πρόταση του ΕΛΚΑ για την διευκρίνηση πρέπει να διευκρινιστούν αυτά όμως. Είπε το ΕΛΚΑ ίση μεταχείριση θα δίνεται για εκείνους ε, που εργάστηκαν ή για εκείνους που ε, έχουν τύχη ε, υποστήριξης. Περιορίζεται δηλαδή αυτό το δικαίωμα σε εκείνους που είναι εργαζόμενοι και όχι δεν δίνεται σε άλλους. Ακόμα έτσι κιόλας είναι ένα δικαίωμα το οποίο δίνεται στους εργαζόμενους που έρχονται με ενιαία άδεια στην Ευρώπη. Το ΕΛΚΑ θα ήθελε να αποκλείονται οι φοιτητέ από την οδηγία του 2004. Δεν χρειαζόταν να το πει κανεί αυτό, αλλά το ανέφερε ω επιθυμία του το ΕΛΚ. Εντάξει, να αποκλείονται λοιπόν οι φοιτητέ. Επαναλαμβάνω, είναι μια οδηγία που αφορά του εργαζόμενου που έρχονται στην Ευρώπη υπό την ενιαία άδεια. Και δεν αφορά εδώ του φοιτητέ ή οποιουσδήποτε άλλου, αλλά μόνο εκείνου που έχουν την άδεια και τι σύμβαση, που τους το συμβόλαιο που τους επιτρέπει να εργάζονται στην ε, Ευρώπη. Εδώ αυτή η ε, διαφοροποίηση επιθυμεί το ΕΛΚ να αναφέρεται ξεχωριστά, ότι πρόκειται μόνο για εργαζόμενους. Ήθελε να αποκλείονται οι υποτροφίες ε, το ΕΛΚ. Εγώ όμως πιστεύω ότι οι εργαζόμενοι που φτάνουν στην Ευρώπη με single permit, ε, αν μπορούν να πάρουν μια υποτροφία, γιατί να τους την αρνηθούμε. Όμως δεν επιθυμεί το ΕΛΚ. Λένε ότι υπάρχουν όροι, προϋποθέσεις κλπ. Εντάξει, το δεχτήκαμε. Όμως από την άλλη πλευρά πρέπει να δώσει κάτι στην ενωτική αριστερά και στους σοσιαλιστές ως ε, ε, αντιπρόταση το ΕΛΚ. Εμείς επιθυμούμε εκείνα τα οποία είναι επαγγελματική κατάρτιση και εκείνα τα οποία αφορούν την πρόσβαση σε ε, φίτηση για εκείνους τους εργαζόμενους που βρίσκονται με single permit στην Ευρώπη, αν δίνεται η δυνατότητα να βελτιωθεί η ικανότητά του η επαγγελματική, να υπάρχει ισότητα μεταχείρισης για την κατάρτισή του, για όσους εργάζονται, για όσα θέματα συναρτώνται άμεσα με την εργασία του. Τι λιγότερο θα μπορούσαμε να δίναμε σε αυτούς ε, σε σχέση όταν κάνουμε λόγο για μια βιομηχανία στην ε, Γερμανία, στη Γαλλία, στο Βέλγιο αλλού και υπάρχει δυνατότητα μέσω κάποιων μαθημάτων να βελτιωθεί η επαγγελματική κατάτηση. Ε, δεν θέλουμε τίποτα να δίνεται δωρεάν, ούτε θέλουμε να αφαιρέται τίποτα, αλλά μόνο όταν αφορά ένα θέμα την βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης, τότε μόνο να επιτρέπεται. Καταλήξαμε στο Καταλήγουμε στον συμβιβασμό ΔΕΛΤΑ. Τον διαρέσαμε σε δύο τμήματα. Δύο λεπτά, Πρόεδρε, και να... θα καταφέρω να τα ολοκληρώσω. Είναι θέματα που απαιτούν ολόκληρη ώρα συζήτηση και όχι λίγα λεπτά στο θέμα αυτό θίγουμε το καυτό, δικαίωμα, το καυτό θέμα. Ποια δικαιώματα έχουν εκείνοι οι εργαζόμενοι που ήρθαν εδώ όχι για να εργαστούν μια μέρα ή συγκυριακά, αλλά θέλουν να μείνουν να εργαστούν εδώ με άδεια εργασία για δύο, τέσσερα και τα λοιπά χρόνια. Να ζήσουν και να εγκατασταθούν στην Ευρώπη με την ενιαία άδεια, ε, single permit. Ποια δικαιώματα θα έχουν. Εδώ υπάρχουν προβλήματα. Πρέπει να υπάρχει κάποια κοινωνική ασφάλιση που θα συνδέεται και σε σχέση με τα θέματα τη ε, διαμονή του και όχι μόνο της εργασίας. Θα αφήσουμε εκτός, θα αφήσουμε στα, ε, στην αρμοδιότητα των κρατών μελών να θέσουν όρους και προϋποθέσεις, να άρουν τις αυτόματες ε, εκείνες προϋποθέσεις της ισότητας μεταχείρισης. Η προστασία όμως ε, της οικογένειας και η ανεργία είναι σημαντικά θέματα. Δεν, δεν θέλουμε όμως να αφήσουμε εκτός πλαισίου την υγειονομική περίθαλψη και την ιατροφαρμακευτική κάλυψη. Ποια σώματα μπορούν να έχουν τέτοιες, ε, αυτού του είδους την προστασία και σε σχέση με τις συμβάσεις ε, μικρότερης διάρκειας από έξι μήνες ε, θα επιτρέψουμε στα κράτη-μέλη να περιορίζουν το δικαίωμα σε σχέση με δικαιώματα ανεργίας και σε σχέση με τα δικαιώματα ε, προστασίας της οικογένειας. Θα αφήσουμε και εκτός ε, τους φοιτητές. Εντάξει, δεν χρειαζόταν να το πούμε αυτό για τους φοιτητές, αλλά θα το εξετάσουμε ξεχωριστά μετά από το αίτημα το, του ΕΛΚ. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν έχει νόημα να αποκλειστούν άλλοι. Και τώρα με ποιο δικαίωμα θα τους αποκλείσουμε. Δεν είχε ε, κανένα νόημα να αφαιρέσουμε αυτό το δικαίωμα σε που έχουν έχουν μακροπρόθεσμη άδεια να εργαστούν στην Ευρώπη. Με αυτές τις παρατηρήσεις νομίζω οι συμβαστικές ε, τροπολογίες και η τελευταία αυτή η συμβαστική πρόταση που είναι ο συμβασμός, η συμβαστική πρόταση ε αναφέρεται απλά στην ε, δυνατότητα να εισπράττονται οι συντάξεις ε, εκτός στο εξωτερικό πάλι υπό την ίση μεταχείριση όπως προαναφέραμε. Ολοκληρώνω Πρόεδρε. Νομίζω βρισκόμαστε σε μια πολύ θετική κατάσταση και με... για την ομάδα μου με μεγάλη θυσία, διότι σε σχέση με το εύρος τη οδηγίας και τα λοιπά, τις αρχικές μας απόψεις τις αλλάξαμε. Δεχθήκαμε πολλές τροπολογίες ε, του ΕΛΚ για να γνωρίζετε ότι δεν θέλουμε να διευρύνουμε απεριόριστα, αλλά θέλουμε να καθορίσουμε ένα ενιαίο πλαίσιο δικαιωμάτων. Όχι όμως για μια μέρα, αλλά για χρόνια, για εκείνους που έρχονται εδώ, να υπάρχει δυνατότητα να ενταχθούν, να αποφύγουμε με την ξενοφοβία και τον ρατσισμό όσον αφορά εργαζόμενους από τρίτες χώρες, αλλά που δεν θα έχουν λιγότερα δικαιώματα. Να έχουμε νόμιμους εργαζόμενους που θα εργάζονται στην Ευρώπη με τους δικούς μας εργαζόμενους. Γι' αυτό υποσχεθήκαμε την ισότητα μεταχείρισης. Θέλω να ζητήσω από τους συναδέλφους να υπερψηφίσουν αυτό το συμβιβασμό που είναι θυσία για όλους, αλλά που επιτρέπει ο συμβιβασμό σε όλους να αποκαταστήσουμε την ισορροπία μεταξύ των διαφορετικών θέσεων και να πάμε στην Ολομέλεια ε, την επόμενη εβδομάδα. Υπέρ τη ανθρώπινη αξιοπρέπειας, της αξιοπρέπειας των εργαζομένων με την δέσμευση να ενταχθούν στην κοινωνία μα. Όχι να πούμε να ενταχθούν και να του αρνηθούμε τα μέσα να ενταχθούν. Σα ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σαρή μου ζήτησε το λόγο πριν από Όμεν Ράιτεν. Ευχαριστώ, ε, Πρόεδρε. Νομίζω ότι αυτά τα σημεία, αυτά τα θέματα στην ημερήσια διάταξη είναι ιδιαίτερα περίπλοκα και είναι πολύ κρίμα που δεν έχουμε ε, αρκετό χρόνο. Συμφωνώ με τα σχόλια του κυρίου Θέρκας ήταν πολύ δύσκολο το θέμα και θα πρέπει να έχουμε την ευρύτερη δυνατή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Ενώ ήμασταν πιο περιοριστικοί στην ερμηνεία μας, στις χώρες μας έχουμε πολιτικά κόμματα τα οποία ε, βρίσκονται στο δεξί φάσμα και στο δεξί πολιτικό φάσμα και στη Φιλανδία και στη χώρα μου θα πούνε ότι βασιζόμαστε στην άδεια παραμονής και δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε σε πολλούς αλλοδαπούς να ε, μπουν στις χώρες μας διότι το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης θα καταρρεύσει. Η άλλη πλευρά του νομίσματος όμως, πρόεδρε, είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε μία κατάσταση όπου οι εργαζόμενοι κάνουν χρήση των ε, τρίτων χωρών και έχουν ε, χαμηλότερα επίπεδα κοινωνικής ασφάλισης για να ανταγωνιστούν εργαζόμενους των δικών μας κρατών μελών. Άρα θα πρέπει να επιζητήσουμε μία ισορροπία εδώ και να είμαστε συνεπείς θα πρέπει να παραδεχτώ ότι στις τροπολογίες που υπέγραψα εγώ, καταρχήν, ανέκυψαν προβλήματα αργότερα που δεν είχαν ε, προκύψει αρχικά. Ως προς τους ε, συνδυασμούς Δέλτα 1 και Δέλτα 2, επειδή το θέμα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο, ίσως ε, οι τροπολογίες συμβιβασμού να σημαίνουν ότι ένα πρόσωπο που έχει άδεια εργασίας και βρίσκεται σε μια χώρα λιγότερο από έξι μήνες, για λιγότερο χρονικό διάστημα από έξι μήνες, το πρόσωπο αυτό δεν μπορεί να λάβει επιδόματα, οικογενειακά επιδόματα ή επίδομα ανεργίας. Θα πρέπει όμως να θυμόσαστε και εδώ διαφέρει θέσιμο θέση από το Συμβούλιο, θα πρέπει να θυμηθείτε ότι αυτό το πρόσωπο, αν πέσει από τις καλοσχές ενός κτηρίου, τότε και εκείνος και η οικογένειά του θα πρέπει να τύχουν υποστήριξης. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει ε, σύνταξη αναπηρίας, να χορηγηθεί σύνταξη αναπηρίας. Εάν μιλάμε για κοινωνική πολιτική στην χριστιανοδημοκρατία θα πρέπει να θυμόμαστε τι είναι σωστό και τι είναι δίκαιο. Εγώ το συζήτησα αυτό στη δική μου πολιτική ομάδα. Αυτό που κάνουμε εδώ είναι το εξής. Προσπαθούμε να εγγυηθούμε το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης, όπως αναφέρεται στον κανονισμό 803. Και αυτό αναγνωρίζουμε, την ίση μεταχείριση. Παράλληλα όμως λέμε ότι υπάρχει ίση μεταχείριση μόνο για αυτόν που λαμβάνει την άδεια εργασίας. Hm. Δηλαδή, ε, εάν έχει ασφάλιση κοινωνικής ε, απασχόλησης και αυτό αφορά τον κανονισμό 803 πολλές φορές όταν κάποιος έρθει στη Γαλλία, Ολλανδία και Φιλανδία με, ε, ένα, με μια άδεια εργασίας, μπορεί να αποφασίσει να σπουδάσει, να την εργαστεί. Τότε υπόκειται σε ορισμένα κριτήρια, όπως γλωσσικά και άλλα. Και νομίζω ότι αυτό το πρόσωπο, αυτός ο πολίτης θα πρέπει να έχει πρόσβαση εργασίας. Δηλαδή, αν προσλάβουμε έναν ειδικό στους υπολογιστές από την Ινδία, θα πρέπει να μπορεί να έχει πρόσβαση σε ένα πρόγραμμα κατάρτισης, όπως θα έχει και ο αντίστοιχος Γάλλος, Ολλανδός και ούτω καθεξής, διότι κρατά το ίδιο επίπεδο δεξιοτήτων που μπορούν να έχουν και οι κάτοικοι της συμμεταπής. Αυτό είναι το θέμα ίσης μεταχείρισης. Βεβαίως υπάρχουν και ορισμένοι περιορισμοί που είναι δίκαιοι και εδώ μιλώ για τα επιδόματα παιδιού, επιδόματα ε, ανηλίκου. Ένα τελικό σχόλιο. Τι έχει κάνει το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο λέει ότι κάποιος που έχει ε, θεώρηση έχει λιγότερα δικαιώματα. Δεν έχει δικαίωμα κοινωνικής ασφάλισης ούτε ίσης μεταχείρισης σε σχέση με ε, εκείνο που έχει ενιαίο, ενιαία άδεια. Αυτό που μας οδηγεί όμως. Μας οδηγεί στο εξής. Αν μιλάτε για έναν εργαζόμενο θα φτάσετε σε δύο διαφορετικές κατηγορίες εργαζομένων από τρίτες χώρες και πάντα θα επιλέξουμε το πιο φτηνό, εκεί που δεν υπάρχουν υποχρεώσεις. Και αυτό που είναι το χειρότερο είναι το εξής. Η ενιαία άδεια έχει στόχο να υπάρχει δυνατότητα άδειας παραμονής και εργασίας ε, από κοινού, δηλαδή να είναι μια συνδυασμένη άδεια. Και στόχος είναι να έχουμε μια άδεια παραμονής που να επιτρέψει κάποιον και να εργαστεί. Να έχουμε δηλαδή ένα απλό σύστημα χορήγησης άδειας παραμονής και εργασίας. Και τώρα φαίνεται ότι περιπλέκεται το ζήτημα θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Τρεις ζητούν το λόγο. Νομίζω ότι μπορούν να παραμείνουν ε, οι διερμηνείς ε, πέντε λεπτά ακόμα, ακόμα και μετά θα συνεχίσουμε αγγλικά. Ευχαριστώ. Καταρχήν κάτι τυπικό και επίσημο για τη διαδικασία, διότι πολλά σε αυτό το χαρτοφυλάκιο δεν τα βρήκα καλά έτσι όπως εξελίχθηκαν. Το ένα είναι ότι γενικά, μια και τώρα, λόγω της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής ε, ΛΥΜΠΕ που απορρίφθηκε η πρόταση στο Κοινοβούλιο, ξανασχολούμαστε εμείς με αυτό το θέμα ο τρόπος με τον οποίο όμως έγινε αυτό πρόεδρε δεν είναι σωστός διότι γίνεται λόγος ότι ε, α, τοποθετούνται εξ ονόματος της ε, Κοινοβουλευτικής Επιτροπής όμως εγώ ως κοιόδηση συγγήτρια και οι συντονιστές ε, δεν ε, είχαμε ενημερωθεί. Πρέπει πάντα να γίνεται αυτό για να είμαστε δίκαιοι ο ένας απέναντι στον άλλον. Να γίνονται όλα σωστά από πλευράς διαδικασίας για να εργαζόμαστε δημοκρατικά όπως πρέπει. Αυτό με ενόχλησε δεν έγινε και με ενόχλησε το δεύτερο το οποίο δυσκολεύει τη δουλειά μας και σήμερα είναι το ότι την τελευταία διατύπωση των συμβιβασμών την πήρα ως ε, έγγραφο μόλις μπήκα στην αίθουσα. Δεν γίνεται αυτό και ως διαδικασία πρέπει να το έχουμε στη διάθεσή μας πιο πριν. Είχα μια τελική διατύπωση που ήταν από χθε το, μεσημέρι, αλλά σήμερα το απόγευμα δεν είχα τίποτα που να είναι πιο επικαιροποιημένο πρέπει να εργαζόμαστε καλύτερα γιατί από αυτό εξαρτάται. Είναι δύσκολο θέμα το θέμα της ενιαίας άδεια, single permit. Είναι σαφές αυτό. Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε σε κανένα τίποτα. Πρέπει να ξέρουμε τι ακριβώς εμπεριέχεται, με ποια διατύπωση, σε, κάποια, σε ποια τροπολογία. Και όταν εδώ αλλάζουν κάποια πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρώτον να παρακολουθήσουμε και δεύτερον να ξέρουμε αν το δεχόμαστε ή όχι. Και σε σχέση με τη σημερινή εξέλιξη, μέχρι πριν από την ψηφοφορία στην Ολομέλεια όλα πήγαιναν καλά, αλλά και μπορώ να επενέσω τον κύριο Θέρκας γι' αυτό, αλλά ε, σε σχέση με κάποιες ε, τροπολογίες ε, που είχαν κατατεθεί και που τώρα στρέφον, ήταν κατά της δικής του άποψης ε, βρίσκω ότι δεν ήταν σωστή η αντιμετώπιση θα έπρεπε να ήταν δυνατόν ως σκιώδης εισηγήτρια να είχα και εγώ συμμετάσχει σε αυτές τις διαβουλεύσεις ε, αυτό σε σχέση με τη διαδικασία τα διαδικαστικά δεύτερον όσον αφορά τα θέματα ουσίας συμβαίνει το εξής ακριβώς δύο παρατηρήσεις δύο τροπολογίες κατέθεσα που αφορούν το άρθρο 3 στο 3β πρόκειται για την οδηγία για την απόσπαση εργαζόμενων το κείμενο το οποίο εγκρίνεται, τίθεται υπό έγκριση τώρα ενώ είχα κάτι άλλο στη διάθεσή μου έχουμε εδώ μια τροπολογία που αφορούσε πριν από την τελική ε, ψηφοφορία την απόρριψη που ε, επίθε μετά και τώρα να λέμε θα αποσπώνται μόνο κατά τη διάρκεια της απόσπασης. Και εδώ όχι σε σχέση με την οδηγία. Είναι δύσκολο αυτό να το ε, παρακολουθήσει κανείς. Είχε δοθεί διασφάλιση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι όταν θα παίρνουμε την οδηγία 96-71 ότι αυτό τι θα σήμαινε. Θα μπορούσαν ε, οι πίκοοι τρίτων χωρών που αποσπώνται από τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν καλύτερη θέση από εκείνους που αποσπώνται και αποστέλλονται από χώρες Τη ε, της Ευρώπης. Και αυτό πάλι δεν μπορεί να γίνει δεκτό. Και δεύτερον, και δεν είμαι η μόνη που αυτή την ε, τροπολογία την είχε καταθέσει μία φορά ε, στο παρελθόν, διότι αυτό είναι σημαντικό θέμα. Με βάση αυτό εξαρτάται η έκβαση της πρώτης ανάγνωσης. Εδώ και 12 χρόνια εργαζόμαστε για αυτό το συμβιβασμό. Και φυσικά το λέει και ο κύριος Θέρκας, ένα συμβιβασμός είναι συμβιβασμός για όλους. Δεν μπορεί να είναι ιδανικός για κανέναν, αλλά πρέπει να τον ολοκληρώσουμε και να μπορέσουμε να να δημιουργήσουμε θεμέλια να οικοδομήσουμε με αυτόν. Αν διατηρήσουμε τώρα το συμβιβασμό Α ως έχει, τότε δεν θα υπάρχει πρώτη ανάγνωση και δεν θα έχουμε τίποτα πάλι στα χέρια μα. Και δεν θέλω να γίνει κάτι τέτοιο. Πρέπει να έχουμε κάτι στο οποίο να μπορούμε να οικοδομήσουμε. Το δεύτερο που κατέθεσα είναι η τροπολογία 47, ταυτόσημη με τη 46. Πρόκειται για το άρθρο 12, παράγραφο ε. Πρόκειται πάλι εδώ ακριβώς γι' αυτό ποια δικαιώματα, κοινωνικά δικαιώματα μπορεί να έχει κάποιο ως εργαζόμενος, ο οποίο έχει άδεια εργασίες αλλά δεν έχει εργαστεί ούτε μια μέρα. Έχει τα ίδια δικαιώματα με κάποιον υπήκο που έχει ήδη εργαστεί και έχει ήδη πείρα ω εργαζόμενο. νέου. Ναι, βλέπω ε, αυτή τη στιγμή κατανέβεται, αλλά θέλω να ξέρω τι είναι εφικτό. Τι μπορούν οι άνθρωποι που έρχονται στην Ευρώπη να έχουν ω δυνατότητα σε σχέση με την εργασία τους και την προστασία τους. Δεν, μπορούν όλα να τα κατα... δεν μπορούμε όλα να τα καταφέρουμε. Δεν είμαστε παράδεισος. Πρέπει να δούμε τι είναι εφικτό και τι μπορεί να γίνει. Και να δούμε, να κάνουμε το πρώτο βήμα σε σχέση με την οδηγία. Γι' αυτό θέλω να πω ότι αυτά τα οποία αναφέρονται στο ένα και στο άλλο είναι με ακριβώς την διατύπωση αυτή, αλλά κάτι λείπει ακριβώς. Γιατί αν λείπει κάτι υπάρχει διαφορετικό νόημα στο τέλος. Και δυστυχώς με αυτή τη μορφή και με αυτόν τον τρόπο δεν μπορώ να τα δεχτώ εγώ, παρότι θα ήθελα να έχουμε μια κοινή έκβαση με έγκριση όλων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δεν θέλω να σπαταλήσω το χρόνο σας. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ, πρέπει να πω, όταν έχουμε αποσπόμενους εργαζόμενους και όταν θα έχουμε την συζήτηση της οδηγίας αυτής θα έχουμε χρόνο το δεύτερο εξάμεινο του 2011 να τα συζητήσουμε. Ας μην αναλώσουμε το χρόνο μας με αυτό τώρα. Το πρόβλημά μου όμως και δεν ξέρω αν είναι γλωσσικό πρόβλημα ή πρόβλημα ουσίας κάνω λόγο για το συμβιβασμό C, τον συμβιβασμό Γ και την πρόσβαση σε κατάρτιση και εκπαίδευση και όρους και προϋποθέσεις για την πρόσβαση στην εκπαίδευση και κατάρτιση. Equal treatment, η συμμεταχείριση αναφέρεται στο αρχικό κείμενο. Αν κάποιος έχει μια τέτοια ενιαία άδεια, έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση και στην εκπαίδευση και κατάρτιση. Και μετά εισάγονται κάποιοι περιορισμοί, όροι και προϋποθέσεις. Όμως, αρκετές χώρες ε, έχουμε και οργανισμούς ε, στους οποίους ε, καταλήξαμε να μας συμβουλέψουν για αυτά τα θέματα δεν επιθυμούν, δεν τους αρέσει να περιοριστεί η πρόσβαση στους εργαζόμενους που έχουν εργασία ή που είχαν εργασία κατά το παρελθόν, που έχουν, εργάζονται τώρα ή είχαν εργασία κατά το παρελθόν. Διότι αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει όρο και προϋπόθεση περιοριστικό, λένε αυτοί οι οργανισμοί και οι ΜΚΟ. Κάποιοι οι οποίοι προσκαλούνται, ακόμα και ένας μεγάλος αριθμός ατόμων που προσκαλούνται από μια εταιρεία να εργαστούν σε αυτήν. Όταν η εταιρεία πτωχεύσει, όταν πέσει έξω, τότε έχουν το ίδιο δικαίωμα αυτοί οι εργαζόμενοι να έχουν πρόσβαση σε εκπαίδευση ή κατάρτιση όπως οι πολίτες αυτής της χώρας και δεν χρειάζεται και να πληρώσουν ίσως κιόλα. Πώς είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο, είναι δύσκολο να επεξηγήσει κανείς κάτι τέτοιο και δεν πρέπει να είμαστε αμφίσιμοι σε τέτοια θέματα. Αν παραμείνει αυτό έτσι, τότε δεν θα υπάρξει πρώτη ανάγνωση, δεν θα υπάρξει συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Ας είμαστε λοιπόν πιο λογικοί, ας επικρατήσει ο κοινός νους για να προχωρήσουμε. Euh, θα μιλήσω φιλανδικά. Σας ευχαριστώ για την Επιτροπή για το γεγονός ότι άλλαξε το κείμενο σε σχέση με την πρώτη ανάγνωση και για το ότι δυσχεραίνεται η εξέταση όπως είπαν κάποιοι. Όμως είχαμε προτάσεις για την πρώτη ανάγνωση και ε, αν μπορούσαμε να τα αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα δεν θα καταλήγαμε σε αυτή την κατάσταση τώρα. Αυτή η ενιαία αντιμετώπιση αντιφάσκει με την αρχή ότι κάθε κράτος μέλος έχει δικαίωμα να διασφαλίζει τα θέματα της ασφάλισης όπως επιθυμεί και για τις σκανδιναβικές χώρες. Αυτό ακριβώς επειδή έχουμε ευρύτατη, ας το πω έτσι, βάση για το σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων που διασφαλίζει ευρύτατη πρόσβαση ε, και δικαιώματα σε όσους ε, εργάζονται. Το σύστημα των σκανδιναβικών κρατών δίνει το υψηλότερο επίπεδο προστασίας ε, πανευρωπαϊκά από ό,τι γνωρίζω. Κατανοώ βέβαια τώρα την δυσκολία που έχουν οι εκπρόσωποι πολλών άλλων χωρών σε σχέση με αυτά τα θέματα δυσκολίες που θα ε, δημιουργούσε μια υιοθέτηση του προτύπου των σκανδιναβικών χωρών, διότι αυτό διευρύνει τις δυνατότητες πρόσβασης σε τέτοια δικαιώματα και για την οικογένεια και για ε, απεριόριστη πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, οδοντιατρική ε, σε πρόσβαση σε οδοντιατρικές ε, ε, υπηρεσίες ε, και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Κατανοώ λοιπόν για την, τα προβλήματα που υπάρχουν με τους συμβιβασμούς αυτή τη στιγμή, διότι αν δεν είναι δυνατόν να αλλάξει η διατύπωση θα πρέπει να αποσύρω εγώ την πρόταση αυτή και δεν θα την υπερψηφίσω. Για εκείνους που πιστεύουν ότι αν κάποιο πέσει από ένα ικρίωμα, για παράδειγμα, ως εργαζόμενος σε μια σκανδιναβική χώρα, δεν θα υπάρχει κάλυψη ασφαλιστική για τέτοιου, τέτοιου, τέτοιου είδους εργαζόμενους. Κανένας στις σκανδιναβικές χώρες δεν μπορεί να ανέβει σε ένα ικρίωμα αν δεν έχει ε, επαρκή ασφαλιστική κάλυψη. Λοιπόν, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο λοιπόν να επεκταθεί κάτι τέτοιο από ό,τι κατανοώ. Ευχαριστώ. Τελειώσαμε. Ευχαριστή πρόεδρος του διερμηνεί.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 But, but, but all, all the directive, all the directive is only for the worker and the, the single permit. All the directive. No, the, we speak about the attendez, student alors, Attendez, parce que comme il est quand même euh, 7h moins le quart... Euh, my, my final word. My final non, word. attendez. Attendez. Je vais